έκλεισε.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 Buenos días, les ruego que vayan tomando asiento porque ya hemos dado seis minutos de plazo a todo el mundo para que llegue. Y... Καλημέρα. Ήδη καθυστερήσαμε πέντε λεπτάκια για να δώσουμε σε όσους καθυστέρησαν το χρόνο να καθίσουν. Το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι το 10. Πρόκειται για την πράσινη βίβλο για τη μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Η συγγήτρια είναι η κυρία Πατράων Νέβες. Στην προηγούμενη με συνεδρίαση είχε κάνει μια πρώτη παρουσίαση ήδη και θα ήθελα να την ευχαριστήσω. Γιατί ήταν πολύ καλή η δουλειά της και γρήγορη ώστε να μπορέσουμε να εξετάσουμε στην Ολομέλεια του Φεβρουαρίου το θέμα της. Εχθές στις συντονιστές πήραμε μια απόφαση να γίνει μια ακρόαση την 1η Δεκεμβρίου λάβαμε μία απόφαση να γίνει μία κρόαση την 1η Δεκεμβρίου για το θέμα αυτό ειδικότερα της Πράσινης Βίβλου. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Πατράο Νέβες. Σας ευχαριστώ πολύ και καλημέρα σας. Και εγώ θα ήθελα να πω σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του συναδέλφου από όλα τα κράτη-μέλη σε αυτή την Επιτροπή Αλίας που χαιρετίζω στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων στο παρελθόν. Ξεκίνησα την παρέμβασή μου με μια αξιολόγηση γενικότατη της ε, πραγματικότητας όπως έχει σήμερα στην Αλία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να καταδείξουμε την ανάγκη να υπάρξουν εντοπίσεις, ε, ταυτοποίησης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Όχι μόνο ε, τομεακά ή κλαδικά, υπο, περισσότερο υπό το εγκάρσιο ολικό ε, συγκροτημένο πλέγμα για όλους τους εμπλεκόμενους που είτε έμεσα είτε άμεσα αφορώνται από αυτό το τομέα. Καθώς επίσης και την, το σύνθετο χαρακτήρα των δράσεων και συνέχισα με μια ευρεία ταυτοποίηση, όχι εξαντλητική βέβαια, των κυριότερων προβλημάτων που αφορούν τη σταθερότητα και την ανάπτυξη της αλληλευτικής δραστηριότητας σήμερα και που σε μεγάλο βαθμό αναφέρονται στην πράσινη βίβλο για τη μεταρρύθμιση της κοινή πολιτικής αλλίας. Αυτά λοιπόν τα προβλήματα είναι πολύ γνωστά και συνενετικά τα αντιμετωπίζουμε και πέρα από το θέμα της υπεραλίευσης όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των πόρων και πέρα από το πλεονάζον δυναμικό του στόλου της κοινότητας και την απώλεια, στο πω έτσι, διασπάθηση πόρων και άλλοι συντελεστές αξίζουν να ληφθούν υπόψη η κρίση οικονομική και χρηματοοικονομική παγκόσμια, οι αλλαγές οι που οξύνονται η πραγματικότητα των αυξημένων τιμών καυσίμων, το χαμηλό εισόδημα όσον αφορά τα αλλιεύματα για τους αλείς, η δυσκολία για να βρεθούν επενδύσεις όσον αφορά την ευρωπαϊκή αγορά, η απουσία πολιτικών κινήτρων που θα είναι καλά διατυπωμένα και θα είναι σε θέση να συντελέσουν την αναγκαία μεταβολή στον τομέα της αλλία η, ε, θα έλεγα, βραχυπρόθεσμη κυριότερα αντιμετώπιση η ε, παρουσία των εκπροσώπων των αλλιέων, η απουσία στρατηγικής ε, για μια στρατηγική ε, με, και πολλοί άλλοι λόγοι. Και καθόρισα τις ε, μεγάλες αυτές ε, θα έλεγα παραμέτρους όσον αφορά τα προβλήματα της, του τομέα και θα έλεγα τρεις άξονες εδώ υπάρχουν πρώτον προστασία και διατήρηση των αποθεμάτων, των αλευτικών απο, αποθεμάτων, δεύτερον αξιοπρεπής, αξιοπρεπές εισόδημα για τους αλληλείς και οι προοπτικές αηφορίας για τον τομέα. Χωρίς αυτά τα τρία στοιχεία η αηφόρος ανάπτυξη στην αλληλεία δεν θα είναι εφικτή. Και πάλι σε σχέση με αυτή την πτυχή θεώρησα ότι θα ήταν εύκολο, είναι εύκολο να επιτευχθεί συνένεση. Υπάρχει συνένεση. Τώρα, για την μεταρρύθμιση, εδώ τοποθετείται στο επίπεδο των διαβουλεύσεων για την λήψη αναγκαίων μέτρων για τον τομέα αυτόν. Διότι σε αυτόν τον τομέα υπάρχουν διαφορετικές προοπτικές και απόψεις που συγκρούονται για να υπάρξει μια αξιολόγηση το δυνατόν ευρύτερη και συνενετική για τόσο επίμαχα θέματα, προσπάθησα τις τελευταίες εβδομάδες να συνέρθω με όλους τους εμπλεκόμενους από τους πιο διαφορετικούς τομείς στον τομέα της Αλίας, κυρίως τους αρμόδιους της Γενικής Διεύθυνσης ΜΑΡ, ΤΕΖΕΜΑΡ, που θα συμμετάσχουν σε ε, που σε σχέση με τη συμμετοχή ε, σε workshops στις Αζόρες και στο Πόρτο και τη συμμετοχή τους εκεί έχουμε και μια συνάντηση με τον κύριο Επίτροπο Μπόργκ για μια ανταλλαγή απόψεων για την Πράσινη Βίβλο και συναφή θέματα. Προσπάθησα εξίσου κατά τη διάρκεια αυτών των τελευταίων εβδομάδων να ε, λάβουμε υπόψη σε ευρύτερο πλαίσιο τις ε, θέσεις που έχουν παρουσιάσει οι εκπρόσωποι των ε, συλλόγων και ενώσεων και τις θέσεις τους για τα πιο σημαντικά θέματα για τη μελλοντική μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Αναφέρομαι για παράδειγμα στα γνωμοδοτικά συμβούλια, τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια Επίσης ε, συμμετείχα, υπήρξε συμμετοχή σε διάφορες ε, παραμέτρους για την πράσινη βίβλο. Πράγμα το οποίο επέτρεψε να εκτεθεί όχι μόνο η αξιολόγησή μου για αυτό το θέμα, για αυτό το έγγραφο, αλλά να ακούσουμε κυρίως τις ε, αντιδράσεις και τις απόψεις που προκάλεσε η πράσινη βίβλος από τον τομέα σίγουρα μια περίοδος ε, μεγαλύτερη θα ήταν κάτι το οποίο θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα λαμβάνοντα υπόψη τη μεγάλη σημασία και για το παρόν και για το μέλλον του θέματος και το εύρος ε, της εργασίας που έχει επιτευχθεί. Δυστυχώς όμως το χρονοδιάγραμμα δεν επέτρεπε μεγαλύτερη προθεσμία. Και όσο, όσο αφορά αυτό και με τους περιορισμούς ε, και σε σχέση με όλες τις, ε, ε, τις παραμέτρους αυτές θα σας παραδοθεί η έκθεση. Δεν είναι τόσο ευρία και σφαιρική όπως θα επιθυμούσα αρχικά. Όμως εδώ έχουμε και δυνατότητα με τροπολογίες που υστερότερα θα κατατεθούν για την έκθεση σε ευρύτερο, στο πλαίσιο. Αυτή η έκθεση έχει εκπονηθεί όσον αφορά τα θεματικά πλέγματα, τα σημαντικότερα που έχουμε και τον τίτλο όπως αναφέρεται για μια σκόπιμη παρέμβαση, αποτελεσματική παρέμβαση και αντίδραση όλων των εμπλεκόμενων. Κάποιες πτυχές θα ήθελα να τονίσω, όπως η προάσπιση μιας καλύτερης επένδυσης στην έρευνα και στην ανάπτυξη, την επιστημονική όσον αφορά την αλία και καλύτερη ένταξη στον τομέα της αλίας των θεματικών πλεγμάτων του προγράμματος πλαισίου υποστήριξης στην ανάπτυξη, όπου η αλία είχε πραγματικά επουσιώδη ρόλο σε αυτό το πλαίσιο. Επίσης την υδατοκαλλιέργεια που πρέπει να είναι ισχυρή και αναζωογονημένη και που αποτελεί καταλήτη για την ανάπτυξη σε τομείς ε, συναφής ε, και που συνεισφέρει για την ανάπτυξη των παράκτιων ε, περιοχών με σαφή ωφέλη για τους καταναλωτές με τη μορφή τροφικών προϊόντων υψηλής ποιότητας που είναι υγιεινά προϊόντα, υγιή προϊόντα και που παράγονται με οικολογικό-βιολογικό τρόπο επίσης υπέρ της αύξησης μιας υδατοκαλλιέργειας που θα υλοποιεί όρους και προϋποθέσεις και στόχους και τα κράτη-μέλη θα διασφαλίζουν τις ευθύνες τους όσον αφορά τον έλεγχο και τον συντονισμό μεταξύ τους και θα μπορούν να υποφελούνται από διαθωτικά ταμεία και άλλες υποστηρικτικές δράσεις. Είμαι υπέρ της ενίσχυσης ε, της κοινοτικής παρουσίας ε, στις ε, περιφερειακές οργανώσεις και στις ε, διεθνείς ε, οργανώσεις και οργανισμούς και φόρα, ώστε να υπάρξει σωστή και καλή διαχείριση της αλίας και της αλλιευτικής προσπάθειας διεθνώς και καταπολέμηση της παράνομης αλίας. Είμαι υπέρ επίσης του, της θέσπισης μηχανισμών προστασίας για τα κοινοτικά προϊόντα της αλίας εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διοργάνοντας εκστρατείες ε, διεθνείς που θα υποστηρίζονται και θα βασίζονται σε, σε χρηματοοικονομικά μέσα, παρόμοια όπω γίνεται και με κάποια γεωργικά προϊόντα από πλευρά μα. Είμαι υπέρ τη νέα σύναψη νέων συνθήκων συμβάσεων για την αλληλεία με τρίτε χώρε που θα επιτρέπουν την πρόσβαση στον αλληλευτικό στόλο τη κοινότητα σε νέε αλληλευτικές περιοχέ είμαι υπέρ τη εκπώνηση συστημάτων γεωγραφική πληροφόρηση που θα επιτρέπουν την χωροταξική διάρθρωση και συντονισμό όσον αφορά τις αλληλευτικές δράσεις με βάση το πρότυπο του, ε, της οργάνωσης του Ευρωπαϊκού ε, Θαλάσσιου Χώρου που είναι άξονα της ε, ολοκληρωμένης πολιτικής μας. Σε σχέση με αυτή την έκθεση <clears throat> αντιμετωπίζω κάποια θέματα τα οποία πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα ζωτική σημασία και είναι ακαθόδη και δυσχερή και θα ήθελα πολύ να βασίζομαι στη δική σας άποψη και αξιολόγηση για αυτά. Υπογραμμίζω εδώ τρία από αυτά τα θέματα που θεωρώ είναι από τα πιο σημαντικά. Το πρώτο αφορά την αρχή της σταθερότητας, της ε, σχετικής σταθερότητας. Η σχετική σταθερότητα ήταν ένα μέσο που χρησιμοποιήθηκε κατά τις τελευταίες δεκαετίες για να διασφαλιστεί από τα κράτη-μέλη μια προνομιακή πρόσβαση στις δυνατότητες αλληλείας. Και ήταν ένας μηχανισμός ε, κατανομής των τάξ δίκαιος και σταθερός μακροπρόθεσμα στο χρόνο. Ωστόσο όμως πρέπει να διαρωτηθούμε σήμερα. Η εφαρμογή αυτής της αρχής ακόμα δικαιολογείται σήμερα λαμβάνοντας υπόψη τις πρακτικές που είναι κάθε φορά όλο και πιο κοινέ της αλλαγής, ανταλλαγής ποσοστώσεων μεταξύ κρατών μελών ή και της αλλαγής σημαία από πλευράς των αλλιευτικών επιχειρήσεων. Πώς μπορεί αυτό να διασφαλιστεί όταν έχουμε διαφορετικά συστήματα για τη διαχείριση της ε, αλίας από πλευράς μας, για την προσπάθεια της αλίας όταν μπορούμε να έχουμε αλλαγή ε, καθεστώτος με μεταφορά ποσοστώσεων. Εν ώψη αυτών των ερωτημάτων θα έπρεπε να προβληματιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη θέσπιση ενός ρυθμιστικού μηχανισμού που ενώ δεν θα διαμφισβητεί τα δικαιώματα των κρατών μελών από τη μία πλευρά Όσον αφορά την δυνατότητα εκμετάλλευσης των ε, υφιστάμενων αλληλευτικών δυνατοτήτων, θα πρέπει να διασφαλίζει μια σωστή διαχείριση. Ένα δεύτερο ζήτημα αφορά τα συστήματα ακριβώς διαχείρισης. Πιστεύω ότι είναι συνενετική αυτή τη στιγμή η τοποθέτηση ότι το σύστημα διαχείρισης αλίας μέσω των τάξ παρουσιάζει ευάλωτα στοιχεία και δεν έχει καταφέρει να επιλύσει τα θεμελιώδη προβλήματα της, του αλλιευτικού τομέα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο επιβάλλεται βαθύς προβληματισμός και ε, σοβαρές σκέψεις για να δούμε πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε μέχρι το 2005 τα αλλιευτικά αποθέματα στην κοινότητα να μπορέσουν να φτάσουν συγγνώμη, μέχρι το 2015 διορθώνει η ομιλήτρια, όχι 2005, 2005 είναι ήδη στο παρελθόν, 2015, να μπορέσουν να διασφαλίσουν την μέγιστη αηφόρο απόδοση. Πράγμα το οποίο κατά τα άλλα είναι και δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην συνάντηση του Johannesburg το 2002. Με αυτόν τον τρόπο συζητήθηκαν ήδη κάποιες εναλλακτικές οδοί και τρόποι, όπως είναι θέσπιση εναλλακτικών μεταφερόμενων δικαιωμάτων αλλιευμάτων, η διαχείριση των αλλιευμάτων στην προσπάθεια της ε, στην αλλιευτική προσπάθεια. Μέσα σε αυτά τα θέματα που έχουμε μπροστά μας πρέπει να δούμε ποιες είναι οι νομικές επιπτώσεις μιας ή περισσότερων τροποποιήσεων σε αυτό το επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη μελετήσει μελετησει και έχει προβλέψει επίσης ε, την, επι περιβαλλοντική επίπτωση και κοινωνική ε, και οικονομική επίπτωση των διαφορετικών εναλλακτικών σεναρίων όσον αφορά την διαχείριση των κοινοτικών προσπαθειών αλληλείας ταυτόχρονα και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιομορφίες που έχει η κοινοτική αλληλεία και που είναι τόσο διαφορετικές μεταξύ κρατών μελών θα πρέπει να διαρωτηθούμε αν διασφαλίζεται και δικαιολογείται αυτή τη στιγμή μια εξαντλητική ευρεία μελέτη που θα επέτρεπε μια ταυτοποίηση και έναν εντοπισμό σε σχέση με αυτά τα θέματα όσο αφορά τον ε, κοινοτικό στόλο. Σε σχέση με ένα πρότυπο διαχείριση και ένα, μια διαδικασία διαχείρισης, η διαχείριση των αλλιευμάτων δεν είναι θέμα αποκλειστικά τεχνικού χαρακτήρα εδώ θα πρέπει ο κοινοτικό νομοθέ, νομοθέτης να συνεχίσει να προσπαθεί να επιτύχει τους στόχους και να επιβάλλει τις κοινέ αρχές για τη διαχείριση της αλίας, καθώς επίσης λαμβάνοντας υπόψη και τα θεμελιώδη θέματα τα νομοθετικά για αυτή τη διαχείριση, χωρίς όμως να αμελεί, να αποκεντρώνει την ε, διάρθρωση των αποφάσεων όσον αφορά τεχνικά μέτρα και διατάξεις, δίνοντας σε κάποιες περιπτώσεις στα κράτη-μέλη ή ε, στην Επιτροπή ή και στις περιφέρειες και στον ίδιο ακόμα τον τομέα κλαδικά εξουσίες για την επίτευξη των στόχων που θα έχουν προσδιοριστεί προηγούμενα. Ένα τρίτο θέμα που εδώ θα ήθελα να παρουσιάσω αφορά τη διαχείριση, διαφοροποιημένη διαχείριση αλληλείας... Πράγματι θεωρώ ότι η πολυμορφία του τομέα της αλίας στην κοινότητα καθορίζει διαφορετικές προσεγγίσεις στα προβλήματα και διαφορετικές στρατηγικές για την επίλυσή τους. Ένας μικρός βιοτέχνης αλληλείας δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίζεται μέσα στο πλαίσιο της κοινή αλληλευτικής πολιτικής όπως ένας μεγάλος εφοπλιστής ή πλειοκτήτης ε, βιομηχανικής αλληλείας. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι η μεταρρύθμιση της κοινή αλλιευτικής πολιτικής θα πρέπει με ένα διαφοροποιημένο τρόπο να αντιμετωπίζει την διαχείριση διαφορετικών τύπων του στόλου. Η καθοριστική σημασία, το καθοριστική σημασία θέμα θα είναι η διαφοροποίηση μεταξύ βιοτεχνικής και βιομηχανικής αλίας. Σήμερα πράγματι με τις μεγάλες τεχνολογικές προόδους μια μικρή, ένα μικρό σκάφος δεν είναι υποχρεωτικά ένα μικρό βιοτεχνικό σκάφος, βιοτεχνικής ε, θα έλεγα χειροτεχνικής αλίας εδώ σε σχέση με το δυναμικό αλίας που διανοίγεται μπροστά του, σε σχέση με άλλου τύπου σκάφη. Δεδομένων λοιπόν όλων αυτών των θεμάτων που επέλεξα σε σχέση με την, ε, ε, το πιο επίμαχο που μπορεί να προκαλέσουν ως θέμα, <clears throat> θα ήθελα να, να προσκαλέσω να υποβάλλετε σχόλια και προτάσεις που θα εμπλουτίσουν τη συζήτηση και που είναι πολύ σκόπιμο ακόμα να διεξαχθεί και θα μπορέσουν να ληφθούν υπόψη στη συνέχεια για την εκπόνηση της τελικής έκδοσης αυτής της έκθεσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίασή σας και για το ότι θέσατε νομίζω τα θέματα αυτά τα οποία ακριβώς είναι τα πιο σημαντικά σε αυτή τη μεταρρύθμιση της ε, κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Πρώτα απ' όλα ζήτησε τον λόγο η κυρία Ανδρές Βάρια παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν πρώτα απ' όλα να συγχαρώ την εισηγήτρια για την παρουσίασή της έθιξε σχεδόν όλα τα σημεία τα οποία είναι σημαντικά για τη μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Και σε τέσσερα σημαντικά στοιχεία θα ήθελα να πω εδώ ότι ε, θέλω να κάνω κάποια σχόλια και συμφωνώ με αυτά βέβαια και θέλω να κάνω μια παρατήρηση το εξωτερικό κριτήριο σε σχέση με την, ε, τα διαφορετικά άλλα κριτήρια για τη διασφάλιση της αηφορίας για τα παιδιά μας και στο εσωτερικό επίπεδο, όπως πολύ καλά σχολίασε στην αρχή, της αποτελεσματικότητας και ανταγωνιστικότητας του στόλου μας. Πιστεύω ότι είναι αναγκαίο να γίνει μια πραγματική σε βάθος αξιολόγηση, αντικειμενική αξιολόγηση της κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε και του μέλλοντος που θα αντιμετωπίσουμε. Να γίνει αυτό χωρίς να ωρεοποιούμε πράγματα και χωρίς να ε, λέμε θέλουμε να διατηρήσουμε το στόλο αν δεν υπάρχει δυνατότητα διασφάλιση ενός μέλλοντος, μελλοντικής προοπτικής για αυτόν. Επίσης η σταθεροποίηση, η σταθερότητα το, και το θέμα των τάξ Πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα. Πρέπει να δούμε ότι ίσως δεν ήταν αποτελεσματική αυτή η διαχείριση έτσι και να βασιστούμε στο θέμα της αλληλευτικής προσπάθειας ουσιαστικά διανοίγεται μια νέα δυνατότητα, μια νέα προσέγγιση για να δοθούν λύσεις σε πολλά προβλήματα που, είναι, που πρέπει να αντιμετωπιστούν και τα τάξα και η κατάσταση όπως έχει που προκαλούν. Ένα τρίτο σημείο, ο έλεγχος και οι επιθεωρήσεις θεμελιώδες ε, θέμα και το θέμα της παράνομης αλίας επίσης, ε, αλλά και αυτά που κάνουν ε, οι αλλιευτικοί στόλοι στα κοινοτικά ύδατα. Η ανταγωνιστικότητα δηλαδή των αλλιευτικών, ας το περιοχών και εδώ θα πρέπει να ληφθεί μέγιστη πρόβλεψη και προφύλαξη για να μην υπάρχουν στρεβλώσεις. Και μία ε, θα έλεγα αξιολόγηση και πιστεύω ότι θα ε, συμφωνούσε εδώ η συγγήτρια να ενισχυθεί ο ρόλος ε, της γυναίκας και στο έγγραφο και στην αλληλευτική πολιτική. Είναι σημαντικό να πάρει πρωταγωνιστικό ρόλο η γυναίκα. Τον έχει αυτόν. Έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στα αλληλευτικά και θέματα που συνδέονται με τη θάλασσα και πρέπει αυτό να το τονίσουμε. Αυτό το έγγραφο θα πρέπει ακριβώς να αντανακλά το σημαντικό ρόλο των εργατικών χεριών, των γυναικών, της, του ρόλου της γυναίκας σε αυτόν τον τομέα. Είμαι βεβαία ότι θα το λάβει υπόψη και θα το δεχθεί η συγγήτρια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριος Φάρτον παρακαλώ. Uh, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ την συγγήτρια που μας ε, μίλησε για το συλλογισμό της ως τώρα. Υπάρχει ένα κατάλογο ζητημάτων ε, για τα οποία μίλησε και πιστεύουμε όλοι ότι θα πρέπει να γίνει μεγαλύτερη έρευνα, ότι πρέπει να έχουμε καλύτερη δατοκαλλιέργεια γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία, ειδικά στην Ήπεθρο. Ορθώς ε, αναγνώρισε ορισμένα ζητήματα ιδιαίτερης ε, δυσκολίας, όπως για παράδειγμα το θέμα της ε, σταθερότητας, ε, η δική μου άποψη, το πώς το βλέπουμε δηλαδή εμείς στη Σκοτία το θέμα της μεταρρύθμισης της κοινή αλληλευτικής πολιτικής, ε, η σχετική σταθερότητα είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Θέλουμε μια κοινή αλληλευτική πολιτική που θα ήθελαν να που θα δημιουργεί μια μεγαλύτερη σταθερότητα και για την αλλιευτική ε, δραστηριότητα στη Σκωτία. να υπάρχει μια κατανομία αλλιευτική ε, προσπάθειας ε, όσο το δυνατόν ε, πιο ισότιμη και πιο δίκαιη, ειδικότερα στοχευμένη σε συγκεκριμένες χώρες. Αυτή στιγμή θα υπάρξει κάποια συμφωνία σε θέματα φορολογίας, για παράδειγμα. Η Σκωτία, που είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο γνωρίζει πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα των των αλλιευμάτων, των μέγιστων επιτρεπόμενων αλλιευμάτων, των ποσοστώσεων. Είναι επίσης πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η Σκωτία έχει πολύ μεγάλο ποσοστό των ε, υδάτων αλίευσης Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, οπότε θα ήθελα να επαναλάβω κάτι το οποίο έχω πει πολλές φορές. Δεν έχουμε ε, μία λογική διαχείριση η οποία να εξασφαλίζει σε ένα συγκεκριμένο κλάδο, όπως για παράδειγμα ε, στην Αλία, στη Σκοτία, που να Τη δίνει τη δυνατότητα σε, πρόθεσμο χρονικό διάστημα να μπορεί να επωφεληθεί από μια βιώσιμη αλία. Να υπάρχει δηλαδή κοινοτική αλληλεία και κοινοτικά ύδατα αλλιεύσεις όπου δεν θα πηγαίνει κανείς να αλλιεύει όποιος προλάβει δηλαδή χωρίς ε, να τον ενδιαφέρει τίποτε άλλο. Να υπάρχει ένα σύστημα ε, και διατήρησης των αλλιευτικών πόρων, ώστε να γνωρίζουν όσοι ε, εργάζονται στον κλάδο ότι πρέπει να συμμορφώνονται με ορισμένα μέτρα τα οποία θα είναι απαραίτητα ε, κατά διάφορε χρονικέ περιόδου. Τώρα όσον αφορά την αποκέντρωση, νομίζω ότι τελευταία φορά που κάναμε τη συζήτηση όσοι ε, πήραν το λόγο ανέφεραν το θέμα αυτό σε κάποιο βαθμό, αλλά ευτυχώ. Ευτυχώ μεν που το συζητήσαμε, αλλά δυστυχώ η συγγήτρια μία ακόμη φορά το ανέφερε στο τέλο ε, τη Παρουσίασή τη. Ό,τι λοιπόν συζητηθεί ε, εδώ στις Βρυξέλλες, καλό είναι, αλλά η εφαρμογή δεν αρκεί να είναι αποκεντρωμένη. Θα έπρεπε να υπάρχουν πραγματικές αποφάσεις διαχείρισης, πραγματικές αποφάσεις για το πώς μπορεί να μεταρρυθμιστεί η αλληλευτική πολιτική. Ε, αυτές οι αποφάσεις πρέπει να γίνονται με αποκεντρωμένο τρόπο. Και αυτό είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό αν θέλουμε να επιτύχουμε κάτι το οποίο θα έχει κάποιο αποτέλεσμα. Δεν έχω να προτείνω κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο, αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι πιο επαναστατική η προσέγγισή μας σε σχέση με τους τρόπους λήψης αποφάσεων εδώ στις Βρυξέλλες και μετά της εκχώρησης κάποιων ε, συνηθισμένων καθηκόντων ε, σε αποκεντρωμένο επίπεδο δεν είναι τόσο πολύ σημαντικό αυτό όσο σημαντική είναι η διαχείριση των αποφάσεων αυτών. Να υπάρχει δηλαδή το κίνητρο της ε, συμμόρφωσης και να μάθουμε και από όλα τα προβλήματα ε, πραγματικής εφαρμογής που είχαμε στο παρελθόν. Αν δεν υπάρχει λοιπόν μια διαφοροποιημένη προσέγγιση, και νομίζω ότι και η συγχύτρια κάτι τέτοιο επιθυμεί, δεν θα υπάρξει και η αποκέντρωση. Το ένα συνδέεται άμεσα με τον άλλο. Το ένα συνδέεται άμεσα με το άλλο. Δεν ε, είναι θέμα μόνο ετησίων προσαρμογών είναι μια συνεχόμενη, μια συνεχιζόμενη διαδικασία και χρειάζεται συνεχόμενη ε, προσπάθεια διαχείρισης ε, με λογικό και δίκαιο τρόπο, γιατί δεν έχουμε μόνο κοινοτικό στόλο, έχουμε πολλούς στόλους σε διάφορες ε, θάλασσες και επομένως αυτό επηρεάζεται τις διάφορες περιφέρειες με διαφορετικό τρόπο. Κύριε Σπερέκ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, συγχαίρω την εισηγήτρια και την ευχαριστώ για τις εργασίες της. Αληθεύει ότι δεν είχε πολύ χρόνο στη διάθεσή της, αλλά τα κατάφερε πάρα πολύ καλά. Συγχαρητήρια. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για την υδατοκαλλιέργεια, γιατί αναφερθήκατε στην αρχή σε αυτό το θέμα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε το πλεονέκτημα και θα συνεχίσουμε να το έχουμε ε, το πλεονέκτημα λοιπόν της ολικής ε, ε, Αυτό δεν συμβαίνει όμως ε, όταν μιλάμε για τον τομέα αλλά στις τρίτες χώρες. Για τη σχετική σταθερότητα που αναφέρατε, δεν κρύβω ότι έχω κάποιες ανησυχίες σε σχέση με αυτή την αρχή των μεταβάσιμων ποσοστώσεων. Η θέσπιση αυτής της αρχής τουλάχιστον όταν ε, δεν ε, ορίζουμε την ελάχιστη χωρητικότητα του σκάφους ή το μέγεθος του σκάφους, μπορεί να οδηγήσει σε κερδοσκοπία σε σχέση με τις επιχειρήσεις και ε, άρα δεν θα επιτύχουμε το στόχο μας να διατηρηθεί και η ερασιτεχνική αλία, γιατί θέλουμε να την προστατεύσουμε όλοι. Θα είναι λίγαν επικίνδυνη αυτή η κερδοσκοπία γιατί θα μιλάμε για μεγάλες ομάδες ε, που θα συγκεντρώνουν τα μικρά σκάφη και θα θέσει αυτό σε κίνδυνο το ισχύον ε, αλληλευτικό μοντέλο. Ε, πρέπει να προσέξουμε. Αυτό το κριτήριο των μεταβάσιμων ποσοστώσεων ε, πρέπει να είναι συνάρτηση του προσδιορισμού ενός ελαχίστου μεγέθους σκάφους, ελάχιστης χωρητικότητας. Είναι απαραίτητο κατά τη γνώμη μου. Επίσης, ε, για Πρέπει να γίνει μια σωστή διάγνωση του αλλιευτικού, της αλλιευτικής υποδομής και του αλλιευτικού εξοπλισμού. Πρέπει να δούμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, είναι απαραίτητο. Και κάτι άλλο, όπως είπε και ο φίλος μας από τη Σκοτία, ε, και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε, υπάρχει η εδαφικοποίηση ή τουλάχιστον η περιφερειοποίηση των αποφάσεων ε, που θα λάβουμε ε, και αυτό είναι σημαντικό. Αντίθετα, ένα άλλο στοιχείο που δεν αναφέρθηκε αλλά έχει βαρύτητα είναι το θέμα των εισαγωγών. Αν δεν ελέγξουμε τις εισαγωγές, ε, είτε προέρχονται από την ε, υδατοκαλλιέργεια είτε από την αλία, ε, ουσιαστικά δεν θα βρούμε λύση και θα φάμε τα μούτρα μας. Μιλώντα για τι εξαγωγέ από τι τρίτε χώρε προ την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε μιλάμε για λιεύματα, είτε μιλάμε για προϊόντα εκτροφή. Πρέπει να περιορίσουμε και να προσδιορίσουμε τις, ε, το καθεστώ των εισαγωγών. Αυτά τα σχόλια είχα να κάνω για την έκθεση της εισηγήτριας, για το πράσινο πράσινη βίβλο και τη μελλοντική αλληλευτική πολιτική. Ούτως όλος θα μας ξαναδοθεί η ευκαιρία να συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχετε τον λόγο εσείς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με την παρέμβασή μου να ξεκινήσω ευχαριστώντας για το έργο της εισηγήτριας. Δεν μπόρεσα να την ακούσω ολόκληρη την εισήγηση από την αρχή, αλλά άκουσα προηγούμενα και κάποιες παρατηρήσεις ε, και γνωρίζω κάποιες απόψεις της. Θα ήθελα απλά και μόνο κάποια σημεία να αναφέρω που θα μπορούσαν να έχουν ενδιαφέρον όσον αφορά την αντιμετώπιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Πρώτον, κάποιες θεσμικές πτυχές με τη μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτική πολιτική, υλοποιούμε μέσα στο πλαίσιο της νέας αυτής συνθήκης τη Λισαβόνα, ένα φιλόδοξο έργο. Θα είναι σημαντικές οι μεταβολές ε, όσον αφορά τι εξουσίε των θεσμικών οργάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό πιστεύω ότι θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη ο ρόλος που θα διαδραματίζει η Ευρωβουλή μα και ταυτόχρονα ένα όραμα, ε, α το πω, μια προοπτική μελλοντική του τομέα στη μελλοντική διαχείριση τη αλίας. Όλα αυτά πρέπει είναι προφανέ να ληφθούν υπόψη στον αλληλευτικό τομέα που αναπτύσσεται μέσα σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία και γι' αυτό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι παράμετροι που θα έχουν επιπτώσεις ε, στον τομέα αυτό μέσα στο πλαίσιο των αλληλευτικών δραστηριοτήτων. Θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε μια ενσωματωμένη, ολοκληρωμένη προσέγγιση των δραστηριοτήτων του τομέα σφαιρική προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη και την έρευνα και, την, και για την ανάπτυξη. Συζητούμε διάφορα προγράμματα και σχέδια για την ανάκαμψη των πόρων και υπάρχουν πολλά κοινά ελλείψεις γνώσεων, ε, απουσία γνώσεων και στοιχείων. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα στοιχεία για να διασφαλίσουμε μια πιο αηφόρα ε, πολιτική αλίας αλλά επίσης να δούμε και τις εξορρυκτικές δραστηριότητες και βιομηχανικές δραστηριότητες. Όλα αυτά θα πρέπει να είναι σημείο αναφοράς για τέτοιου είδους δραστηριότητες και επιπλέον όσον αφορά τις σχέσεις στην ε, τροφική αλυσίδα. Τώρα έχουμε και κάποιες ε, μελέτες ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην, τροφοδο... τροφική αλυσίδα υπάρχει έμφαση στα γαλακτοκομικά προϊόντα αλλά και τα αλλιευτικά προϊόντα πρέπει εξίσου να λαμβάνονται υπόψη και όσον αφορά και τον ανταγωνισμό κάποια αναφορά θα έπρεπε να γίνει μέσα στο πλαίσιο τέτοιων ερευνών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι και το θέμα των κλιματικών αλλαγών. Οι κλιματικές αλλαγές θα έχουν τεράστιες επιπτώσεις ε, υπό πολυσχηδείς, ε, ας το πω έτσι, παραμέτρους, ε, αλλά και στον ενεργειακό τομέα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό, πρέπει να λάβουμε υπόψη για το μέλλον. Και όλα αυτά που αφορούν την ανάπτυξη του τομέα προς μια οικονομία, στο πω έτσι, πιο, αηφορ, πιο ε, αποτελεσματική στην αηφορία της. Υπάρχουν εδώ τρεις πτυχές που με ανησυχούν, τρία θέματα που με ανησυχούν. Η τροφική αλυσίδα, το ανέφερα αυτό πιο πριν, αλλά επίσης και ένα άλλο σε αυτά τα προϊόντα. Τα προϊόντα που ανταγωνίζονται στην αγορά. Κάποια, σαν συνέπεια, ε, α το πω έτσι, ε, εξορρυκτικών δραστηριοτήτων, άλλα λόγω εισαγωγών και εδώ έχουμε και το θέμα των πόρων που αφιερώνονται σε αυτόν τον τομέα από τρίτε χώρε. Πρέπει όμω οπωσδήποτε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει δίκαια αντιμετώπιση. Ισόπεδο, θα έλεγα, ε, ίσο πεδίο με έντιμου όρου ε, για τον ανταγωνισμό και την εμπλοκή όσων ενδιαφέρονται και μέσα στο πλαίσιο των διατάξεων του ΠΟΕ, Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, αλλά και ταυτόχρονα όλο μεγαλύτερη ποιότητα, θα έλεγα αναβαθμισμένη ποιότητα της πληροφόρηση για αυτά τα προϊόντα. Θεμελιώδες στοιχείο και αυτό. Εγώ απλά Δύο πράγματα θέλω να αναφέρω. Τη σημασία πρώτον ότι σε αυτήν την κοινή αλληλευτική πολιτική θα πρέπει να γίνει μια πολύ συγκεκριμένη αναφορά στο βιοτεχνικό τομέα αλληλείας, ιδιαίτερα για τον κοινωνικό, την κοινωνική σημασία και των προϊόντων που έχουν ιδιαίτερη αξία, αλλά και το θέμα των, ε, ε, θα έλεγα, ε, υδατοκαλλιεργειών και την εμπλοκή των γυναικών σε σχέση με τα, ε, τις ε, καλλιέργειες αυτές και να λαμβάνονται υπόψη οι γυναίκες και στην κοινή αλλιευτική πολιτική και σε σχέση με τις κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες. Επίσης, μία αναφορά πρέπει να γίνεται μέσα στο πλαίσιο της γενικής πολιτικής για τη σύναψη αλλιευτικών συμβάσεων. Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί και να παγιωθεί αυτή η πτυχή και να προσπαθήσουμε σε πολλές ε, περιπτώσεις σε σχέση με τρίτες χώρες να ε, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά μας, να μην είναι εις, βάρος δηλαδή αυτές οι συμβάσεις των, των ε, ε, ψαράδων, να προσπαθήσουμε να, είναι, να προασπίζουν τα συμφέροντά τους, να διασφαλίζεται η δραστηριότητά τους δηλαδή και η αεφορία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Λεβίν παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την ε, εισηγήτρια. Ήγηρε πολλά ε, σημαντικά ζητήματα. Η πράσινη βίβλος Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είναι καλή κατά τη γνώμη μου και είναι σημαντικό έγγραφο γιατί αναφέρεται σε όλα τα σημαντικά ζητήματα που πρέπει να ρυθμίσουμε. Αρχικά, θα ήθελα να υπογραμμίσω πόσο σημαντικό είναι να έχουμε μια βιώσιμη αλλιευτική πολιτική, γιατί έχουμε και την απειλή των κλιματικών αλλαγών σήμερα που θα επηρεάσουν ε, το οικοσύστημα της ε, θάλασσας ε, και η αλληλεία επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη σύνθεση, τα είδη που υπάρχουν στη θάλασσα. και επηρεάζουμε σε, μεγάλο βαθμό με την αλληλεία 70 έως 90% των ειδών και έχουμε μια, ένα αποτέλεσμα ντόμινο που επηρεάζει το οικοσύστημα και το καθιστά πολύ ευάλωτο. Χρειαζόμαστε σταθερά οικοσυστήματα για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την ε, απειλή της υπερθέρμανσης ε, του πλανήτη και της αλλαγής ε, στα θαλάσσια ρεύματα. Χρειάζεται λοιπόν ε, να έχουμε σταθερά οικοσυστήματα, σταθερή πρόσβαση στα αλλιεύματα για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρειαζόμαστε και μια βιωσιμότητα στον τομέα. Η δυναμικότητα στην αλληλεία είναι το σημαντικότερο πρόβλημα, δηλαδή έχουμε μεγάλους τόλους και όλα είναι και λιγότερα ψάρια. Ε, ε, αναφέρθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις διάφορες επιδοτήσεις ε, που δίνονται σε αυτά τα σκάφη για να συνεχίσουν να μπορούν να ασκούν την αλληλευτική δραστηριότητα χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αηφορία, διότι δεν υπάρχουν αρκετά ψάρια αλλά πρέπει να κατοχυρωθεί το εισόδημά τους παρόλα αυτά. Επίσης υπάρχει και το θέμα της ατέλειας των καυσίμων ε, είναι μια πολιτική που εφαρμόζεται στη χώρα μου και έγινε μια μελέτη η οποία δείχνει πως αν ε, επιδοτούμε 92 ιδιοκτή, ε, ιδιοκτήτες σκαφών με εκατομμύρια ευρώ, δεν μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ε, κλιματικές ε, αλλαγές. Ε, δεν είναι λογικό να επιδοτούμε τους ιδιοκτήτες αλλιευτικών σκαφών. Ουσιαστικά θα ε, χρειαζόταν να αναθεωρήσουμε το σύστημα των αλλιευτικών ε, προσπαθειών, ε, να δούμε ακριβώς τι ισχύει με την ατέλεια, όπως είπα, των καυσίμων και άρα φορολογικά κίνητρα για τη συνέχιση αυτών των αλλιευτικών δραστηριοτήτων και πώς όλα αυτά συνάδουν με μια βιώσιμη αλλιευτική πολιτική. Τώρα για το ΤΑΚ. Όταν μειώνεται το ΤΑΚ αυξάνονται οι διαμάχες διότι πολλοί αλήσε θα πρέπει να μεγιστοποιήσουν την αξία των αλλιευμάτων τους, να κάνουν το επωνομαζόμενο upgrading. Ε, αλλά προς το παρόν είναι και το ε, βέλτιστο δυνατό σύστημα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Η περιφερειοποίηση νομίζω είναι η σωστή οδός. Θα πρέπει να έχουμε ένα στόχο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να έχουμε τους ίδιους κανόνες παιχνιδιού, κυρίως ως προς τον έλεγχο και να ε, είμαστε αυστηροί. Να απαιτούμε από τον τομέα που έχει πρόσβαση στη φύση και στα άγρια ζώα χωρίς να καταβάλει το τίμα πρέπει να Απαιτούμε να έχουν εποπτεία, να, να έχουν ηλεκτρονικό ημερολόγιο στα σκάφη. Οι μεγαλύτεροι ιδιοκτήτες θα πρέπει να περιγράφουν συγκεκριμένα την δραστηριότητά τους, όπως και οι βιομήχανοι στη ξηρά, σε άλλους τομείς. Και εάν έχουμε μια υποπτία που θα βασίζεται στα αλλιευτικά δικαιώματα. Δεν πρέπει να εκχωρούμε, πώς να το πω, δωρεάν αυτά τα δικαιώματα. Θα πρέπει να θεσπίζουμε απαιτήσει για αυτούς που έχουν αυτό το προνόμιο να αλλιεύουν ε, θα πρέπει να έχουμε αυστηρότερα κριτήρια για όσους έχουν το προνόμιο να αλλιεύουν γιατί χρησιμοποιούν ε, τους πόρους που ανήκουν σε όλους μας. Ε, Όπω και η βιομηχανία στην ξηρά και εκεί ισχύουν αυστηρές απαιτήσει για τι εκπομπές ε, αερίων του θερμοκηπίου παραδείγματο χάρη Ε, και όταν υπάρχει υποψία ότι θα ανατώνονται ζώα ισχύουν ε, αυστηρέ απαιτήσει ε, και για τα ψάρια όμω δεν ισχύει αυτό και κάθε φορά που μειώνουμε το τάξα να λέω δημιουργούνται μεγάλες διαφορές και διαμάχες. Πρέπει να υπάρχουν απαιτήσει και πρέπει ο κλάδο να επομίζεται την ευθύνη του γιατί έχει αυτό το προνόμιο να αποκομίζει εισοδήματα αλλιεύοντα τους φυσικούς μας πόρους. Επίση, να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα ανάμεσα ε, με μεγάλους και τους μικρούς ε, ιδιοκτήτες ε, σκαφών και αλείς. Συμφωνώ με τον κύριο Κουντέκ όλοι θα πρέπει να προστατεύσουν ε, τους ιδιοκτήτες των ε, μικρών σκαφών, να δούμε ποιες λύσεις ε, υπάρχουν, πώς, πρέπει, πώς θα γίνει αυτή η διαφοροποίηση. Στην Δανία λειτουργεί καλά το σύστημα με τις διαβιβάσιμες ποσοστώσεις και την παράκτια λία όπου αλλιεύουν αυτά τα μικρά σκάφη κοντά στις ακτές δηλαδή λειτουργεί καλά αυτό το σύστημα και κατοχυρώνει μια σχετική σταθερότητα. Λοιπόν, αυτή η αρχή της σχετικής σταθερότητας είναι σημαντική. Πώς ακριβώς πρέπει να τοποθετηθούμε εμείς ε, μας απασχολεί εδώ και χρόνια αυτό το ζήτημα και έχει αλλάξει η κατάσταση όπως σωστά είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει αλλάξει το σύστημα ανταλλαγής των ποσοστώσεων ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Είναι λογικό όμως να διατηρήσουμε αυτό το σύστημα που βασίζεται στο ότι ε, οι χώρες που ιστορικά έχουν αλλιεύσει περισσότερο από τις άλλες θα πρέπει να συνεχίσουν να έχουν και τις υψηλότερες ποσοστώσεις. Εγώ θεωρώ ότι οι αλληλείς που αποδεικνύουν ότι αλλιεύουν με βιώσιμο τρόπο, αυτοί θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στους αλλιευτικούς πόρους, ε, να καταδείξουν ότι δεν καταναλώνουν πολλά καύσιμα, ότι αλλιεύουν επιλεκτικά, ότι δεν βλάπτουν ευαίσθητους βιοτόπους κτλ. Αυτοί πρέπει να έχουν τη μεγαλύτερη πρόσβαση. Ε, θεωρώ ότι αυτή θα πρέπει να είναι η θεμελιώδη αρχή. Ε, ε, τώρα, για τι αλληλευτικέ συμφωνίε με τι τρίτε χώρες, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με κάποιες τρίτες χώρες με τις οποίες έχουμε συμφωνία, γιατί επικρατεί πολιτική αστάθεια και σε αυτές τις χώρες και ότι θα πρέπει και εμείς ε, μέσω των συμφωνιών να στηρίξουμε τον κλάδο μου. Αυτό δεν συμβαίνει συχνά και στη σελίδα 24 της πράσινης ε, βιβλού βλέπουμε ότι υπάρχει χαμηλή ε, χρήση ή μηδενική χρήση των ε, αλλιευτικών πόρων και δεν υπάρχει πραγματική αλλιευτική πολιτική ε, σε αυτές ε, τις τρίτες χώρες και νομίζω ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε με σοβαρότητα και να αναθεωρήσουμε την πολιτική μας για τις τρίτες χώρες είναι πολύ θετικό που αρχίσαμε τη συζήτηση, είναι πολλά υποσχόμενη και ε, ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε ένα καλό κείμενο στο οποίο θα βασιστούμε για τις μελλοντικέ μας εργασίες. Ευχαριστώ. Ε, σε ευχαριστώ. Κύριε Κούν, παρακαλώ. Ε, σε ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω και εγώ στην εισηγήτρια την Μαρία Πατράου Νέβης να επενέσω την προσπάθειά της ε, την Ενώ και αυτό είναι έργο μας ως Κοινοβούλιο όσον αφορά την εκπόνηση, την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως εκτελεστικού σκέλους να έχουμε ένα καλό αντίβαρο, ας το πω έτσι, με το οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αποτελεσματικά. Το πιο αποφασιστικό ζήτημα φυσικά που τα ρυθμίζει, από το οποίο εξαρτώνται όλα και το γνωρίζουμε αυτό στην Επιτροπή Αλίας είναι πώς θα καταφέρουμε στο μέλλον να πετύχουμε τα αποθέματα μας τα αλλιευτικά να, να τα διατηρήσουμε και να τα προστατεύσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε ως οικονομικός παράγοντας σε πολλά κράτα μέλη μας να διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και στο μέλλον επίσης. Και εδώ σίγουρα μπορεί να έχει διαφορετική άποψη κάποιος, όμως από την άλλη πλευρά είμαι ακράδαντα πεισμένο ότι <clears throat> για τα αποθέματά μας θα πρέπει και με τα αντίστοιχα tax, τα total, total allowed catches, τα μέγιστα επιτρεπόμενα αλλιεύματα, να ρυθμίσουμε τα πράγματα έτσι ώστε για την αλληλεία και την μεταποιητική βιομηχανία να διασφαλίζεται ένα μέλλον στην Ευρώπη. Πολλές προσπάθειες λοιπόν πρέπει ακόμα να γίνουν. Και πρέπει να συζητήσουμε και αυτά τα θέματα αν θέλουμε να πετύχουμε μια νέα αλληλευτική πολιτική. Τι σημαίνει νέα πολιτική όμως ε, αλληλευτική πολιτική. Να, ε, να έχει δυνατότητες στο μέλλον. Πώς θα το καταφέρουμε λοιπόν στο μέλλον με, το, με τους στόλους στην αλία μας να πετύχουμε το δυνατόν τη μέγιστη αποτελεσματικότητα οικονομικά για τον οικονομιών μας. Αυτό είναι το ερώτημα. Και πρέπει να δούμε στη συνέχεια μήπως συμβαίνει ίσως το ότι η κοντινή στα παράκτια αλληλεία με ιδιαίτερο τρόπο θα έπρεπε ίσως να υποστατευτεί και να υποστηριχθεί και να πούμε να ορίστε εδώ πάρα πολλοί άνθρωποι μπορούν να έχουν θέση απασχόληση σε αυτόν τον τομέα πολιτικό μας έργο είναι ως ε, ε, αιρετοί εκπρόσωποι των πολιτών που είμαστε στην, Ευρωβουλή να δώσουμε τη μέγιστη προτεραιότητα σε αυτά τα θέματα. Και όσον αφορά τις τεχνικές δυνατότητες ε, για τους παράκτιους αλληλείς, ε, Φυσικά θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος των δραστηριοτήτων και όλες οι τεχνικές δυνατότητες θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε, να διασφαλίζεται η διαφάνεια. Δεν μπορούμε να πούμε για τους μικρούς επιχειρηματίες. Αυτοί θα διαφεύγουν των ελέγχων και μόνο οι μεγάλοι στόλοι θα μπορούν να ελέγχονται αποτελεσματικά. Όχι. Πρέπει όλες οι δυνατότητες να εκμεταλλευτούμε, να υφίστανται αυτά τα πλαίσια και αυτό είναι προϋπόθεση για το μέλλον. Αλλά δεν θα γίνουν όλα με την παράκτη αλία, δεν μπορούν όλες οι ανάγκες να καλυφθούν, το ξέρουμε και αυτό. Οι οικονομίες μας έχουν τέτοια τάση, ας το πω έτσι, που εξαρτώνται και από τα μεγάλα, τις, τα, ας το πω έτσι, την βιομηχανική αλληλεία με, με μεγάλα αλλιεύματα και αυτό είναι σημαντικό στοιχείο μέσα σε όλα αυτά. Και έτσι πιστεύω ότι η συγγήτριά μας κατάφερε πολλά σημαντικά σημεία να καλύψει στην έκθεσή της. Και θα έλεγα σίγουρα από την άλλη πλευρά ότι θα έπρεπε να προβληματιστούμε τι θα γίνει με τις χιλιάδες χιλιόμετρα ακτών παρακτήων περιοχών που έχουμε στην Ευρώπη. Από πάρα πολύ, ας το πω έτσι, όμορφα μικρά λιμάνια βιοτεχνικής αλίας μικροαλληλαίων που από τους τουρίστες επιλέγονται ως στόχοι των ταξιδιών τους για τουρισμό. Θα πρέπει και εδώ να προβληματιστούμε να δούμε πώς πραγματικά μπορούμε να καταφέρουμε την ιστορική αυτή και πολιτιστική κληρονομιά που έχουμε σε σχέση με την αλία, να μην αμελήσουμε την αλία να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε τέτοιου είδους ε, περιοχές που ασχολούνται με την κοντινή στις ακτές αλληλεία. Αλλά ταυτόχρονα να τονώσουμε και την ε, δυνατότητα στις ε, τουριστικές περιοχές της μεταποίησης των αλλιευμάτων, του καπνίσματος των ψαριών, της μεταποίησης Ταυτόχρονα φυσικά η αλληλεία ανοιχτή θαλάσση πρέπει να συνεχιστεί. Είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό. Έχουμε μεγάλε επιχειρήσει που ασχολούνται με την μεταποίηση αλλιευμάτων. Αλλά αυτά τα θέματα τα οποία απορρέουν από αυτή την εξέλιξη πρέπει να τα συζητήσουμε από κοινού. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρο. Ο κύριο Κάγκλουγκ παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που παίρνω το λόγο. Δεν χρειάζεται όμως να επαναλάβω και όλα αυτά που ακούσαμε. Νομίζω ότι πάνω κάτω συμφωνούμε για πολλά ε, από αυτά τα σημαντικά ζητήματα. Πρέπει να προωθήσουμε αυτές τις εργασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και θα έπρεπε να βρούμε μια κοινή προσέγγιση. Σε αυτό το στάδιο και ε, ζωτική σημασία είναι να έχουμε μια πράσινη βίβλο που θα ορίζει τις προκλήσεις τις οποίες καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε και με κριτικό μάτι πρέπει να ε, προσδιορίσουμε τα προβλήματα και τις ε, οδούς που θα ακολουθήσουμε για να τα επιλύσουμε. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε και το θάρρος και την τόλμη να λάβουμε τις δύσκολες αποφάσεις ε, που μας, περιμένουμε, που μας περιμένουν. Ας αρχίσω με το θέμα των μικρών σκαφών που αναφέρθηκε από πολλούς ε, συναδέλφους. Πρέπει να προστατεύσουμε και τους εραστέχνες ελίες και τους ιδιοκτήτες μικρών αλληλευτικών σκαφών υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες ε, σχετικά με το αν θα υπάρξει διαφοροποίηση της αλληλευτικής πολιτικής και φυσικά το βάρος πρέπει να ρίχνεται στη βιωσιμότητα αυτής της πολιτικής. Το βασικό είναι η προσέγγιση μας ε, να αποσκοπεί στην προστασία του οικοσυστήματος και αυτό θα πρέπει να είναι και το εφαλτήριό μας. Θα ήθελα να αναφερθώ στον κύριο Όστρομ που κέρδισε τον Νόμπελ φέτος και έχει μελετήσει τη διαχείριση την ε, δημόσια διακυβέρνηση ε, στον κλάδο και μίλησε για την ε, αυτοδιακυβέρνηση, self-governance και ότι αυτή είναι η καλύτερη οδός που έχουμε να ακολουθήσουμε. Ε, δηλαδή πρέπει να αποφεύγουμε τους άκαμπτους ε, κανόνες ε, διαχείρισης και να κάνουμε όλοι μαζί κάτι για να επιτύχουμε τα αποτελέσματα που επιθυμούμε. Για την περιφερειακή προσέγγιση Ελπίζω να μπορέσουμε να ορίσουμε ακριβώς ε, τι εννοούμε με την περιφερειακή διαχείριση ελευτικής πολιτικής, δηλαδή σε πολιτικό επίπεδο να συμφωνήσουμε ακριβώς ε, τι επιδιώκουμε ε, για τις επιδοτήσεις που θα δώσουμε και στήριξη που θα δώσουμε, τόσο ώστε σε περιφερειακό επίπεδο να υπάρχει διαχείριση της πολιτικής. Σε πολλά φόρα στην Ευρώπη έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα και πρέπει να διαπιστώσουμε ακριβώς ποιοι κοινοί κανόνες υπάρχουν και αν θέλουμε περιφερειακή ε, προσέγγιση ε, δεν χρειάζεται να περιοριζόμαστε στη συζήτηση για τους ισχύοντες κανόνες. Πρέπει να δούμε οι ίδιοι που τι μπορούν να κάνουν για να συμβάλλουν στην αλληλευτική πολιτική. Τώρα για την αλλιευτική ικανότητα. Πρέπει να ε, εξασφαλίσουμε την βιωσιμότητα του αλλιευτικού στόλου και να προστατεύσουμε και τις οικονομίες που εξαρτώνται από την αλληλεία. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη πρόκληση. Ξαναλέω ότι θα πρέπει να έχουμε το θάρρος να πάρουμε τις αποφάσεις που χρειάζεται ε, και ε, ο σκιώδης εισηγητής από την ομάδα μας ε, θα βοηθήσει την εισηγήτρια για να εμβαθύνει αυτά τα ζητήματα. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Χάγκλουν. Τώρα η κυρία Ντόμψη παρακαλώ. you, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και την εισηγήτρια Συγγνώμη που έχασα ένα τμήμα της παρουσίασής σας, αλλά από την συζήτηση που άκουσα μπορώ να πω ορισμένα πράγματα. Όταν και η μεταρρύθμιση κοινή αλληλευτικής πολιτικής, υπήρχαν πολλοί αλληλείς και εκπρόσωποι του κλάδου με τους οποίους ε, συνομίλησε, που ήταν κάπω σκεπτικοί κατά πόσο θα ήταν πράγματι μία μεταρρύθμιση ή μήπω ε, μήπως θα ήταν ε, ξανά τα ίδια δηλαδή στην αλληλευτική πολιτική αυτό που νομίζω ότι εμείς πρέπει να κάνουμε ως Επιτροπή ώστε να εξασφαλίσουμε ότι και οι αλληλείς και οι εκπρόσωποι του κλάδου ε, είναι να τους δείξουμε ότι μας ενδιαφέρει μια πραγματική μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Και αυτό σημαίνει και αναφέρομαι και σε αυτά που είπε ο Σκοτσέζο συνάδελφος πρέπει να υπάρχει μια αποκέντρωση της ευθύνη προς τις περιφέρειες για τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις περιφέρειες. Πολλοί από τους συνομιλητές μου μου είπαν ότι ο ρόλος της Βρυξέλλες θα ήθελαν απλώς να, να, είναι, να θέτει τις πολιτικές και μετά να δίνει τη δυνατότητα στις περιφέρειες να δράσουν ε, σε τοπικό επίπεδο ε, εντός των οργανώσεών τους. Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να πω κάτι ακόμη. Η τελευταία μεταρρύθμιση τη κοινή αλληλευτική πολιτική ίδρυσε τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια που έδιναν τη δυνατότητα στους αλληλεί και στους εκπροσώπους του κλάδου να δίνουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξισορροπημένη ε, θεώρηση της κατάστασης ε, και των τελευταίων εξελίξεων. Υπάρχουν πολλοί ε, αλληλείς και συμμετέχονται στα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια που ανησύχησαν όταν είδαν ότι υπάρχει ένας νέος κανονισμός τον οποίο ε, παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο γιατί ανησυχούν ότι θα υπάρξει μία ακόμη προσπάθεια ε, πίεσης ώστε να υπάρχει ένας τεχνικός κανονισμός που θα περάσει στο Συμβούλιο τον Νοέμβριο. Αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε έναν πραγματικό ρολό σκηνοβούλιο και αν θέλουμε ο, ο κλάδος να έχει ένα πραγματικό λόγο, τέτοιου είδους ε, δραστηριότητες πρέπει να αντιμετωπιστούν και από εμάς και από τους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής αν είναι εδώ σήμερα. Θα ήθελα να πω ότι η Εθνική Ομοσπονδία ε, Οργανώσεων Ολιαίων ε, Μα είπε σε σχέση με το τι συνέβη τον Οκτώβριο και το τι θα συμβεί κατά πάσα πιθανότητα τον Νοέμβριο είναι ότι η μεταρρύθμιση πρέπει να ε, συνοδεύσει την θέση σε ισχύ της ε, συνθήκη της Λισαβόνα, να υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στον αλληλευτικό κλάδο και να μην υπάρχουν πλέον αντιφάσεις. Στην πράσινη βίβλο ε, αναφέρεται ότι αυτή η Αναφέρεται ότι είναι λάθος αυτή η από πάνω προ τα κάτω προσέγγιση του κλάδου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να δουλέψει πολύ σκληρά για να αποδείξει στους αλληλεί και στον κλάδο ότι πιστεύουν αυτά που αναφέρονται στην ε, πράσινη βίβλο και ότι δεν θα συνεχίσουν ε, να επιβάλλουν κανονισμούς ε, πριν από την μεταρρύθμιση της κοινή ελευτικής πολιτικής. Πρέπει να συνεργαστούμε, όχι να μας τα υπαγορεύει όλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέτοιου είδους βήματα δείχνουν στους αλληλείς ότι ενώ γίνεται η μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής δεν την έχουμε πάρει επαρκώς στα σοβαρά και νομίζω ότι εμείς ως Επιτροπή πρέπει να δουλέψουμε πολύ σκληρά για να εξασφαλίσουμε ότι ο κόσμος καταλαβαίνει ότι έχουμε πάρει σοβαρά την κοινή αλληλευτική πολιτική και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να το δείξει αυτό στην πράξη με τις πράξεις της και το τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι ε, ε, επειδή πλησιάζει και η προθεσμία ε, αντίδρασης ε, και σχολιασμού της ε, ε, πράσινης βίβλου, νομίζουμε ότι πρέπει να συμμετέχουν πιο ενεργά οι αλληλείς και οι εκπρόσωποι του κλάδου και αυτό είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να το πω, να επιμείνω σε αυτό. Πρέπει να υπάρχει συνεχιζόμενη δέσμευση και συμμετοχή των αλλιέων από όλα τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. <coughs> Ο κύριος Αντινόρο παρακαλώ. Io per complimentarmi con la relatrice anche se è contemporaneamente. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχά, επιτρέψτε μου να συγχαρώ την εισηγήτρια και να τη ζητήσω και συγγνώμη αν δεν την άκουσα από την αρχή, αλλά άκουσα ένα μεγάλο τμήμα τη παρουσίασή τη. Ε, θα ήθελα απλώ να σα πω να κάνω κάποιε παρατηρήσει. θα ήθελα να πω ότι δεν είναι απλό αυτό που μας περιμένει. Αυτό μπορώ να το πω με βεβαιότητα, γιατί πρέπει να υπάρξουν κοινοτικοί κανόνες, να υπάρχουν ε, οι τοπικές απαιτήσει που θα ληφθούν υπόψη, όπως επίσης και η οικολογική βιωσιμότητα. Γνωρίζουμε ότι είναι ουσιαστικής σημασίας και για τις δεκαετίες που θα ακολουθήσουν σε ένα κόσμο που είναι πραγματικά πολύ περίπλοκος. Οι εργασίες που δρομολογούνται σήμερα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μου έμαθαν πολλά πράγματα. Κανένας δεν γνωρίζει πλήρως το σύνολο του κλάδου και εγώ έχω λιγότερες ε, τεχνικές γνώσεις ε, από εσά, αλλά η ουσία είναι να ληφθούν υπόψη όλες οι ιδέες. Οπότε, μιλούμε για περιφερειοποίηση. Ε, πρέπει να ξέρουμε και τι είναι η περιφερειοποίηση, γιατί η Βαλτική θάλασσα δεν είναι ίδια με τη Μεσόγειο. Στη Μεσόγειο μπορεί να μην υπάρχουν οι ίδιες ε, απαιτήσει που υπάρχουν στο Βορρά. Η περιφερειοποίηση, συνεπώς, είναι κάτι στο οποίο όλος ο κόσμος αναφέρεται, αλλά μπορεί από την περιφερειοποίηση να μην καταλαβαίνουμε όλοι το ίδιο πράγμα και παρόλα αυτά πρέπει να βρούμε μια κοινή λύση. Ένας συνάδελφος προηγουμένως είπε ότι θα έπρεπε να επανέλθουμε στην ιστορία ε, γιατί και, και συμφωνώ με αυτό που είπε γιατί δείχνει τη σημασία της βιομηχανικής αλίας, η οποία μπορεί ενδεχομένως σε κάποια τμήματα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης να δουλεύει καλά, αλλά σε άλλα όχι. Υπάρχει η αριστεχνική αλία, πρέπει και αυτή να τη λάβουμε υπόψη, τέλος πάντων του τουρισμού που έχει σχέση και με την αλία. Άρα πρέπει ε, οι ίδιες οι περιφέρειες να μπορούν να διαχειρίζονται ε, τις, την αλλιευτική τους δραστηριότητα με ε, ε, δραστηριότητες οι οποίες θα οδηγούν σε μια εναλλακτική οικονομία και ελπίζω ότι αυτό το, αυτή, η νέα, ε, αυτή η πράσινη βίβλος για την κοινή αλλιευτική πολιτική θα μας δώσει γενικούς προσανατολισμούς αλλά, και ζητώ στο σημείο αυτό από την εισηγήτρια να το ε, αποσαφηνίσει σε ορισμένα κεφάλαια που πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι, να δώσουν συγκεκριμένες, να δώσουν συγκεκριμένες ενδείξεις στα κράτη-μέλη και βεβαίως να υπάρξουν και συγκεκριμένε οδηγίε προ τι περιφέρειες. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι δυνατόν να το παρατραβήξουμε και να μπούμε σε πάρα πολλέ λεπτομέρειε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η αλήθεια είναι ότι αν παραμείνουμε από την άλλη πάρα πολύ αόριστοι και ασαφεί, σε μερικά χρόνια θα ξαναχρειαστεί μεταρρύθμιση τη κοινή αλληλευτικής πολιτική. Ελπίζω να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε σε μια πραγματική κοινή αλληλευτική πολιτική ε, και μικρή κλίμακα και μεγάλη κλίμακα, να ανακαλύψουμε εκ νέου όλες αυτές τις περιφέρειες ε, όπου ε, η αλληλεία θεωρείται ένας φτωχός κλάδος, αλλά δεν ισχύει πάντοτε. Ευχαριστούμε κυρία Ρόντος, παρακαλώ. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα θερμά να ευχαριστήσω τη Μαρία για την εξαιρετική δουλειά που έκανε. Υπέροχη δουλειά. Ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της πίεσης χρόνου μέσα στην οποία αυτή η πίεση χρόνου εργάστηκε Θέλω όμως να ευχαριστήσω και σε σχέση με την ομάδα εργασίας μας που πάντα μας ενημέρωνε όπως έπρεπε. Εδώ συζητάμε για την κοινή αλληλευτική πολιτική, για την αντιστάθμιση, ισορρόπηση αφενός των προσπαθειών αλλίευσης, από την άλλη πλευρά διατήρησης όμως των αποθεμάτων και προστασίας του περιβάλλοντος και προστασία των θέσεων απασχόλησης. Και αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο ως εγχείρημα για μας να βρούμε τη σωστή ισορροπία των παραγόντων. Με τη μεταρρύθμιση του 2002, ήδη ο στόχος της αηφορίας στην αλλιευτική πολιτική και σημαντικές άλλες αρχές όπως διατήρηση του οικοσυστήματος ε, και της διασφάλισης αηφορίας. Κατοχυρώθηκαν αυτά. Παράλληλα όμως ε, και τα οικονομικά προγράμματα και σχέδια και η περιφερειακή γνωμοδοτική διάσταση των συμβουλίων και η καταπολέμηση της παράνομης αλίας είναι σημαντικά μέτρα τα οποία ελήφθησαν ε, και θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτές τις προσπάθειες. Ως πρόσθετο μέσο όμως θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει απαγόρευση απορρίψεων ή απαγόρευση εκφόρτωσης τέτοιων αλλιευμάτων. Ταυτόχρονα χρειάζονται αναγκαία συγκεκριμένα μέτρα ώστε να δούμε πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ευάλωτα είδη και ευάλωτες ε, περιοχές αλλιευμάτων. Το θέμα της ε, σχετικής ε, σταθερότητας από το δικό μας πρίσμα είναι κάτι που απορρίπτουμε. η απαγορευση εκφορτωσης τετοιων αλλιευματων ταυτοχρονα χρειαζονται αναγκαια συγκεκριμενα μετρα ωστε να δουμε πως μπορουμε να διασφαλισουμε ευαλωτα ειδη και ευαλωτες περιοχες αλλιευματων το θεμα της σχετικης σταθεροτητας απο το δικο μας πρισμα ειναι κατι που απορριπτουμε πιθανή εισαγωγή εμπορεύσιμων ποσοστώσεων και ανταλλάξιμων ποσοστώσεων είναι κάτι που με κριτικό πνεύμα, με επικρίσεις αντιμετωπίζουμε. Έτσι λοιπόν θα καταθέσουμε τροπολογίες ως προς αυτά. Ευχαριστώ. Sí, bueno, ναι, σας ευχαριστώ. Δεν έχουν ζητήσει άλλη τον λόγο. Και τώρα θα παρέμβω και εγώ για να δώσω κάποιες σκέψεις που έχω στην εισηγήτρια και φυσικά και θέλω και εγώ να συγχαρώ διότι όπως αναφέρθηκε ε, κάλυψε τα ουσιοδέστερα προβλήματα και θέματα στην Πράσινη Βίβλο για την κοινή ελευθερική πολιτική. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια αλληλευτική πολιτική που θα είναι αηφόρος, όπως αναφέρθηκε. Αλλά για την αηφορία, η αηφορία δεν μπορεί να είναι απλά μόνο περιβαλλοντική. Πρέπει να είναι και οικονομική και κοινωνική αηφορία ταυτόχρονα. Πρέπει να μετράτε λοιπόν η αηφορία ως προς αυτούς τους παράγοντες και για την κοινή αλληλευτική πολιτική πρέπει να το δούμε ότι δεν πρέπει να θεωρείται μόνο αποτελεσματική με κάποια ανανεώσιμα κριτήρια. Πρέπει να είναι μια οικονομικά αποδοτική δραστηριότητα που θα λειτουργεί αποτελεσματικά. Τον παράγοντα της απόδοσης και αποδοτικότητας είναι κάτι που πρέπει να το δούμε μέσα σε αυτό το πρίσμα. Να είμαστε αποτελεσματικοί στην αλληλεία μας το κυριότερο πρόβλημα της κοινή αλληλευτικής πολιτικής είναι το θέμα της διαχείρισης ε, και ε, διατήρησης ε, των αλλιευμάτων. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να το δούμε. Τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε τώρα στην κοινή αλληλευτική πολιτική, εγώ θεωρώ ότι είναι το υπερπλεονάζον δυναμικό που έχουμε ε, από τον αλλιευτικό στόλο και υπεραλή, η υπεραλίευση. Εδώ πρέπει να διαχειριστούμε σωστά τα πράγματα όσον αφορά την υπεραλίευση που προώθησε τις απορρίψεις. Αλλά να έχουμε ένα σύστημα που, όπως αυτό που έχουμε σήμερα των ποσοστώσεων προωθούμε με αυτόν τον τρόπο τα, απορρί, τα, τις απορρίψεις. Πρέπει εδώ να έχουμε και είναι απόδειξη τα καλά προγράμματα ανάκαμψης. Ε, είναι όμως όλα αυτά πολύ δύσκολο να ελεγχθούν και όσους και ε, ε, όσες διατάξεις και να έχουμε για ελέγχους η έλεγχη των εκφορτώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τέτοιον αριθμό, μεγάλον αριθμό σκαφών είναι πολύ δύσκολο, ανέφικτο πράγμα. Πρέπει να καταλήξουμε σε συστήματα πολύ πιο αποτελεσματικά. Από την άλλη πλευρά έχουμε ένα σύστημα που όπως ε, ε, αφορά τις ε, αρχές της συνθήκης, δηλαδή την ελευθερία της πρόσβασης, Βρισκόμαστε σε ένα σύστημα το οποίο ε, πολλές φορές αντιβαίνει τους ε, όρους ε, της ενιαίας εσωτερικής αγοράς με όρους εθνικοποίησης και πρέπει να δούμε και το θέμα των ποσοστώσεων. Αν πρέπει να συνεχίσουμε με, αυτά τα, με αυτές τις μάστιγες που δεν λειτουργούν καλά. Έχουμε και δύο πτυχές που υποχρεωτικά θα πρέπει να μας κάνουν να αλλάξουμε αυτό το πρότυπο. Είναι η μέγιστη απόδοση, έχουμε δέσμευση όσον αφορά το Johannesburg όσον αφορά αυτά και την ε, οικολογική ε, προσέγγιση που είναι και αυτό κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Έχουμε παγκόσμιες διεθνείς δεσμεύσεις εδώ. Αυτές οι επικεντρώσεις πρέπει υποχρεωτικά να μας κάνουν να αλλάξουμε το σημερινό σύστημα αληθεύει το ότι το οικολογικό ε, συστημικό πλαίσιο απαιτεί μια επικέντρωση διαφορετική στην έρευνα που δεν έχουμε προετοιμάσει όπως πρέπει. Και αυτό θέλω να πω. Βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα πρέπει να δοθούν λύσεις σε αυτό. Το θέμα της μέγιστης αηφορίας ε, είναι κάτι που πρέπει να το δούμε. Εδώ είχαμε και επίμαχο θέμα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η μέγιστη απόδοση δεν μπορεί αναλύευμα να εξετάζεται, διότι στο τέλος τέλος θα καταφέρουμε να μειώσουμε τα τάκ και βλέπουμε ότι δεν λειτουργούν τα πράγματα με μειώσει των τάκ. Αλλά η μέγιστη αηφορία, αποτελεσματική αηφορία πρέπει να εξετάζεται αναειδιομορφία του είδους. Εδώ, ανάλογα με τον, το σύστημα ελέγχου αναείδος και αναπροσπάθεια θα μας δώσει αποτελεσματικότητα και θα αποφύγουμε τις απορρίψεις. Έτσι θα έχουμε και για τη βιομηχανική αλία ένα σύστημα ατομικών μεταφερο... μεταφερόμενων δικαιωμάτων. Και αυτό είναι πολύ αποτελεσματικό για την αντιμετώπιση της, ε, του υπερπλεονάζοντος δυναμικού. Ε, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πολλούς που παρενέβησαν, πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τους ε, στόλους μας. Το είπαμε από το 1996 το θέμα των ε, παράκτιων αλλιέων και το θέμα των βιομηχανικών αλλιέων είναι το ένα διαφορετικό από το άλλο και πρέπει να τα δούμε διαφοροποιημένα. Ε, ε, απασχολεί πολύ περισσότερα άτομα η παράκτεια βιοτεχνική αλληλεία από τη βιομηχανική αλληλεία και πρέπει να δούμε το πρότυπο διαχείρισης που θα υιοθετήσουμε. Υπάρχει ένα ουσιώδες όμως στοιχείο. Πρέπει να καθορίσουμε και πρέπει να εντοπίσουμε, να τα, ε, ταυτοποιήσουμε στην έκθεσή μας, να προσδιορίσουμε την βιοτεχνική αλληλεία. Δεν ξέρω αν αυτό θα εξυπηρετήσει πανευρωπαϊκά την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι αν θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε μεταξύ στόλων. Πρέπει όμως να καθορίσουμε κάποια πράγματα. Το όριο των 12 μιλίων, για παράδειγμα, μια ζώνη που πρέπει να συνεχίσει να διασφαλίζεται, πρέπει οπωσδήποτε όμως να καθορίσουμε, να προσδιορίσουμε κάποια πράγματα και έτσι να δοθεί ένα σύστημα το οποίο θα μπορεί αποτελεσματικά να λειτουργεί. Μια και είναι αυτό το οποίο είναι αποτελεσματικό. Και παράλληλα με το θέμα των βιοτεχνικών, των βιοτεχνών αλλιέων, έχουμε και την αποκέντρωση. Εδώ γίνεται λόγος για αποκέντρωση Ελπίζω ότι δεν θα αναφέρουμε επανεθνικοποίηση, γιατί και αυτό είναι αποκέντρωση. Εγώ φυσικά είμαι όχι υπέρ μιας επανεθνικοποίησης, αλλά υπέρ μιας σημαντικής αποκέντρωσης. Και στην βιοτεχνική αλληλεία, εκεί όπου η προσπάθεια στο περιφερειακό επίπεδο μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα από ότι η προσπάθεια στο κοινοτικό, στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Εδώ θα πρέπει να δούμε τη βιοτεχνική αλία σαφώς σε ένα αποκεντρωμένο πλαίσιο. Αποκεντρωμένο πλαίσιο και της διαχείρισης ακόμα. Και εδώ προσωπικά θα έλεγα ότι εγώ είμαι υπέρ αυτής της αποκεντροποιημένης διαχείρισης, αλλά όχι επανεθνικοποίησης. Εντάξει, υπάρχει ένα σημαντικό θέμα το οποίο προανέφερα. Είναι το θέμα του υπερβάλλοντος υπερβολικού αλευτικού δυναμικού και της υπεραλίευσης. Πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν πρότυπα διαχείρισης ε, που λειτουργούν, ε, για την, μπορούν να λειτουργήσουν για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Αν θέλουμε πρότυπα να είναι αποτελεσματικά πιο πριν, πρέπει να κάνουμε βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μία ανάλυση, μία συγκεκριμένη πρόταση για τη μείωση του δυναμικού. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αναφέρει αυτό το θέμα, αλλά η υποχρέωση που έχουμε όλοι μας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κράτη-μέλη κτλ, κτλ, είναι να κάνουμε μια αποτίμηση, μια αξιολόγηση ποιο, σε ποιο τομέα της αλίας υπάρχει αυτό το υπερπλεονάζον δυναμικό. Γιατί πρέπει άμεσα να το αντιμετωπίσουμε. Δεν πρέπει να πούμε είναι το υπερπλεονάζον δυναμικό αυτό το οποίο δημιουργεί το πρόβλημα τελεία και παύλα. Να δούμε πού υπάρχει πλεονάζον δυναμικό και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε εκεί όπου υφίσταται γιατί δεν είναι όλοι οι κοινοτικοί στόλοι μας ίδιο ένας με τον άλλον και υπάρχουν διαφορές και αυτό πρέπει να εντοπίσουμε να δούμε και σε σχέση με τους οργανισμούς που προαναφέρθηκαν επίσης για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτή την προσπάθεια να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα θα πρέπει να υπάρξει ένα ταμείο για τα προβλήματα ε, αυτά. Νομίζω μεγάλο, πρόβλημα του, μεγάλο μέρος του προβλήματος που υπήρξε για τις ελλείψεις στη διαρθρωτική πολιτική οφείλεται στο ότι πολλά κράτη-μέλη δεν βοήθησαν με κανένα τρόπο σε σχέση με τους στόλους τους και σε σχέση με τα προβλήματα αυτά συνέχισαν να υφίστανται. Πρέπει αυτά τα προβλήματα όμως να τα αντιμετωπιστούν σε κοινοτικό επίπεδο, να έχουν όλοι τις ίδιες δυνατότητες πρόσβασης ε, και να μην έχουμε μόνο διαφοροποιημένη αντιμετώπιση σε σχέση με την αφαίρεση, απόσυρση πλοίων όσον αφορά κάποια κράτη. Αυτές είναι οι πρώτες αναφορές που θα ήθελα να κάνω σε ένα τέτοιο θέμα τεράστιο ενδιαφέροντος για την κοινοβουλευτική μας Επιτροπή και είναι αυτονόητο ότι δεν θα ασχοληθώ με θέματα αγοράς ή εξωτερικής πολιτικής. Όμως θέλω να πω, το θέμα της εξωτερικής πολιτικής μου φαίνεται το πιο αδύναμο από όλα στην Πράσινη Βίβλο. Κάνει μια αυτοκριτική η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμφωνώ με κάποια από τα στοιχεία αυτοκριτικής, αλλά δεν προτείνονται λύσεις. Το θέμα της εξωτερικής πολιτικής πρέπει να το ξαναδούμε σε σοβαρό πλαίσιο και σε βάθος και να ξαναδούμε τι πρέπει να γίνει σε σχέση με την αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για κάποια θέματα. Πρέπει να δούμε ποιες λύσεις θα επιλεγούν και θα δοθούν. Εγώ υπό το πρίσμα της νομικής αυτής προσέγγισης, νομοθετικής προσέγγισης, είμαι υπέρ του να δοθούν λύσεις, αλλά δεν με πείθει μια ε, αυτοκριτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά μετά να μην δίνει λύσεις, να μην προτείνει τίποτα. Πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα. Ίσως αυτό δεν είναι το πιο κατεπήγον για την ε, έκθεση αυτή που είναι σε πρώτο επίπεδο από πλευρά σας. Πρέπει όμως στο πλαίσιο της κοινή αλληλευτικής πολιτικής να δώσουμε κάποιες ιδέες και προτάσεις, να δούμε μια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μας δίνει κάποιες προτάσεις, εμείς να κάνουμε και να δούμε πώς θα αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά. Το θέμα αυτό έχει μεγάλη σημασία και στην Ευρωβουλή μας. Κυρία Εισηγήτρια. Είμαι πρόθυμη να βοηθήσω όπως μπορώ και σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο που έχετε αναλάβει. Στη συνέχεια θα δώσω τον λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Merci, Madame. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι σας, σας ακούμε ε, στη γενική μας διεύθυνση. Δεν έχουμε έτοιμη λύση να σας προτείνουμε. Σας ακούμε, διαβουλευόμαστε. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2009 και θα εξετάσουμε στη συνέχεια τις ε, πολλές και διάφορες απαντήσεις που θα έχουμε πάρει. Κάναμε, είχαμε πολλοί αριθμές επαφές με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ε, με τις ε, τοπικές αρχές, ε, με τη βιομηχανία, με το κοινοβούλιο. Θα περιμένουμε να τοποθετηθεί το κοινοβούλιο σε αυτή την έκθεση πριν εισηγηθούμε οτιδήποτε. Η πρόταση που θα υποβάλουμε θα ακολουθήσει μία πλήρη μελέτη αντικτύπου όπου θα εξετάζουμε όλα αυτά τα ζητήματα που αναφέρατε, δηλαδή τις επιπτώσεις και τους κινδύνους μία τέτοια αναθεώρησης πολιτικής για την ε, ε, σταθερότητα και την ισορροπία όχι μόνο του τομέα αλλά και των παρακτήων περιοχών που εξαρτώνται από την ελευτική δραστηριότητα. Θα γίνει πλήρης μελέτη αντικτύπου λοιπόν. θα ε, εξετάσουμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο την ε, μεταρρύθμιση της αλλιευτικής πολιτικής. Ε, έχουμε ήδη επαφές με την συγγήτρια του Κοινοβουλίου, την κυρία Νεβές. Έχουμε κάνει ήδη ενδιαφέρουσες συζητήσεις, διεξοδικές συζητήσεις και θα τις συνεχίσουμε. Παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τι εξελίξεις για την εκδήλωση που διοργανώνει στο Πόρτο τον Νοέμβριο για το θέμα αυτό. Ε, ακούσαμε πληθώρα παρεμβάσεων που κάλυψαν όλα τα ζητήματα που αναφέρονται στην Πράσινη Βίβλο. Τονίστηκαν τα τρία-τέσσερα βασικά ζητήματα που προανέφερε και η συγγήτρια. Ε, λοιπόν συμφωνούμε απολύτως μαζί σας. Αυτά τα τρία-τέσσερα ζητήματα είναι στον πυρήνα της ελληνικής πολιτικής, όπως τόνισε και η Πρόεδρος, η κυρία Φράγκα. Πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτό το σκληρό πυρήνα της αλλιευτικής ε, πολιτικής ε, διατήρηση, υπερδυναμικότητα, υπεραλίευση, αλλιευτικές προσπάθειες. Είναι περίπλοκα, πολυσύνθετα αυτά τα προβλήματα, κυρίως όταν μιλάμε για την περιφερειοποίηση ή την αποκέντρωση ή όταν μιλάμε για τη σχετική σταθερότητα. Τα κράτη-μέλη στη συντριπτική τους πλειοψηφία, ξέρετε, υπεραμείνονται ε, ε, αυτής της αρχής της ε, σχετικής σταθερότητα. Το θέμα είναι να δούμε στην κοινή αλληλευτική πολιτική ορίζεται σωστά αυτή η αρχή. Αν χρησιμοποιηθούν οι ποσοστώσεις, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν και ατέλειες, διότι υπάρχουν ατέλειες ως προς την ανταλλαγή, ε, τη διακρατική ανταλλαγή των ποσοστώσεων. Δηλαδή δεν υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στον εθνικό στόλο και στις ποσοστώσεις πρόσβασης στους αλλιευτικούς πόρους. Ε, για πώς ε, λοιπόν να εξασφαλίσουμε αυτή την σχετική σταθερότητα χωρίς να καταργήσουμε την ισορροπία που επιθυμούμε στον τομέα αυτό. Ε, όσοι είπαν ότι πρέπει να μιλάμε μάλλον για αλλιευτικές προσπάθειες και όχι για ποσοστώσεις, είναι δύσκολο να μετρήσουμε ή να αξιολογήσουμε την ε, μετάβαση στο νέο σύστημα. Δηλαδή, τον ορισμό της πρόσβασης ε, στους αλλιευτικούς ε, πόρους και την έννοια της Ε, τις αλλιευτικής προσπάθειας. Ε, μην ξεχνάτε τις απορρίψεις που πρέπει να, στη θάλασσα που πρέπει να συνδυαστούν ε, με τις ποσοστώσεις. Οι απορρίψεις συνδέονται με τεχνικά μέτρα και η λύση για τις απορρίψεις κατά τη γνώμη μας, ε, πρέπει να γίνει μέσω της αναθεώρησης των τεχνικών ε, μέτρων. Ε, και δεν είναι αλήθεια ότι δεν έχει γίνει διαβούλευση του τομέα για το σχέδιο τεχνικών μέτρων που συζητείται αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο, γιατί κατηγορηθήκαμε και γι' αυτό. Πρόκειται για μία πρόταση που κάναμε τον ε, Ιούνιο το 2008 και όλα τα αράκτα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια απεφάνθησαν για αυτό το σχέδιο τεχνικών μέτρων. Έχει γίνει η διαβούλευση. Για αυτά για τη σχετική σταθερότητα υπάρχει και άλλο ένα πολύ σύνθετο πρόβλημα, όπως είπαμε, αυτό της αποκέντρωσης, περιφερειοποίησης. Τόνιζε η Πρόεδρος ότι θα πρέπει να γίνει ήδη διεξοδική νομική ανάλυση του ζητήματος. Λοιπόν, για πρώτη φορά η συνθήκη της Λισαβόνας αναφέρει ρητά την αποκλειστική αρμοδιότητα της ε, κοινότητας ε, για την ε, κοινή αλληλευτική πολιτική. Ξέρετε, ο, επίσης θα ενισχυθούν σε μεγάλο βαθμό οι αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου χάρη στη συναπόφαση. Τα αναφέρω αυτά γιατί όλοι είμαστε υπέρ μιας bottom προσέγγισης Βέβαια δεν θα αποφασίσουν μόνο τους τα περιφερειακά συμβούλια και θα ακολουθήσουν οι Βρυξέλλες. Αυτό ε, δεν συνάδει με την ε, συνθήκη ως νομικό καθεστώς. Ε, αντίθετα, δεν, μπορούν, δεν μπορούμε να λειτουργούμε βάσει των επιταγών των Βρυξελών. Και σίγουρα η στάση των περιφερειακών συμβουλίων είναι ευφιέστερη σε σχέση με αυτά που μπορούμε εμείς να φανταστούμε εδώ στις Βρυξέλλες και άρα ε, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ενισχύσουμε τη δυνατότητα του κλάδου να υποβάλει προτάσεις, ε, να συμμετέχει συζητήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ΜΚΟ, ε, σεβόμενοι όμως ε, τη συνθήκη της Λισαβόνας, ας μην την αφισβητούμε ενώ ακόμη δεν έχει τεθεί σε ισχύ. Το τρίτο εξαιρετικά ενδιαφέρον ζήτημα στο οποίο αναφερθήκατε είναι αυτό των αλλιευτικών δικαιωμάτων και την αρχή της μεταβασιμότητάς τους. Για, ε, μιλώντας για τη μεταβασιμότητα, έχετε κατά νου ότι γίνεται ανταλλαγή ανάμεσα στα κράτη-μέλη ανάμεσα σε κράτη που έχουν σταθερά δικαιώματα για πρόσβαση βάσει της σχετικής σταθερότητας. Και όταν ε, μιλάμε για ένα κατώτερο επίπεδο, δηλαδή εκτός από τη διακρατική μεταβίβαση δεν έχει καμία, κανένα νόημα η συζήτηση. Η μεταβιβασιμότητα είναι αντικείμενο διαπραγμάτευση σε ιδιωτικές αγορές. Ας μην περιορίσουμε τη συζήτηση μιλώντας αποκλειστικά για διακρατική ε, μεταβιβασιμότητα των ποσοστώσεων. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Η διαχείριση των αλλιευμάτων που θα βασίζεται σε αλλιευτικά δικαιώματα είναι θέμα που μέσα στην πράσινη βίβλο έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Γιατί βάσει ε, της εμπειρίας που έχουν κάποια κράτη-μέλη για αυτόν τον τρόπο διαχείρισης ε, των δικαιωμάτων προκύπτει σαφώς ε, ότι μειώνεται έτσι σε σημαντικό βαθμό η υπερδυναμικότητα. Βέβαια, η μείωση της υπερδυναμικότητας δεν οδηγεί αυτόματα σε μείωση της υπεραλίευσης. Πρέπει να κάνουμε διάκριση σαφή ανάμεσα σε αυτές τις δύο αρχές. Αυτό το θέμα όμως ε, έχει θεμελιώδη σημασία και είναι στην καρδιά της αλληλευτικής πολιτικής. Πρέπει να συνδυαστεί με τον ε, σεβασμό της αρχής της ε, σχετικής σταθερότητας, όπως επιθυμούν τα κράτη-μέλη. Εξετάζουμε διάφορους μηχανισμούς που θα μπορούσαν να το καταστήσουν δυνατό. Ε, η συγκέντρωση των αλλιευτικών δικαιωμάτων ε, στα χέρια κάποιων ε, αλλιευτικών επιχειρήσεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε αφαίρεση των σχετικών δικαιωμάτων από, τις, από τους μικρούς αλλιείς και άρα πρέπει να τους προστατεύσουμε δεν πρέπει να υπάρξει υπερβολική συγκέντρωση αυτών των ε, δικαιωμάτων για να προστατεύσουμε και τις ε, πολυάριθμες θέσεις απασχόλησης ε, του κλάδου και την κατάσταση των παρακτήων ζωνών που ζουν από αυτή τη δραστηριότητα. Εδώ για να κλείσω θα έλεγα ότι χρειάζεται και μια στρατηγική για την υδατοκαλλιέργεια που εγκρίθηκε πέρσι άλλα σημεία στη μερίσια διάταξη θα μας επιτρέψουν να το ξαναστήσουμε το θέμα. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ και για να ολοκληρώσουμε θα λάβει τον λόγο η συγγήτρια παρακαλώ. Το Σας ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να ξεκινήσω ακριβώς ευχαριστώντας για όλα τα σχόλια που έγιναν. Κατά τα άλλα ήδη, με την πρώτη αφορμή ανταλλαγών απόψεων, πήρα πολλές ε, τέτοιες παρατηρήσεις και σχόλια που με εμπλούτησαν και τώρα με διαφορετικό τρόπο διαπιστώνω ότι και αυτά τα σχόλια είναι πάλι ε, χρήσιμα πέρα από το επί της ουσίας, για να καταδείξουμε ότι εμείς εδώ στην Ευρωβουλή, στην Επιτροπή Αλληλείας έχουμε μπροστά μας μεγάλη σύγκληση απόψεων, μεγάλη συνένεση θα έλεγα απόψεων. Πράγμα το οποίο οδηγεί σε μια ενίσχυση της θέσης που θα υιοθετήσουμε και θα παρουσιάσουμε από πλευράς της Επιτροπής μας και ως Ευρωβουλή όσον αφορά την Πράσινη Βίβλο. Αληθεύει λοιπόν ότι ουσιαστικά το σύνολο των πτυχών που εδώ αναφέρθηκαν βρίσκονται ήδη κατά κάποιο τρόπο, ας το πω έτσι, αναφέρονται κατά κάποιο τρόπο στην έκθεσή μου. Από την άλλη πλευρά πάλι αληθεύει ότι τα όρια <clears throat> και οι περιορισμοί που υπάρχουν δεν δίνουν δυνατότητα για πολλά από αυτά τα θέματα να κάνουμε κάτι περισσότερο από το απλά και μόνο να τα επισημάνουμε ή να τα ανοιχνεύσουμε σε σχέση με την προώθηση, την επεξήγηση, την ε, ανάλυση που θα ήταν αναγκαία και που αυτό πάλι χρειάζεται και ελπίζω ότι θα έχουμε ευκαιρία να το κάνουμε αυτό σε μια υστερότερη χρονική στιγμή μεταγενέστερα. Όμως, από την άλλη πλευρά, δεν θα ήθελα να αμελήσω, να αγνοήσω, να υπογραμμίσω κάποιες από τις πτυχές που εδώ αναφέρθηκαν. Και έτσι, καθώς πραγματικά έχουν προτεραιότητα και μεγάλη σημασία, πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και επίσης για να καθησυχάσω κάποιους συναδέφους για θέματα για τα οποία μου επέστησαν την προσοχή μου. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω λέγοντας ότι έχει τεράστια σημασία η αλεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρθηκε αυτό σε σχέση με την παράκτη αλεία. Αλλά γενικά η αλεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι απλά και μόνο μια μεγάλη σημαντική πραγματικότητα υπό οικονομικό πρίσμα κοινωνικό πρίσμα μέσω της απασχόλησης έμεσης και άμεσης που διασφαλίζει, αλλά επίσης υπό το πρίσμα το ιστορικό, το πολιτισμικό και πολιτιστικό, τουριστικό επίσης. Δηλαδή, εμείς δεν μπορούμε να έχουμε μια προσέγγιση περιοριστική της αλίας, διότι πραγματικά αυτός ο τομέας αλίας έχει ζωτική σημασία σφαιρικά στην Ευρώπη για την ίδια την εικόνα που δίνει και πρέπει να λαμβάνεται. Και δεν πρέπει παρά να υπογραμμίσουμε αυτή τη σφαιρική σημαντική πτυχή. Διότι κατά τα άλλα επίσης ενισχύει. Ενισχύει το όραμα και την προσέγγιση που πρέπει να έχουμε για τις αλίες συνολικά, για την αλία σφαιρικά και τη σημασία της. Διατήρηση και διασφάλιση των αλλοιευμάτων των αποθεμάτων διασφάλιση της επαγγελματικής δραστηριότητας και της αποτελεσματικότητάς της. Είναι πτυχές που με κανένα τρόπο δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε. Πώς όλα αυτά όμως, όλες αυτές οι πτυχές θα ενταχθούν και θα είναι σεβαστές. Έγινε λόγος και ανέφεραν οι συνάδελφοι σχεδόν όλοι στην αποκέντρωση. Η αποκέντρωση τώρα είναι πραγματικά σημαντική και είναι μια αποκέντρωση που δεν θα πρέπει να προέρχεται, να, να βλέπει το στόχο μόνο, αλλά πρέπει να είναι παρούσα η αποκέντρωση σε όλη την αλυσίδα διαχείρισης του τομέα. Αναφέρθηκε επίσης εδώ ότι χρειαζόμαστε, πρέπει να καθησυχάσουμε κάπως τον τομέα των αλλιέων, διότι δεν είναι πολύ ικανοποιημένοι και ευχαριστημένοι με αυτό το οποίο προαναγγέλθηκε με τη μεταρρύθμιση και τα όσα έχουμε κάνει. Με αυτές τις αφορμές που είχα στο παρελθόν, παρέμβασης για την Πράσινη Βίβλο σε διάφορα φόρα, αυτό το οποίο είδα και η εντύπωση που αποκόμισα ήταν ότι μετά τη συζήτηση που γίνεται καθησυχάζουν περισσότερο οι άνθρωποι. Όταν γίνεται λόγος για την ανάγκη αποκέντρωσης, για παράδειγμα, στο επίπεδο λήψης αποφάσεων είναι σημαντική αυτή η αποκέντρωση για μια πολιτική υπεύθυνη λήψη αποφάσεων που θα μειώνει τι απώλειες και τη διασπάθηση πόρων για μια καλύτερη βέλτιστη παρέμβαση στην αλία και την ίδια την εμπορία, την αξιολόγηση και αναβάθμιση του αλιεύματο και των ηχθείων. Πρέπει λιγότερο να ε, αλλιεύουμε, αλλά με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Να μην υπεραλλιεύουμε, αλλά να είμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί και για την αηφορία των αποθεμάτων και τη διατήρησή τους και είναι επίσης ε, απαραίτητο και την διασφάλιση της ευημερία του τομέα αυτού και για την διασφάλιση των εισοδημάτων των ανθρώπων που ασχολούνται με την αλληλεία. Τα άτομα δηλαδή που ασχολούνται με αυτό το επάγγελμα. Δεν θα ήθελα να χάσω εδώ την ευκαιρία να πω ότι πέρασα το προηγούμενο Σάββατο σε μια συνάντηση στην ε, Σίνες, μια περιοχή αλλιέων στην Πορτογαλία, μιλώντας για την Πράσινη Βίβλο. Και ήταν μια συνάντηση που διοργανώθηκε από τις γυναίκες ακριβώς, Ψα... Ε, γυναίκες που ψαρεύουν, γυναίκες ε, αλλιείς. Ιδιαίτερα λοιπόν είμαι ευαίσθητη σε σχέση με αυτά τα θέματα, λαμβάνοντας υπόψη και την ίδια μου την παρουσία, αυτό το βίωμα που είχα και την συμμετοχή στις συζητήσεις. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή αυτές οι πτυχές που προαναφέρθηκαν μόνο σε αυτές θα πρέπει να μείνουμε. Πρέπει να πω επίσης ότι σε μεγάλο βαθμό όλοι συμφωνούμε για όλα αυτά και θα ολοκλήρωνα αναφέροντας ε, ακόμα την πτυχή που θεωρώ ότι είναι ουσιώδης και θεμελιώδης και πρέπει να ληφθεί υπόψη σε αυτή την έκθεση και να τονιστεί. Μια σφαιρική προσέγγιση και αντιμετώπιση του τομέα της αλίας σφαιρικά συμπεριλαμβάνοντας όλους τους παράγοντες και πτυχές που συμμετέχουν και που είναι αποφασιστική σημασία για την αηφορία της αλληλεία στο μέλλον, κατανοώντας ότι δεν πρέπει να υπάρξει μία, ας το πω έτσι, απλά και μόνο ιεραρχημένη προσέγγιση, αλλά θα πρέπει απλά να λάβουμε όλους τους παράγοντες υπόψη στη διασύνδεσή τους και στη διάρθρωσή τους. Απομένει ακόμα να πω ότι στον χρόνο που ακόμα έχουμε για να δουλέψουμε για αυτά τα θέματα μπροστά μας θα είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για όλα τα σχόλια και τις προτάσεις που θα μου υποβάλλετε και θα τα μελετήσω προσεκτικά για να προσπαθήσω να τα λάβω υπόψη όλα αυτά, ιδιαίτερα από πλευρά των σκιωδών εισηγητών, ώστε να καταλήξω σε μια έκθεση αρκετά δυνατή και αποτελεσματική και έτσι να μπορέσουμε να ασκήσουμε πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να έχουμε με αυτόν τον τρόπο κάποιο λόγο να πούμε κι εμείς ως Ευρωβουλή για αυτόν τον τομέα, επομιζόμενοι των ευθυνών μας και επομιζόμενοι των αρμοδιοτήτων που έχουμε για να μπορέσουμε να διευρύνουμε αυτό το πλαίσιο και να μπορέσουμε να καλύψουμε όλες τις ευθύνες αυτές που έχουμε έναντι των ψηφοφόρων μας και έναντι όλων εκείνων που εργάζονται στην Αλία. Πρέπει να πούμε και να αρθρώσουμε ένα λόγο υποστήριξης και λύσεις που πρέπει να τους δώσουμε για τη δραστηριότητά τους στο μέλλον. Πρόεδρος, ευχαριστώ κυρία εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ και εσάς κύριε για τις επεξηγήσεις που μας δώσατε από την Επιτροπή που ήταν σαφής. Και απλά θα ήθελα να σας πω τώρα στη συνέχεια ότι η επόμενη συζήτηση θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου όταν η κυρία εισηγήτρια θα έχει ήδη συντάξει, θα, ε, θα παρουσιάσει την έκθεση από πλευρά τη. Και έτσι λοιπόν θα έχουμε συγκεκριμένο κείμενο για Ολοκληρώνοντα αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη, περνάμε στο επόμενο σημείο, που είναι η παρουσίαση των μελετών σε σχέση με την υδατοκαλλιέργεια. Όπω γνωρίζετε, τρει μελέτε είπαμε ότι έπρεπε να συνταχθούν. Έχουμε σήμερα να, την ευκαιρία να ακούσουμε του συντάκτε των εκθέσεων. Πρώτον, αξιολόγηση των επιπτώσεων τη στρατηγική για την αηφορία στην υδατοκαλλιέργεια. Ολοκληρώθηκε και θα το δείτε στα αγγλικά, στην τεκμηρίωση που διανεμήθηκε σήμερα και οι μεταφράσει αυτή τη μελέτη μελέτης καθώς επίσης και των άλλων μελετών για τις ε, διαρθρώσεις και τις διατάξεις ε, για την ε, υδατοκαλλιέργεια στην Ευρώπη και την ανταγωνιστικότητα θα διανεμηθούν υστερότερα στο μέλλον. Δίνω τον λόγο στον κύριο Λέιν για να μας κάνει την παρουσίαση ακριβώς για τη μελέτη της αξιολόγησης επιπτώσεων για τη στρατηγική για την αηφόρο ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ιδατοκαλλιέργειας. Για 15 λεπτά το πολύ έχετε τον λόγο, εντάξει, έχετε τον λόγο, παρακαλώ.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 Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας κάνω την παρουσίαση αυτή ε, για την υδατοκαλλιέργεια. Έχετε την πλήρη μελέτη στα αγγλικά. Αφορά την αξιολόγηση της ε, στρατηγικής του 2002 για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας που είχε τρεις στόχους ε, αναφέρονται εδώ. Ο πρώτος ήταν η αύξηση του, της απασχόλησης από 8.000 ε, έως 10.000 2003 ε, έως 2008. Το δεύτερο ήταν η εξασφάλιση προϊόντων ε, υγιεινών, ασφαλών και καλής ποιότητας και επίσης η ανάπτυξη ενός κλάδου περιβαλλοντικός κατάλληλου. Αυτό που επίσης πρέπει να πω είναι ότι μόνο ο πρώτος στόχος και ο τέταρτος υποστόχος μπορούν να ε, ποσοτικοποιηθούν στην αξιολόγηση. Επίσης είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι κατά τη στρατηγική του 2002 ήταν η πρώτη φορά που υπήρξε μια ειδική στρατηγική για την υδατοκαλλιέργεια ε, παρά το γεγονός ότι γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ε, χρόνια υπάρχει η υδατοκαλλιέργεια στην, Ευρωπαϊκή, στην Ευρώπη Ευρώπη και ήταν η πρώτη φορά που υπήρχε στρατηγική για το θέμα αυτό. Λοιπόν, θα αναφερθώ πρώτα σε μία έρευνα ενδιαφερομένων φορέων που έγινε, επίσης σε μία ανάλυση των ε, ε, διαφόρων ε, κενών που υπάρχουν και επίσης το τρίτο μέρος θα είναι κάποιες συστάσεις. Προσπαθούμε λοιπόν να αξιολογήσουμε την επιτυχία, όπως επίσης και την εφαρμογή των μέτρων υποστήριξης της στρατηγικής ε, και ε, θα δώσουμε και τη δυνατότητα σχολείων ε, και απόδοσης για παράδειγμα λόγων για τους οποίους ήταν ανεπιτυχή σε μερικούς τομείς ευρωπαϊκές οργανώσεις, εθνικές οργανώσεις παραγωγών, ε, ηγέτες του κλάδου, ε, συντονιστές ε, θεμάτων RTD, όπως επίσης και οργανώσεις καταναλωτών στα κράτη-μέλη, μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Όλοι αυτοί ήταν οι εμπλεκόμενοι φορείς. Δεν θέλαμε μόνο να ακούσουμε εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη, αλλά θα θέλαμε και την άποψη εκείνων που γνωρίζουν λιγότερα για τις υδατοκαλλιέργειες θα δείτε ότι το ίμιση των ερωτηθέντων προέρχονταν από τον κλάδο, ένα τρίτο από τον επιστημονικό ε, τομέα, από τους επιστήμονες και το ένα τρίτο από τους καταναλωτές μη κυβερνητικής οργανώσεις και κυβερνητικούς φορείς. Θα ήθελα επίσης να πω ότι η έρευνα ήταν λιγότερο ευνοϊκή ε, και η συμμετοχή συνεπώ ήταν και λιγότερο ε, σημαντική από πλευράς των χωρών όπου η δατεκολιέργεια έχει μικρότερη σημασία και αυτό ήταν πραγματικά κρίμα. Σε γενικέ γραμμές πρέπει να πούμε ότι 57% ε, ήταν οι απαντήσει στις ερωτήσει μας και πιστεύουμε ότι είναι αρκετά καλό ποσοστό. Να σα πω ορισμένα πράγματα τώρα για, τους, για τα μέτρα υποστήριξη. Θα δείτε τι πιο σημαντικέ και πιο επιτυχημένες συνεχής δράσης. Ε, βλέπετε ε, και τα ποσοστά ανά ε, στόχο και τα ποσοστά ανά ενδιαφερόμενους φορείς. Σας δίνω λίγο το χρόνο να τα διαβάσετε και μετά πηγαίνω στις λιγότερο επιτυχείς δράσεις. Βλέπετε και πάλι τα ποσοστά, τα αντίστοιχα ποσοστά. Βλέπετε και τους βασικούς στόχους. Οι επόμενες δύο διαφάνειες αφορούν τα συμπεράσματα όσον αφορά το πώς αντιλαμβάνονται τις ε, την επιτυχία αυτή ε, όλους τους τομείς που είχαν να κάνουν με την ε, ασφάλεια και το περιβάλλον, την ευημερία και την κατανάλωση και την μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου. Αυτά ήταν, ήταν ιδιαίτερα κατανοητά ως στόχοι. Ε, επίσης επιτυχή ήταν τα ζητήματα που αφορούσαν τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων φορέων, τα, τα θέματα των ηχθειοτροφών, τις ε, δυνατότητες χρηματοδότησης RTD, όπως επίσης και τον εντοπισμό των προτεραιοτήτων των, ε, ε, της έρευνας. Αυτά θεωρήθηκαν οι σημαντικότερες επιτυχίες. Όσον αφορά τώρα τις αποτυχίες, ήταν σαφές ότι η αύξηση, ο στόχος της αύξησης της απασχόλησης δεν επετεύχθη, ούτε επίσης, ούτε ο στόχος της αύξησης της παραγωγής και επίσης δεν μπορέσαμε να επιλύσουμε ζητήματα χωροταξικά ή ζητήματα ανάπτυξης της αγοράς. Επίσης, ανεπιτυχή ήταν, οι προσπάθειες ε, για την βιολογική και περιβαλλοντικώς φιλική υδατοκαλλιέργεια, όπως επίσης και την ενσωμάτωση της ε, υδατοκαλλιέργειας ε, μέσω ζωνών στρατηγικής. Θα ήθελα να σας αναφέρω και ορισμένα αριθμητικά στοιχεία όσον αφορά τις εκτιμήσεις από το 1997 μέχρι το 2006 σε θέματα απασχόλησης. Βλέπατε ότι δεν καταφέραμε να αυξήσουμε σημαντικά την απασχόληση σε πέντε έτη. Ε, αυτό το γράφουμε εδώ σας δείχνει την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 αύξηση της παραγωγής κατά 0,5% για την περίοδο 2001-2008 σε σχέση με, με 7,6% για τις ε, μη ε, μέλη, για τις ε, χώρες Ευρώπης που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βλέπετε επίσης και, ένα, και, και σύνολα χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευρωπαϊκών χωρών που δεν είναι μέλη. Βλέπετε τις διαφορές και πώς έχουν τα πράγματα ε, και σε παγκόσμιο επίπεδο και θα ήθελα να σας πω και πώς αντιλήφθηκαν όλη αυτή την αξιολόγηση όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς. Ε, αυτή ήταν η βάση της ανάλυσής μας. Επίσης, ε, τα ζητήματα των πρωτοβουλειών για την αγορά και τον κλάδο, όπως για παράδειγμα την πλατφόρμα τεχνολογίας και γεωμαϊκής ε, και Επίσης ε, υπήρξε και ένα σύστημα σηματοδότησης ε, για την αξιολόγηση των σημαντικότερων κενών. Ε, η αντικειμενική μας αναθεώρηση ήταν μάλλον πιο απεσιόδοξη από αυτή που είχαν οι ενδιαφερόμενοι φορείς όσον αφορά τώρα τους στόχους και τα σχετικά συμπεράσματα, υπήρχαν και οι επιμέρους στόχοι των, της ε, αύξησης της παραγωγής και της πρόθεσης της αγοράς, που αντιλήφθηκαν με διαφορετικό τρόπο οι ενδιαφερόμενοι ε, φορείς. Ε, και υπήρχαν και συνοδευτικές δράσεις υποστήριξη, όπως για παράδειγμα η αύξηση των ε, ε, μονάδων ποιότητας, οι εκστρατείε προώθησης, ε, και δεν υπήρχαν ιδιαίτερα μεγάλες διαφορές όσον αφορά τον ε, στόχο 2, την ε, εξασφάλιση της ποιότητας για τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Υπήρχαν όμως διαφορές στον τρίτο στόχο για τις τέσσερις συνοδευτικές δράσεις, τη διαχείριση των άγριων ηχθείων, τα κριτήρια και τις κατευθυντήριες γραμμές, όπως επίσης και την προστασία των ε, άγριων ειδών. Και θα ήθελα να φτάσω στο τελευταίο τμήμα που έχει να κάνει με τις συστάσεις. Το 2007 ε, υπήρξε διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τους ενδιαφερόμενους φορείς για την ανάπτυξη της ε, ανακοίνωσης του 2009. Δεν θα σας αναφέρω όλες τις συστάσεις, μπορεί να τις δείτε και στην έκθεση, αλλά θα επικεντρωθώ σε μερικές. Η πρώτη μας πρόκληση είναι η βελτίωση της εικόνας της ε, τομέα της υδατοκαλλιέργειας. Ε, το, η στρατηγική του 2002 αύξησε το πώς γινόταν κατανοητή η συμμετοχή των ενδιαφερομένων φορέων και αυτό είναι κάτι που μας δίνει τη δυνατότητα βελτίωσης τη εικόνα. Αυτή η βελτίωση συνάδει με τη σύσταση του Συμβουλίου για την προώθηση της υδατοκαλλιέργεια, αλλά θα δείτε ότι υπάρχουν κάποια επιμέρους σημεία που πηγαίνουν πέρα από την, από την ε, παραγωγή των τροφίμων στο πλαίσιο του τομέα, αλλά α πούμε μιλάει για την ε, για τα αποθέματα ε, και την ε, διατήρηση των ε, απειλουμένων ειδών, της, την αξιολόγηση των, του ωφέλους των νέων και παραδοσιακών πρακτικών υδατοκαλλιέργειας στις παράκτιες ζώνες. Ολόκληρη λοιπόν η, η εικόνα της ε, υδατοκαλλιέργειας πρέπει να βελτιωθεί. Δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει αυτό μέσω νομοθεσίας ε, ε, ή σύστασης. Είναι ζήτημα επικοινωνίας κατά κάποιο τρόπο. Επίσης, ε, θελήσαμε να υπάρξει ένα παρατηρητήριο για την ε, επαρκή παρακολούθηση της, υδατοκαλλιέργειας, ε, ένα σύστημα των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας σε ολόκληρη τη διατροφική αλυσίδα. Υπήρξαν πάρα πολλά σενάρια για την συλλογή των δεδομένων και μάλιστα προκηρύχθηκε και ένας διαγωνισμός για το πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα τέτοιου είδους παρατηρητήριο στο πλαίσιο της υδατοκαλλιέργειας για να βοηθηθεί ο τομέα, όχι μόνο να προγραμματίζει την παραγωγή του, αλλά να μπορέσει να αντιμετωπίσει τιμές, ε, κρίση τιμών που υπήρχαν για παράδειγμα στον, ε, στην λεκάνη της Μεσογείου τα τελευταία 10 χρόνια. Όσον αφορά το περιβαλλοντικό σφυλικό της υδατοκαλλιέργεια, πολύ γρήγορα πηγαίνουν τα πράγματα θα υπάρξει ένα σύστημα πιστοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την περιβαλλοντικό φιλική ε, υδατοκαλλιέργεια που πρέπει να συμπεριλάβει ε, ενημερωτικές εκστρατείες ε, για την προώθηση της αποδοχής των προϊόντων με οικολογικές ετικέτες. Επίσης να επιτραπούν διακρατικά προγράμματα προώθησης που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, όπως επίσης και η ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο του διαλόγου για την υδατοκαλλιέργεια και την ύπαρξη ενός ε, συμβουλίου για την καθοδήγηση της υδατοκαλλιέργειας που θα αρχίσει να ε, λειτουργεί από το 2011 και υπάρχουν και άλλες παγκόσμιες ε, ε πρωτοβουλίες ε, ε, και επομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μείνει πίσω, γιατί υπάρχουν και πολλέ ενδιαφέρουσε ε, πρωτοβουλίε σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτά είναι τα τομεακά ζητήματα. Το να περάσουμε σε δύο συγκεκριμένε συστάσει, ε, όπου υπάρχουν νομοθετικέ δυνατότητε, ε, είναι απολύτω απαραίτητο να είμαστε πολύ πιο συγκεκριμένοι στην ερμηνεία και στην εφαρμογή τη μελέτη αξιολόγηση αντικτύπου. Πρέπει να επιτύχουμε την διευκόλυνση των διαδικασιών αδειοδότηση, όπω επίση και τη βελτίωση ολοκλήρωση ε, ε ε, μέσων πληροφορικής που έχουμε. Να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να παρουσιάσουν τις κατευθυντήριες γραμμές και να τα συζητήσουν, όπως επίσης και μελέτες ανάλυσης περιπτώσεων που ε, καταδεικνύουν αποτελεσματική και ταχύη εφαρμογή της ευρωπαϊκής και της εθνικής νομοθεσίας. Είναι κάτι που μπορεί να γίνει πάρα πολύ άμεσα. Είναι πολύ καλές αποφάσεις που μπορούν να, γίνουν πολύ, να ληφθούν πολύ γρήγορα όσον αφορά τη χορήγηση αλλά και τη μεταβίβαση των αδειών ε, για τη χρήση της υδατοκαλλιέργειας. Και το τρίτο θέμα αφορά την εκτροφή Τα, τους άγριους ηχθείες, ε, δεν θα πω σε πολλές λεπτομέρειες, γιατί θα χρειαζόμουν πολύ περισσότερο χρόνο για να το κάνω αυτό. Όσον αφορά λοιπόν τα άγρια είδη και την θύρευσή τους ε, στην Ευρώπη, θα ζητούσαμε τα κράτη-μέλη να εγκρίνουν ε, την ε, νόμη την, ε, την ε, εφαρμογή της ε, σχετικής της νομοθεσίας και της σχετικής ορολογίας που έχουν να κάνουν με τα άγρια πτηνά και τα οικοσυστήματά τους, όπως επίσης και χρειαζόμαστε ένα συντονισμένο πρόγραμμα διαχείρισης των πληθυσμών, και αποτελεσματική εφαρμογή του. Και το τελευταίο τμήμα για τις τεχνολογίες, θα θέλαμε μία ανάλυση του τομέα για την για, τα συστήματα των υδατοκαλλιεργειών, ε, ε, τα χερσαία και όσον αφορά την offshore υδατοκαλλιέργεια θέλουμε να δούμε αξιολόγηση των τεχνικών εξελίξεων που δίνουν τη δυνατότητα λειτουργίας των συστημάτων, όπως επίσης και τη σωστή εφαρμογή τους, την επιτυχή εφαρμογή τους, ε, για παράδειγμα κατευθυντήριες γραμμές, εντός μηχανισμών χωροταξικής χωροτοξικού σχεδιασμού. Όσον αφορά τα συστήματα ε, της υδατοκαλλιέργειας, ε, δεν είναι η βασική πρακτική, ε, γιατί στις παράκτιες ε, ζώνες γίνεται συνήθως η υδατοκαλλιέργεια αλλά πρέπει να δούμε τι αποτέλεσμα έχει αυτό σε περιβαλλοντικό επίπεδο. Η υδατοκαλλιέργεια πρέπει να έχει πολύ πιο σαφή θέση στο χάρτη πορείας ε, για, τον, ε, για τη χωροτεξικό σχεδιασμό, ε, γιατί είναι σημαντικός παράγων και πρέπει να θεωρηθεί βασική ευρωπαϊκή στρατηγική. Ενδεχομένως να είναι το μεγαλύτερο η μεγαλύτερη διαφορά στον αντίκτυπο και στην αξιολόγησή του. Δεν αναφέρεται η σχέση του με, τις, ε, με τη θαλάσσια πολιτική, με άλλες πολιτικές που επηρεάζουν την ε, εφαρμογή της. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή. Ευχαριστώ πολύ. Λέει Πρόεδρος. Αν δεν θέλει ο κύριος Μιλάνα να πάρει το λόγο αμέσως, να περάσουμε στην επόμενη παρουσίαση. Εκτός αν θέλετε να πάρει το λόγο αμέσως. No, no, yeah, yeah. Έλεγα ότι αν θέλετε να κάνετε μια ερώτηση, να την... μπορείτε να την κάνετε τώρα. Ναι, ναι έχω κάποιες παρατηρήσεις. Διότι ε, υπάρχει μια θετική αξιολόγηση ε, και μιλάτε για επικοινωνιακή πολιτική, αλλά σε σχέση με ποιους, ε, γιατί υπάρχουν ε, και προβλήματα στα οποία δεν αναφερθήκατε. Τα συστήματα διοδοτήσεων, οι εκθέσεις ανάμεσα στις χώρες, η επίπτωση των υποδομών υδατοκαλλιέργειας που ήδη υπάρχουν, Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Γιατί αποκλείεται ήδη εξ αρχής την offshore υδατοκαλλιέργεια. Μπορείτε να μου εξηγήσετε. Ευχαριστούμε. Έχετε το λόγο. Ε, μιλώντας για τις ε, διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη και την ανάγκη επικοινωνίας που υπάρχει, θα έλεγα ότι αυτοί που εκπονούν τις πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους γενικότερα στο παρελθόν δεν είχαν επίγνωση της σημασίας της υδατοκαλλιέργειας αυτή που εκπονούσαν τις πολιτικές στον, ε, στη βιομηχανία των τροφίμων. Στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καλούνται τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν ε, μέτρα στον τομέα αυτό και αυτό είναι σημαντικό κατά τη γνώμη μας, διότι τα κράτη-μέλη θέλουν να εφαρμόσουν μία πολιτική που όμως συγκρίνουν με την εθνική τους πολιτική. Το θέμα της ε, offshore υδατοκαλλιέργειας ε, πώς έχει. Η τωρινή κατάσταση στην αγορά μας δείχνει ότι τα κράτη-μέλη δεν θεωρούν καν ότι υπάρχει σχετική στρατηγική. Υπάρχουν περιορισμοί για τη διενέργεια υδατοκαλλιέργειας offshore, μακριά από τις ακτές. Και κάποια κράτη-μέλη όμως ε, τελευταία ανακοίνωσαν σημαντικότατες ε, επενδύσεις στις τεχνολογίες ε, του τομέα. Δεν μιλάμε για την ανοιχτή θάλασσα, μιλάμε για τεχνολογίες υψηλότερες, για τεχνολογίες όπου χρησιμοποιούνται τα κύματα ή άλλες μορφές ενέργειας και δεν περιοριζόμαστε στην παράκτεια υδατοκαλλιέργεια. Είναι μεγάλη σημασία στη στρατηγική για κάποια κράτη όπου δεν υπάρχει λόγω γεωγραφικής θέσης πρόσβαση σε πιο προστατευμένες εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Χάτλικ, ο οποίος θα μας παρουσιάσει την έκθεση του για τις νομικές προϋποθέσεις διατοκαλλιέργειας. Έχετε 15 λεπτά στη διάθεσή σας για αυτή την παρουσίαση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα παρουσιάσω την έκθεση για τους νομικούς ε, και ρυθμιστικούς ε, περιορισμούς που προετοίμασα σε συνεργασία με ένα δίκτυο εθνικών ε, εμπειρογνωμόνων και από τρίτες χώρες και υπό τη χορηγία του Ocean Law και Poseidon ARM. Ο στόχος της έκθεσης ήταν να εξετάσουμε το ρόλο των νομοθετικών ρυθμίσεων ε, στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η βιομηχανία, κυρίως όπως μόλις εξήγησε ο Άλιστερ, ε, μιλώντας για ε, την απουσία ουσιαστικά της πολιτικής για την υδατοκαλλιέργεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα έπρεπε να πούμε κάποια πράγματα για τον ρόλο των ε, ρυθμιστικών ε, διατάξεων σε αυτό το τομέα. Φυσικά είναι ένας μόνο από τους παράγοντες που εξηγούν την έλλειψη ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας. Ο ρόλος είναι περίπλοκος, ο ρόλος των ρυθμιστικών διατάξεων γιατί δεν είναι κακό να έχουμε ρυθμιστικές ε, διατάξεις, ε, αλλά ίσως δεν είναι και καλύτερη προσέγγιση για να λύσουμε κάποια προβλήματα. Λοιπόν, βάσει αυτής της έκθεσης, λάβαμε υπόψη τις σύγχρονες αρχές της ε, καλύτερης νομοθεσίας. Για κάθε πρόβλημα αναρωτηθήκαμε αν χρειάζεται κανονιστική ρύθμιση, τι είδους κανονιστική ρύθμιση χρειάζεται και σε ποιο βαθμό και ή αν υπάρχουν αλλακτικές λύσεις. Ε, για τους εθελοντικούς κώδικες, που μπορεί να χρησιμοποιήσει η βιομηχανία. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο αξιολογήσαμε τους νομοθετικούς περιορισμούς ε, ε, εξετάζοντας το θέμα σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο τρίτων χωρών και επιζητώντας ευέλτιστες πρακτικές που μπορούν να λειτουργήσουν ως υποδείγματα. Για να σας πω εν γέννη ποια είναι τα προβλήματα, θα άρχιζα από το ότι ο κανονισμός υδατοκαλλιέργειας είναι εξαιρετικά περίπλοκος. Δεν υπάρχει η πολιτική για την υδατοκαλλιέργεια σε δέκα τουλάχιστον τομείς. Υπάρχουν διάφορες οδηγίες που καλύπτουν τις επιπτώσεις της πολιτικής και έχουμε φυσικά τη στρατηγική του 2002 που αναθεωρήθηκε το 2009. Αυτό είναι το βασικό νομοθετικό ε, πλαίσιο. Ε, τώρα, Υπάρχουν διαφορέ ω προ την εφαρμογή των ε, ρυθμίσεων στα κράτη-μέλη. Τα γενικότερα προβλήματα μεταφορά στην εθνική νομοθεσία παρατηρούνται σε όλου του τομεί. Δεν μα απασχόλησαν σε μεγάλο βαθμό, αλλά υπάρχουν και ειδικά ε, προβλήματα εφαρμογής των νομοθετημάτων ειδικών για την υδατοκαλλιέργεια. Αυτά φυσικά τα μελετήσαμε. Ε, σύντομα θα ήθελα να απαριθμίσω τα βασικά προβλήματα που εντοπίσαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει πρόβλημα με το καθεστώς και τον τρόπο λειτουργίας του καθεστώτος αδειοδότησης. Ε, συνδέσαμε αυτό το πρόβλημα με όσα συμβαίνουν σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, λίγες ρυθμίσεις υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον έλεγχο το, της αδειοδότησης και τον μηχανισμό αδειοδότησης ε, που διέπεται μάλλον από εθνικές ρυθμίσεις. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη και στο ιστορικό των κρατών μέλων υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Θα επανέλθω σε αυτό. Σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχει μεγάλη αυτονομία σε κάποιες περιφέρειες. Τι σημαίνει αυτό, ότι σε κεντρικό επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχει πολιτική για την αδειοδότηση και μπορεί να προκύψουν διαφορές, σας είπα, και σε επίπεδο κρατών μελών. Άλλο πρόβλημα τώρα, πρόσβαση στους τόπους ε, αυτό εκδηλώνεται περισσότερο σε εθνικό επίπεδο. Δύο πτυχές είναι σημαντικές. Ε, ο χωροταξικός προγραμματισμός, αυτό κυρίως σε θαλάσσιες ε, περιοχές. Ορισμένες φορές ε, βέβαια σημειώνεται πρόοδος ε, λόγω της θαλάσσια πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η IA τώρα, αυτό ο τομέας δεν ρυθμίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ω προ την εφαρμογή της νομοθεσίας υπάρχουν κάποια προβλήματα, αν εφαρμόζονται ομοιόμορφα δηλαδή σε όλα τα κράτη-μέλη. Προς το παρόν, μιλώντας για την κοινοτική νομοθεσία, ε, συνιστά πρόβλημα η εφαρμογή της πολιτικής γιατί μπορεί να επηρεάσει την ιδέα καλλιέργεια, η σχετική νομοθετική ρύθμιση και μία από τις βασικότερες ε, ανησυχίες ε, είναι το θέμα των ε, προστατευόμενων ειδών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ήδη που προστατεύονται βάσει της σχετικής οδηγίας για τα αποθέματα τους για τους, ε, τις οδηγίες δηλαδή για τους βιοτόπους. Υπάρχουν όμως και ειδικά νομοθετήματα που διαπιστώσαμε ότι δεν καλύπταν πλήρως τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Τα, σε επίπεδο κράτων μελών, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι από τις χώρες που αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα. Δεν θα επεκταθώ. Απλά ήθελα να αναφέρω το ότι υπάρχουν κοινά προβλήματα, κυρίως ως προς τις άδειες και την πρόσβαση στους ε, χώρους υδατοκαλλιέργειας. Υπάρχουν ειδικά προβλήματα σε κάποια κράτη-μέλη, τα οποία σε μεγάλο βαθμό προκύπτουν από το ότι υπάρχουν ε, διάφοροι οργανισμοί και εφαρμόζονται πολλά και διαφορετικά καθεστώτα στα κράτη-μέλη. Έλλειψη εναρμόνισης ε, της πολιτικής, διάφορες οργανώσεις αρμόδιες για τον τομέα. Επίσης δεν προσδιορίζονται επαρκώ. οι χώροι υδατοκαλλιέργειας όταν γίνεται χωροταξικό σχεδιασμός. Εν συντομία θα έλεγα ότι εξετάσαμε λίγο και την κατάσταση στις τρίτες χώρες και προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε βέλτιστες πρακτικές. Νορβηγία, ε, Χιλή και άλλες ε, χώρες Ε, τα αριθμιστικά συστήματα και τα προβλήματα που υπάρχουν ε, στον οικονομικό και στον κοινωνικό τομέα διαφέρουν από κράτος ε, σε κράτος και μια λύση που λειτουργεί σε ένα κράτος μέσα δεν σημαίνει ότι αυτόματα θα λειτουργήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην Νορβηγία ε, είδαμε ότι υπάρχουν πολλές θετικές πτυχές. Ε, μία από αυτές είναι η εξής. Υπάρχει το 2005 πέρασε ένα πλήρες νομοσχέδιο για την γεωργική και αλλιευτική πολιτική και υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή στον τομέα. Ε, υπάρχει το σύστημα διοδότησης ενιαία στηρίδα, single window, ένα λεπτάκι να βρω και τη σωστή διαφάνεια. Πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα. Ο ετών υποβάλλει την αίτηση σε έναν οργανισμό υπεύθυνο για την αλία το, τη διεύθυνση Αλείας και η διεύθυνση Αλείας έρχεται σε επαφή με όλους τους ε, υπόλοιπους φορείς. Δηλαδή ο ετών ε, έχει επαφή μόνο με έναν οργανισμό. Όταν η διεύθυνση Αλείας έρχεται σε επαφή με τους συναρμόδιους φορείς ακολουθούνται συγκεκριμένες διαδικασίες και προθεσμίες και λειτουργεί εσύ το σύστημα. Ένα άλλο θέμα είναι ότι υπάρχουν ειδικοί όροι για την υδατοκαλλιέργεια στην περιβαλλοντική νομοθεσία και αυτό έχει σημαντικό ρόλο και στην EIA. Κάτι άλλο εποφελές είναι η υποθήκη των αδειών, η δυνατότητα ενυπόθηκων αδειών. Και αυτό το σύστημα ε, λειτουργεί καλά. Στην Χιλή υπάρχουν κάποια προβλήματα λόγω νόσων έγινε μια νομοθετική μεταρρύθμιση. Εκεί δεν έχουμε τόσο πολλά παραδείγματα να αναφέρουμε, απλά ήθελα να επισημάνω ότι και αυτοί ακολουθούν αυτό το σύστημα της ενιαίας θηρίδας, του single window. Άλλες χώρες έχουν παρεμφερεί προβλήματα ως προς τις νομοθετικές διατάξεις βέβαια σας είπα ότι με το σύστημα του ενιαίου, της ενιαίας θηρίδας λύνονται κάποια από αυτά τα προβλήματα. Είδαμε την κατάσταση και στην Αυστραλία όπου υπάρχει ένας γενικός κώδικας, μια γενική νομοθεσία, ε, ένα γενικό ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο. Μία από τις λύσεις, αναφέρω εν παρόδο, ότι υπάρχουν και διάφοροι περιορισμοί για την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί είστε ζήτημα αρμοδιότητας για κάποια προβλήματα, δηλαδή κάποια θέματα είναι αμυγός εθνικής ορμοδιότητας, χορταξικός σχεδιασμός παραδείγματος χάρη, Υπάρχει το θέμα που προβλέπεται από τη συνθήκη ότι μπορούν τα κράτη-μέλη να προβλέψουν αυστηρότερα περιβαλλοντικά μέτρα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ρόλος της αρχής επικουρικότητας, όλα αυτά θα πρέπει να συνυπολογιστούν ε, όταν εξετάζουμε το τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα. Ε, τώρα δεν ξέρω αν είναι το θέμα της έκθεσης, ε, αλλά ε, μιλώντας για μια κοινή θαλάσσια και αλλιευτική πολιτική, και γιατί λέω ότι είναι εκτός θέματος, ελαφρώς, διότι η καλλιέργεια είναι ένα μόνο θέμα αυτής της πολιτικής. Πάντως, ο Κλάδο ε, δεν ασχολείται με αυτό το θέμα τώρα. Όπως σα εξήγησα, υπάρχουν περιορισμοί που οφείλονται στο ότι πολλά ζητήματα είναι εθνικής και όχι κοινοτική αρμοδιότητα, οπότε εξετάζουν άλλες λύσεις στη βιομηχανία. Στην πράξη τι μπορούμε να κάνουμε Τρει ε, προσεγγίσει ε, προέκυψαν εν μέρη νομοθετική μεταρρύθμιση εισαγωγή ενός συγκεκριμένου κανονισμού ή μια συγκεκριμένη ειδική οδηγία, δεύτερη προσέγγιση, στοχευμένη νομοθεσία για να λύσουμε κάποια συγκεκριμένα τεχνικά προβλήματα και η τρίτη προσέγγιση η βέλτιστη πρακτική να έχουμε μια πληρέστερη και λεπτομερή πολιτική που θα λειτουργήσει ως ενιαίο πλαίσιο. Ε, και καταλήξαμε στο ότι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε εν μέρει και τις τρεις προσεγγίσεις για να αντίστοιχα με το ποιο πρόβλημα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Για, τις, για την αδειοδότηση, γιατί όπως σας είπα και νωρίτερα είναι από τα βασικότερα προβλήματα Υπάρχει θεωρίου για έναν κανονισμό ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να θεσπιστεί μια απλουστευμένη διαδικασία που θα βασίζεται σε αυτή την ενία θηρίδα, θα διευκολύνει τις αποφάσεις, ε, θα προβλέπονται οι ελάχιστες προθεσμίες για τη χορήγηση άδειας κτλ. Τώρα πρόσβαση και χωροταξικός ε, σχεδιασμός. Ε, είναι ελαφρώς δυσκολότερο το θέμα αυτό διότι υπάρχουν όρια λόγω της κοινοτικής και εθνικής αρμοδιότητας αντίστοιχα σε θαλάσσιες περιοχές μπορούμε να ελπίζουμε σε κάποια πρόοδο και να έχουμε συγκεκριμένη προσέγγιση για την υδατοκαλλιέργεια στα πλαίσια της ε, συνολικότερης διαχείρισης των λευτικών πόρων και της ε, θαλάσσιας πολιτικής. Για το ρυθμιστικό πλαίσιο πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε ο ε, να ληφθούν υπόψη ιδεώντα τα συμφέροντα του κλάδου στην εκπόνηση της πολιτική ενδεχομένω μπορεί να χρειαστεί ε, ειδική προσέγγιση για τα ύδατα, για τα οστρακοειδή. Για τα προστατευόμενα είδη ε, ίσως χρειάζεται καθοδήγηση Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ερμηνεία των ειδικών νομοθετημάτων. Ε, υπάρχει ασάφεια στα κράτη-μέλη σχετικά με το πώς ε, οι οδηγίες για τα πτηνά και τους ε, βιοτόπους εφαρμόζονται. Μπορεί να δημιουργηθούν διαμάχες ως προς, διαφορές ως προς την εφαρμογή των νομοθετημάτων και γι' αυτό σας λέω χρειάζεται καθοδήγηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έγινε διαβούλευση για τους κορμοράνους αυτό το ειδικό ζήτημα και καλωσορίζουμε τις ε, προηγούμενες συστάσεις ε, του ε, Κοινοβουλίου γιατί προτείνεται ένα συνολικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα διαχείρισης για τους κορμοράνους. Θα μπορούσαμε επίσης να εκπονήσουμε ειδικά κριτήρια για τις ευέλτιστες πρακτικές στον τομέα αυτό η υγεία των ε, ηχθείων, οι λεπτομερείς κανόνες ε, για την υδατοκαλλιέργεια, διάφορα τέτοια ζητήματα αναφέρθηκαν στη μελέτη μας. Ε, υπάρχουν ειδικά προβλήματα, ξαναλέω, ορισμένες φορές δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα λόγω των περιορισμών ως προς την αρμοδιότητα και πρέπει να τροποποιήσουμε κάποια νομοθετήματα για να καλυφθούν οι ειδικές ανάγκες της υδατοκαλλιέργειας. Και τέλος, γιατί δεν έχω και πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, ε, ε, πρέπει να δούμε και το ρόλο του διεθνούς εμπορίου, το σύστημα ρυθμίσεων που μπορεί να οδηγήσουν σε διάφορους περιορισμούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει να διαδραματίζει ρόλο κλειδί και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να συντονίσουν το ρόλο τους ώστε να εκπροσωπηθεί ο κλάδος της ε, υδατοκαλλιέργειας στις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Ναι, μία ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Δεν ξέρω αν μπορώ ήδη να κάνω ερωτήσεις. Έφτασε αυτή η ώρα. Ωραία. Λοιπόν, ε, είναι με μία ερώτηση που αφορά και τον τομέα της ενέργειας και τον τομέα της ιδεατοκαλλιέργειας. Και θα σας εξηγήσω τι ακριβώς, σε τι συνίσταται αυτός ο παραλληλισμός. Συνήθως αφορά ζώνες ε, που είναι πιο εύκολες. Οι ζώνες αυτές όμως είναι προστατευόμενες ζώνες. Άρα το ίδιο συμβαίνει και στην υδατοκαλλιέργεια. Έχουμε δηλαδή περί, περίπου το ίδιο πράγμα. Στη Γαλλικία, για παράδειγμα, θέλουμε να ε, κατασκευάσουμε ε, μια εγκατάσταση υδατοκαλλιέργειας, παρά το γεγονός ότι γνωρίζουμε ότι βάσει του Natura 2000 ε, δεν, ανα... δεν είναι ότι δεν σεβόμαστε τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά υπάρχουν σημαντικές και σαφείς συνέπειες. Μπορεί να υπάρχουν και αρνητικές συνέπειες λόγω της εγκατάστασης υδατοκαλλιέργειας σε μια ζώνη που είναι αμυγός προστατευόμενη ζώνη ή που είναι πολύ κοντά στην προστατευόμενη ζώνη. Το πρόβλημα λοιπόν σε προκειμένη περίπτωση είναι η προστασία του περιβάλλοντος και αυτό το αναφέρατε ως σημαντικό. Αλλά αυτό που είναι επίσης σημαντικό είναι ότι δεν είναι μόνο το θέμα του αντικτύπου στο περιβάλλον, μπορεί να υπάρχει και κοινωνικός αντίκτυπος, το γεγονός δηλαδή ότι δίνουμε μεγαλύτερη προτεραιότητα σε μία δράση αντί για μία άλλη. Χρησιμοποιώ λοιπόν το συγκεκριμένο παράδειγμα για να σας πω ότι η προώθηση αυτή τη πολύ εντατική προσπάθεια που γίνεται ούτω ή άλλω στο πλαίσιο τη εραστικτικής αλληλεία και που έχει κάποια κοινωνική προστιθέμενη αξία μεγαλύτερη, επειδή γνωρίζω δηλαδή αυτή την ε, περίπτωση. Αλλά, πάση περιπτώσει, στην έρευνά σα μήπω διαπιστώσατε και άλλου τέτοιου είδους περιπτώσεις. Νομίζω ότι διαπιστώσατε. Πώς μπορούμε λοιπόν να ρυθμίσουμε στις άλλες περιπτώσεις το πρόβλημα. Ε, ναι, θα σα δώσω το λόγο, αλλά πρέπει να πω πρώτα κάτι. Μία εγκατάσταση καλλιέργεια. είναι ένα θέμα αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι εις βάρος της παράκτειας αλίας. Σας δίνω το λόγο για να απαντήσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Είναι πολύ σύνθετη η απάντηση. Συμφωνώ με αυτά που είπατε ότι είναι σημαντικό κοινωνικός αντίκτυπος να ληφθεί επαρκώς υπόψη και το πρόβλημα της ε, τοποθεσίας ε, σε προστατευόμενες ζώνες των εγκαταστάσεων υδαλοκαλλιέργειας δημιουργεί μερικά προβλήματα από ρυθμιστικής ε, πλευράς. Καταρχάς υπάρχει η προστασία της οδηγίας των πτηνών και των βιοτόπων. όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, όπως είπε και η Πρόεδρος, δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι η εγκατάσταση μιας, ε, μιας ε, ότι η εγκατάσταση υδατοκαλλιέργειας θα δημιουργήσει, θα, θα έχει αρνητικό αντίκτυπο σε κάποια προστατευόμενη ζώνη. Δεν είναι υποχρεωτική αυτή η συνέπεια. Αυτό που είναι σημαντικό είναι η προώθηση της καλύτερης κατανόησης της υδατοκαλλιέργειας, της υδατοκαλλιέργειας και των συνεπειών της ε, στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. να υπάρξει καθοδήγηση όλων αυτών των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του EIA ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα τα σχετικά με την υδατοκαλλιέργεια με τον σωστό τρόπο. Και κάτι ακόμη το οποίο αναφέρεται και στην ε, έκθεση, αναφερόταν και στην προηγούμενη, αφορά την προώθηση της θέσης της υδατοκαλλιέργειας ως βασικού παίκτη στις παράκτιες ζώνες. Ένα από τα ζητήματα που αναφέρθηκαν στην έρευνα είναι ότι σε μερικές περιπτώσεις ε, υπάρχει μια ευνοϊκή ε, διάθεση προς την υδατοκαλλιέργεια ακριβώς επειδή υπάρχει καλύτερη κατανόηση του τι ακριβώς είναι. Και φυσικά το αντίθετο ισχύει. Όσον αφορά τώρα τη διαδικασία του χωροταξικού σχεδιασμού, το να υπάρχει συγκεκριμένη αναγνώριση, η κατάλληλη αναγνώριση των προβλημάτων αλλά και των θετικών στοιχείων της υδατοκαλλιέργειας είναι ένα θέμα. Και άλλο ένα θέμα είναι η κατάλληλη καθοδήγηση ε, των ε, συγκρούσεων, αν υπάρχουν, με τις ε, προστατευόμενες ζώνες και πώς θα γίνει η διαχείριση αυτής της κατάστασης. Ε, πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια λύση του προβλήματος που να καλύπτει αυτά τα τρία βασικά ζητήματα που ανέφερα. Σε σχέση με την Ισπανία, ναι υπήρξε ένα πρόβλημα, δεν αναλύσαμε συγκεκριμένες ε, μελέτες, συγκεκριμένες περιπτώσεις, δεν μελετήσαμε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αλλά νομίζουμε ότι αυτές οι τρεις συστάσεις θα βοηθήσουν την επίλυση αυτών των ρυθμιστικών προβλημάτων. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ε, υποβάλω ένα ερώτημα. Μιλάτε για τους περιορισμούς περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Θα ήθελα να ξέρω αν μελετήσετε την κατάσταση της υδατοκαλλιέργειας σε τρίτες ε, χώρες, ισχύουν οι ίδιοι κανόνες ε, για την προστασία του περιβάλλοντος ή δεν υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί στις τρίτες χώρες. Ε, φαντάζομαι ότι έχετε μελετήσει τις τρίτες χώρες, το Βιετνάμ, Φερρυπίν, που έχει ιδιαίτερα ανταγωνιστική υδατοκαλλιέργεια Έχω την εντύπωση ότι δεν ε, τηρούνται βασικές περιβαλλοντικές διατάξεις για κάποια είδη. Θέλω να γνωρίζω λοιπόν αν ισχύουν οι ίδιοι οι κανόνες στις τρίτες χώρες γιατί είναι θέμα ανταγωνισμού και υπάρχουν περιορισμοί ε, λόγω της προστασίας του περιβάλλοντος αλλά θα έπρεπε να ισχύουν οι ίδιοι οι κανόνες παντού. Ε, ευχαριστούμε για την ερώτησή σας. Ναι, βεβαίως, σε μεγάλο βαθμό είναι θέμα ανταγωνισμού. Ε, πραγματικά δεν μας απασχόλησε στα πλαίσια της μελέτης σε μεγάλο βαθμό η κατάσταση στις τρίτες χώρες. Ε, φυσικά οι περιβαλλοντικές ε, διατάξεις είναι πολύ αυστηρότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τρίτες χώρες. Τις τρίτες χώρες που μελέτησαμε Ε, τι εξετάσαμε από, και από αυτή την πλευρά, δηλαδή το κατά πόσο περιορίζονται και εκείνοι από διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Πάντως δεν είναι αυτή η γενικότερη προσέγγιση μας, δηλαδή να θεωρήσουμε ότι είναι υπερβολικές ε, οι περιβαλλοντικές ε, διατάξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε άλλες χώρες δεν είναι επαρκή. Στη Χιλή, παραδείγματος χάρη, δεν έχουν τόσες πολλές διατάξει για την προστασία του περιβάλλοντος και τώρα βλέπουμε να, πάρα πολλά κρούσματα διαφόρων νόσων που πλήττουν και τον κλάδο. Τώρα το να κάνουμε ε, την ε, σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, είναι αυτονόητο ότι δεν υπάρχουν εξίσου αυστηρές ε, περιβαλλοντικές διατάξεις στις τρίτες χώρες. Ο κλάδος είναι υπέρ αυτή τη περιβαλλοντική διάσταση κοινοτική νομοθεσία. Ορισμένε φορέ υπάρχουν επιμέρου ανησυχίε σχετικά με την εφαρμογή τη νομοθεσία και το εύρο τη, αλλά εν γέννη ο κλάδος δέχεται ότι χρειάζεται η περιβαλλοντική νομοθεσία και σε μεγάλο βαθμό θεωρούν ότι συνιστά και ένα δυνατό σημείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ότι υπάρχουν δηλαδή αυστηροί περιβαλλοντικοί κανόνες είναι κάτι που υποστηρίζει ο κλάδος. Οπότε θα απαντούσα καταφατικά ότι προκύπτει θέμα ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος λόγω της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, αλλά δεν μπορούμε και να κάνουμε κάτι έναντι αυτούς. Σας ευχαριστούμε, κύριος Γκούλ. Und hat uns eigentlich noch Πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε. Και προφανώς, αν υπάρχει συγκέντρωση εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας, φυσικά αυτό θα έχει αποτέλεσμα στο περιβάλλον. Αν ε, κατάλαβα καλά από αυτό που είπατε, Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να αποδειχθούμε ότι για παράδειγμα υπάρχει κίνδυνος αύξησης του πληθυσμού των κορμοράνων ε, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την αλία μικρής κλίμακας ε, γιατί το αποτέλεσμα στις μικρής κλίμακας ε, αλλιευτικές δραστηριότητες ε, ε, είναι μικρό λόγω της υδατοκαλλιέργειας. Μήπως χρειαζόμαστε κάποιο πρόγραμμα διαχείρισης, είναι κάτι για το οποίο μιλάμε πολλά χρόνια. Οι συνάδελφοί μας από την Αγγλία, από τη Σκοτία ανησυχούν για τους πληθυσμούς της φώκιας και άλλων θαλασσίων οργανισμών που τρέφονται με ψάρια και που είναι αρκετά, τα ψάρια αυτά είναι αρκετά, σε αρκετά υψηλό σημείο στη διατροφική αλυσίδα. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και να προστατεύουμε τη φύση, αλλά και να αγωνιζόμαστε για μια βιολογική ισορροπία. Οι κορμοράνοι τρώνε 500 γραμμάρια ηχθείων την ημέρα και είναι τα προστατευόμενα είδη. Ε, Πώ είναι δυνατόν λοιπόν να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κατάσταση. Προφανώ δεν θέλουμε να εμφανιστούν και πάλι ε, στην ε, κόκκινη λίστα, αλλά αυξάνει το πληθυσμό των κορμοράνων με δυσανάλογο τρόπο. Μήπω και αυτό κάτι είναι που πρέπει να το αντιμετωπίζουμε όταν θέλουμε να επιτύχουμε μια βιολογική ισορροπία. Συνομιλήσαμε και με τους συναδέλφους μας ε, στην ομάδα των ε, Πρασίνων ε, στην Γερμανία. Είναι το πτηνό του έτους η Κορμοράνη. γίνονται... Ε, πολλές φορές θυρεύουν και σε περιοχές μακριά από τις ακτές και τους αποκαλούν τρομοκράτες των ανοιχτών θαλασσών. Μάλιστα, μπορούμε να τους αποκαλούμε από τώρα τότε τους κορμοράνους τρομοκράτες του έτους. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Υπάρχουν πολλές υπηρεσίες που λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο εντός των κρατών, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σαν να μου φαίνεται ότι χρειαζόμαστε μια κοινή πολιτική. Υπάρχει κάτι που με ανησυχεί πάρα πολύ στην ε, απάντηση που δώσατε στην ε, Πρόεδρο. Εδώ μιλούμε για δημόσια υγεία. Υπάρχουν και οι νόσοι των ηχθείων που προέρχονται από τις ε, ιδιοτροφές ενδεχομένως και νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχουν παγκόσμιες απαιτήσει ε, και αυτό συνδέεται άμεσα με την υδατοκαλλιέργεια γιατί όλο και περισσότεροι χθιές θα πρέπει να προέρχονται από την υδατοκαλλιέργεια. Αν δεν υπάρχουν λοιπόν σαφείς κανόνες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και εφόσον οι τρίτες χώρες δεν υπακούν στους κανόνες αυτούς, ε, τότε τι δικλείδες ασφαλείας υπάρχουν όσον αφορά τη δημόσια υγεία των καταναλωτών. Υπάρχει καμιά νομοθεσία. Υπάρχει κανένας έλεγχος. Πολύ συχνά από αυτά που ακούω υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα δημόσιας υγείας που σχετίζεται με την υδατοκαλλιέργεια. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Πατράου Νέβες, ευχαριστώ. Αυτό το θέμα της υδατοκαλλιέργειας ε, μου γεννά διάφορα ερωτηματικά. Θα ήθελα ε, στο μέτρο του δυνατού να πάρω κάποιες απαντήσεις σε πολλά και διαφορετικά ερωτήματα, ξαναλέω. Θα ήθελα αρχίζοντας να πω αυτό που μόλις ακούσαμε, ότι ε, δεν υπάρχει πια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική και θα, αυτό θα ήταν καθοριστική σημασία ούτως ώστε όλα τα κράτη-μέλη να μπορέσουν στη συνέχεια να θεσπίσουν ε, το κατάλληλο πλαίσιο για την άσκηση αυτής της δραστηριότητας. Χωρίς αυτό το πλαίσιο οι επιχειρήσεις δύσκολα θα αναλάβουν ε, πρωτοβουλίες και θα κάνουν σημαντικές επενδύσεις. Αυτό το νομικό, ρυθμιστικό πλαίσιο για αυτή την ε, δραστηριότητα της υδατοκαλλιέργειας θα μπορούσε να προάγει την ε, δραστηριότητα αυτή και να ανεβάσει τα επίπεδα παραγωγικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτό μεταξύ άλλων είναι ένας από τους σημαντικότερους στόχους μας. Επίσης, θα ήθελα να σας ρωτήσω στα ίδια πλαίσια το εξής ε, ε, ο προσδιορισμός των θαλασσίων περιοχών, ε, ο χωροταξικός ε, σχεδιασμός των παρακτήων περιοχών και των γεωγραφικών περιοχών που είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για τη διεξαγωγή αυτής της δραστηριότητας έχει ήδη αποφασιστεί ότι θα γίνει και ποιοι όροι ισχύουν, ειδικοί όροι για το θαλάσσιο περιβάλλον, γιατί δεν είναι μόνο θέμα περιβάλλοντος, είναι θέμα και ειδών για τα οποία θα γίνει επένδυση. Για να μην είμαστε καταδικασμένοι στην επιλογή των ίδιων ειδών κάθε φορά για την υδατοκαλλιέργεια. Μπορούμε να διαρευνήσουμε και άλλε δυνατότητε διαφορετικά είδη εξίσου υψηλή ποιότητα που μα προσφέρουν και μια υψηλότερη προστιθέμενη αξία. Και να προσθέσω εδώ ότι ορισμένα είδη μπορεί να μην δημιουργούν τόσο σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα ε, ε ως προς τη διατροφή των νυχθείων αυτών. Ε, μία άλλη πτυχή τώρα. Ο φόβος διαφόρων αλλιών για την υδατοκαλλιέργεια. Τι λένε, πως ε, φοβούνται ότι η τιμή του άγριου ε, ψαριού πέφτει λόγω της ε, υδατοκαλλιέργειας και πλήττεται περαιτέρω η βιοτεχνική, η ερασιτεχνική αλία με την περαιτέρω ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας. Θα μπορούσατε να μας απαντήσετε. Η υδατοκαλλιέργεια κυρίως η offshore ε, απαιτεί ειδικό εργατικό δυναμικό, δηλαδή αλίησε και όχι οποιοδήποτε άλλος αλληλείς που έχουν υψηλότερη κατάρτιση, παραδείγματο χάρη. Εάν συμβεί αυτό, δεν θα μπορούσε η ιδιατοκαλλιέργεια να συμβάλλει ούτως ώστε ε, να, να έχει μια καλύτερη εικόνα το επάγγελμα και να προσελκύσει και νέους. αυτό είναι ένα από τα προβλήματα της υδατοκαλλιέργειας, ότι δηλαδή δεν έχει δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης. Οπότε με ποιο τρόπο μπορεί να υποφεληθεί από αυτό η υδατοκαλλιέργεια, δηλαδή από αυτά που ήδη ισχύουν ναι, στον αλλιευτικό τομέα αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, έχει γίνει έμονη ιδέα, αλλά θα επανέλθω στι αγωγές από τις ε, τρίτες χώρε. Δεν υπάρχει καμία ιχνηλασιμότητα ε, υγειονομική, ούτε περιβαλλοντική, για είδη όπως ε, η τιλάπια, για παράδειγμα. Διορθώστε με αν κάνω λάθος και άκουσα κάτι το οποίο με σώκαρε πάρα πολύ. Κύριε Λέιν, μα είπατε προηγουμένως ε, ότι είναι ενδεχομένω κάτι με το οποίο θα πρέπει να ζήσουμε. Αυτό μα είπατε. Εγώ δεν έχω καμία όρεξη να ζήσω με αυτό, σας το λέω. Καθόλου. Νομίζω ότι πρέπει να ρυθμίσουμε το πρόβλημα αυτό των εισαγωγών ε, ε, και της χνηλασιμότητας, της περιβαλλοντικής και της υγειονομικής πριν αναπτύξουμε την υδατοκαλλιέργεια, την οποία πρέπει να την αναπτύξουμε. Δεν λέω, αλλά δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να ακούω τέτοια πράγματα. Για μένα είναι απαράδεκτο. Και αφού δεν έχουμε λύσει αυτό το πρόβλημα, αν δεν λύσουμε αυτό το πρόβλημα των εισαγωγών ε, από τις ε, τρίτες χώρες, ε, δεν θα αναπτύξουμε με συνεκτικό και σωστό τρόπο την υδατοκαλλιέργειά μας, γιατί εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε, όλοι το επιθυμούμε αυτό και μάλιστα με υδατοκαλλιέργεια που θα σέβεται το περιβάλλον και επίσης τις τιμές που θα πληρώνουμε στους αλληλείς μας. Δεν είναι δυνατόν, πρέπει να είναι κάτι το συμπληρωματικό, είναι μία από τις απαντήσεις δεν είναι η μόνη απάντηση, παρά το γεγονός ότι είναι απαραίτητη. Ευχαριστώ. Ε, παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο που αφορά πιο πολύ τον πρώτο ομιλητή για την αναπτυξιακή πολιτική, για την ευρωπαϊκή δατοκαλλιέργεια δεν άκουσα πολλά στοιχεία σχετικά με το ποια είδη κατά τη γνώμη σας ε, θα πρέπει να μας απασχολήσουν περισσότερο στην υδατοκαλλιέργεια. Ο ΦΑΟ ε, μας ε, υπολογίζει ότι το 30% των αλλιευμάτων χρησιμοποιούνται ως τροφή για τα εκτρεφόμενα ψάρια. Και στη Σουηδία το ποσοστό αυτό είναι 60% των αλλιευμάτων που γίνονται ηχριάλευρα. Και θα συμφωνήσω ο συνάδελφο από την Πολωνία ότι είναι ιδιαίτερα προβληματική η κατάσταση. Δηλαδή όταν ψαρεύουμε για να έχουμε τροφή για τα εκτρεφόμενα ε, ψάρια, ενώ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ανθρώπινη ε, κατανάλωση. Μιλώ για τη Σαρδελόρεγκα παραδείγματο χάρη στη Βαλτική θάλασσα. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στη Ρωσία. Αυτά τα ψάρια χρησιμοποιούνται και για ανθρώπινη κατανάλωση και τα χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε ηχθιάλευρα και το ίδιο στη Δανία που μεταφέρουν ε, ηχθιάλευρα για τους Σολομούς ε, ε, στη Βόρεια Νορβηγία ή μεταφέρονται στην Κίνα για να τα συσκευάσουν γιατί είναι φτηνότερο και μετά τα ξαναστέλνουν στη Σουηδία και ε, θα είχαμε περισσότερες δρέγγες, περισσότερα άγρια ψάρια, περισσότερα αλλιεύματα τελικά, αν τα προστατεύαμε περισσότερο. Ε, δηλαδή πρέπει να προστατεύσουμε καλύτερα τα αποθέματα άγριων ψαριών ε, για να βελτιώσουμε την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό πρέπει να επενδύσουμε. Αν όντω πρέπει τώρα να αυξήσουμε τα επίπεδα υδατοκαλλιέργειας, θα έπρεπε ίσως να εστιάσουμε σε κάποια διαφορετικά είδη. Αυτό είναι το μέλλον είχα κατά τη γνώμη μου και επίσης ποιες φυσικές προϋποθέσεις υπάρχουν στην Ευρώπη, στην Νότια Ευρώπη παραδείγματο χάρη. Ε, ε, ε, στην Νορβηγία έχουμε όλα τα φιόρντ, όλα αυτά τα χιλιόμετρα παραλίας ανοιχτή ε, θάλασσα που έχει γεμίσει με τα ε, ηχθιάλευρα αυτά, με την τροφή για τα ψάρια και τα περιτώματα των ψαριών λόγω της ε, υδατοκαλλιέργειας. Είναι ε, ουσιαστικό ε, πρόβλημα. Δηλαδή πρέπει να δούμε ποιε είναι οι φυσικές προϋποθέσεις. Ίσως πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κλειστά συστήματα ή παλιά ορυχεία ή... Δεν νομίζω ότι σε όλες τις χώρες υπάρχουν αντίστοιχα καλές προϋποθέσεις ε, για τα άγρια ψάρια, ε, όταν ε, μιλάμε για γάδο, παραδείγματο χάρη για μπακαλιάρο, για σολομό, αφού υπάρχουν, γιατί ε, να επιλέγουμε αυτά τα είδη για την υδατοκαλλιέργεια και να καταστρέφουμε άλλα ψάρια για να θρέψουμε τα εκτρεφόμενα ψάρια. Δεν είναι καλό για την βιωσιμότητα των φυσικών πόρων όταν τώρα Μιλάμε για τις εισαγωγές από άλλες χώρες ε, υπάρχουν πολλά ψάρια που εισάγονται από την ε, Νορβηγία και η Νορβηγία έχει αυστηρότερου κανόνε. Όταν μιλάμε όμω για το Βιετνάμ ή για άλλε ασιατικέ ε, χώρε, ναι, θα πρέπει να απαιτήσουμε υψηλότερε, αυστηρότερε μάλλον διατάξει για να προστατεύσουμε τον καταναλωτή. Υπάρχει και η περιβαλλοντική πιστοποίηση. Αυτό είναι σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση ω προ τον ανταγωνισμό. Θα συμφωνήσω μαζί σα. Χρειαζόμαστε μια περιβαλλοντικού τύπου πιστοποίηση για την ευρωπαϊκή αλία, ούτως ε, θα, και αν ισχύσει αυτό θα το ζητάει ο καταναλωτής για όλα τα προϊόντα, ακόμη και για τα εισαγόμενα. Το βλέπουμε στη Δανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γερμανία, ακόμη και στη ΣΥΠΑ. Δηλαδή ε, θέλουν, ε, θέλει ο κλάδος να μεταπολεί μόνο περιβαλλοντικώς πιστοποιημένα προϊόντα. Έτσι θα υποχρεώσουμε και τις εγκαταστάσεις διδατοκαλλιέργειας που υπάρχουν στις ασιατικές χώρες να ακολουθήσουν την ίδια πιστοποίηση για να καλύψουν τις απαιτήσει των Ευρωπαίων καταναλωτών. Πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν βασικές διαφορές ανάμεσα στη γεωργία και στη διδατοκαλλιέργεια. Περνώ σε ένα διαφορετικό θέμα. Δεν μπορούμε να κάνουμε ε, να επιβάλλουμε τα ίδια μέτρα την αγρανάπαυση ας πούμε στην υδατοκαλλιέργεια πρέπει να καθαρίσουμε ότι πρόκειται για δύο διαφορετικούς τομείς και ελπίζω ότι θα υπάρξει ειδική ευρωπαϊκή στρατηγική για βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια και θα επενδύσουμε ε, στα είδη που πρέπει και θα επενδύσουμε στο eco-labeling και στην περιβαλλοντική πιστοποίηση. Εν πάση περιπτώσει, Στη συνέχεια ο κύριος Μούι θα παρέμβει. Κάποια από τα θέματα λοιπόν θα είναι αντικείμενο της επόμενης μελέτης. Ο κύριος Μούι θα ήθελε να παρέμβει τώρα για να απαντήσει τώρα, ας μην επισπεύσουμε. Για να ολοκληρώσουμε, κύριος ε, Γκάρα και κυρία Μιλάνα, θα απαντήσουν όποιος θέλει από εσά τους τρεις ή τους προσκεκλημένους. Γκάλαγκερ πρώτα και μετά Μιλάνα, παρακαλώ. Yeah, Πάρα πολύ σύντομα, η Πρόεδρε, για τη σημασία των ερευνών, των μελετών για τις ε, υδατοκαλλιέργειες. Ε, υπήρξε μια σημαντική μείωση τα τελευταία χρόνια της απασχόλησης ε, στον τομέα των άγριων ηχθείων, των μη εκτρεφωμένων και είναι γεγονός ότι η υδατοκαλλιέργεια συμβαίνει συνήθως στις παράκτιες ζώνες και μπορεί βέβαια να δώσει πολλές ε, θέσεις απασχόλησης στις περιοχές αυτές και τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη μπορούν να υποστηρίξουν την προσπάθεια αυτή, γιατί είναι εύκολο να ξεκινήσει μια εγκατάσταση υδατοκαλλιέργεια. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει η επένδυση. Νομίζω ότι και ο τοπικό κλάδος μπορεί κάθε φορά να κάνει μια πρώτη επένδυση. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και νομίζω ότι κάποιο από του προλαλήσαντε μίλησε για τον δίκαιο ανταγωνισμό. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει δίκαιο ανταγωνισμός. Ε, οι ελάχιστε τιμέ εισαγωγών, ε, είχαμε κάποια προβλήματα με την Ορβηγία, με τι εισαγωγέ Σολομού, αλλά και με εισαγωγέ από άλλε χώρε Και αυτό μπορεί να έχει επιβλαβεί συνέπειε στην ε, υδατοκαλλιέργεια στο, στη δική μου χώρα. Αυτά όμω είναι στο παρελθόν και ελπίζουμε ότι δεν θα συνεχίσουν τέτοιου είδου καταστάσει. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Μιλάνα, παρακαλώ. Έχω την εντύπωση, όπω και η πρόεδρο, ότι έτσι επισπεύδουμε τη συζήτηση και προδικάζουμε τη συζήτηση που θα διεξαχθεί αργότερα. Το γεγονό είναι το εξή. Οι μελέτε είναι μελέτε. Δεν μπορεί κανεί να απαιτήσει από μια μελέτη να δώσει πολιτικέ απαντήσει σε ένα θέμα. Όμως ένας περιορισμός που βλέπω να υφίσταται εγώ είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει τέτοιου είδους, ας το πούμε έτσι, λύση από μια μελέτη. Θα μπορούσε να αποκλειστεί λοιπόν η ιδέα μιας κοινή πολιτικής ε, υπό ένα κοινοτικό πλαίσιο. Πιστεύω ότι ένα από τα πράγματα που η βιομηχανία και που οι εμπλεκόμενοι στη βιομηχανία δεν θα επιθυμούσαν είναι μια κοινή ενιαία πολιτική. Φυσικά το γεγονός ότι δεν αρέσει στη βιομηχανία μια πολιτική δεν αποκλείει αναγκαστικά αυτή την πολιτική, διότι είναι κάτι το οποίο ξεπερνά τα στενά πλαίσια συμφερόντων. Χρειαζόμαστε όμως περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες εδώ για τα θέματα τα οποία συζητούμε σήμερα. Είναι ένα θέμα εδώ που πιστεύω ότι δεν μας έδωσαν οι μελέτες μια επαρκή εξειδικευμένη απάντηση ακόμα. Ένα φαινόμενο υπήρξε στην εφαρμογή του, της πολιτικής ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2002 όταν είχαμε ποσοστό ανάπτυξης 6 και 7% ενώ στη συνέχεια υπάρχει αποτελμάτωση και τώρα έχουμε και τον ανταγωνισμό από αμφισβητήσιμες άλλες χώρες όπου δεν υπάρχουν κανόνες υγιεινής για παράδειγμα. Και η απάντηση σήμερα δεν είναι ότι χρειαζόμαστε περισσότερες συστάσεις. Όχι, χρειαζόμαστε μια πραγματική πολιτική που θα φέρνει αλλαγές και θα αλλάξει τα πράγματα. Φυσικά γνωρίζοντας ότι οι μελέτες συντάσσονται και στοχεύουν προς την ίδια κατεύθυνση όπως και συστάσεις που διατυπώνονται, χρειάζεται επιτυχία. Και εσείς τώρα που θα παρέμβετε δεν συνεπάγεται ότι οι άλλοι δεν μπορούν να παρέμβουν. Θα περάσουμε μετά στην τρίτη μελέτη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ και πάλι πρόεδρε. Και για το θέμα το οποίο αναφέρθηκε σε ρυθμιστικά θέματα και κάποια από τα θέματα τα οποία αφορούν τις ε, ε, επόμενες μελέτες. Τα ερωτήματα που υπάρχουν μετά την τελευταία παρουσίαση θα μπορούν να εξεταστούν. Θα προσπαθήσω να εξετάσω με τη σειρά τα θέματα τα οποία τέθηκαν. Ξεκινώ με το θέμα της ε, σε εισαγωγικά τρομοκρατίας. Νομίζω ότι το είδαμε αυτό το θέμα στην έκθεσή μας και καταλήξαμε στο ίδιο συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε και εκείνος οι οδηγίες για τους οικοτόπους και τους βιοτόπους προσφέρουν ένα μηχανισμό για να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα των προστατευόμενων ειδών όπου υπάρχουν τέτοιου είδους τριβές και προβλήματα. Το πρόβλημα όμως ε, κυρίως είναι το ότι τα κράτη-μέλη δεν γνωρίζουν ακριβώς πώς να εφαρμόσουν αυτή την νομοθεσία. Υπάρχουν πολλά αμφίσιμα θέματα όσον αφορά την ερμηνεία της νομοθεσίας. Τα κράτη-μέλη υιοθετούν διαφορετικές προσεγγίσεις και δεν υπάρχει, ας το πω έτσι, σε σχέση με τις ε, ε, παρεμβάσεις ε, δεν υπάρχει δυνατότητα για παράδειγμα να προωθηθούν τέτοια θέματα. Εκείνο το οποίο είναι σημαντικό είναι να δούμε το θέμα των μελετών για αυτά τα θέματα και τις, τα προβλήματα που είχαν οδηγήσει σε κάποια πιο αφήσιμα αποτελέσματα. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να είναι σαφές για τα κράτη-μέλη τι επιτρέπει και τι όχι η νομοθεσία. Και κατευθυντήρες γραμμές και προσανατολισμοί που θα αναπτυχθούν με, από κοινού με τους εμπλεκόμενους βοηθούν σίγουρα. Είναι όμως σημαντικό να υπάρξει και μια επιστημονική, ας το πω που θα α, υιοθετηθεί. Το να πει ένας νομομαθής, για παράδειγμα ένας νομικός, ότι εντάξει μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μία ή άλλη προσέγγιση όσον αφορά προβλήματα με φώκες ή ε, ε, πρέπει να δούμε μέσα στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας τι επιτρέπεται. Γι' αυτό συνιστούμε καλύτερες ε, προσανατολιστικές γραμμές, κατευθυντήριες γραμμές. Αποκινούμε τους εμπλεκόμενους και με κοινή επιστημονική συνένεση. Επίσης αναφέρεται ότι αυτό συζητείται και επί μεγάλο χρονικό διάστημα και ένα ευρωπαϊκό τέτοιο πρόγραμμα θα ήταν οπωσδήποτε επωφελές όπως είχε συσταθεί και στο παρελθόν. Δύο-τρία θέματα τα οποία αφορούν και το θέμα της ε, α, κοινής ε, αγροτικής πολιτικής, της ΚΑΠ. Χαιρετίζω τα σχόλια του κυρίου Μιλάνα ότι δεν είναι δουλειά μιας μελέτης να υποβάλει συστάσεις ε, πολιτικές, πολιτικής βρίσκεται εξάλλου και σε μεγάλο βαθμό εκτός του πλαισίου αναφοράς. Όμως σύντομα εξετάστηκαν θέματα που αφορούν και την ΚΑΠ, γιατί είναι ένα προφανές θέμα ότι κάτι τέτοιο θα το ρωτούσε κάποιος. Τώρα, όσον αφορά συνολικά το πλαίσιο της μελέτης, ένα από τα συμπεράσματα είναι ότι δεν υπήρξε μια πλήρης σφαιρική συζήτηση ολοκληρωτικά επ' και φαίνεται ότι υπάρχει περιορισμένο ενδιαφέρον για αυτή την προσέγγιση από πλευρά βιομηχανίας. Το σημειώνουμε αυτό σε σχέση με τις ε, απαντήσεις και αντιδράσεις για την αναθεώρηση της στρατηγικής όσον αφορά το 2009 και για το, την ε, τάση υπέρ της ε, πορείας που ακολουθήθηκε για την ΚΑΠ. Εδώ σε σχέση με τα όσα μπορούν να επιτευχθούν δεν είναι ευρύ το πλαίσιο, διότι πολλά πράγματα βρίσκονται εκτός του εύρους του κοινοτικού δικαίου και της κοινοτικής νομοθεσίας. Η ΚΑΠ δεν μπορεί λοιπόν να επιλύσει αυτά τα ζητήματα που εκκρεμούν. Και υπάρχει και το θέμα ακόμα θα έλεγα, το οποίο δεν μπορούσαμε να απαντήσουμε εμείς, αλλά είναι το ζήτημα κατά πόσο θα βοηθούσε κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε σε αυτή τη φάση ότι ίσως η προσέγγιση της ΚΑΠ θα μπορούσε να ήταν μια προσέγγιση, αλλά δεν βρίσκουμε να είναι πιστικά τα τεκμήρια που να δείχνουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Ένα από τα θέματα τα οποία αναφέρθηκαν ήταν ότι υπάρχει ανάγκη για όπως και για την ΚΑΠ, γιατί χρειαζόμαστε ρυθμίσεις για όλες αυτές τις πτυχές Άλλοι ομιλητές αναγνώρισαν ισχυρό ενδιαφέρον για υγειονομική, για θέματα υγείας που πρέπει να ρυθμίζονται. Αυτό καμιά φορά σε σχέση όσον αφορά με τις ε, βιομηχανίες ε, όσον αφορά τη, τη γεωργία και τα προϊόντα της, τι πρέπει να γίνει. Έχουμε διαφορετικές γενικές διευθύνσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση με διαφορετικά ε, προγράμματα. Ένας ε, ε, τρόπος θα ήταν να υιοθετήσουμε μια περισσότερο συντονισμένη αντιμετώπιση αυτών των θεσμάτων από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Αν βγάλει αυτές τις πτυχές κανείς της γεωργίας, αντιμετωπίζει το πρόβλημα του αντίστροφου σε σχέση με το περιβάλλον και το πώς θα μπορούσαν διάφορες παράμετροι να ρυθμιστούν. Και σε κάποια χρονική στιγμή, ανάλογα με το ποια πλευρά υιοθετεί κανείς, πρέπει να υπάρξει μια ρύθμιση και μια ε, διευθέτηση. Τελικά το συμπέρασμα είναι δεν, ότι δεν είναι κάτι το οποίο έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη αυτή τη στιγμή. Ναι, μπορούμε να μιλάμε για την ΚΑΠΑ, όμως βρίσκεται ε, αρκετά μακριά από το σενάριο αυτή τη στιγμή. Πρέπει να υιοθετήσουμε μια πιο πρακτική προσέγγιση για το τι μπορεί να γίνει σύντομα και πιο αποτελεσματικά, πιο γοργά και με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Κάποιος ανέφερε ανησυχίες για τα θέματα δημόσιας υγείας, για τα θέματα ασθενειών ε, ηχθείων. Μπορώ να πω ότι υπάρχει ρύθμιση, αλλά όχι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν τέτοιες ρυθμίσεις όσον αφορά υγειονομικούς ελέγχους και σε σχέση με τις ε, ε, δράσεις όσον αφορά την γεωργία. Υπάρχει αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, είναι δεδομένο και η εντύπωση είναι ότι υπάρχει εξειδίκευση στη ρύθμιση και έτσι σε σχέση με τους κινδύνους δεν είναι οι ίδιοι όπως υπήρχαν αλλού. Θα συνεχίσω αν επιτρέπετε, έχω κάποιες σημειώσεις εδώ, κάποια θέματα. Αναφέρθηκε επίσης ε, για τις παράκτιες περιοχές ε, και τον σχεδιασμό και αν όλα αυτά εντάσσονται μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Η απάντηση είναι ότι δεν, είναι αυτό σε, δεν γίνεται αυτό σε μεγάλο εύρος. Μέσα στο πλαίσιο λοιπόν της πολιτικής για τις ε, δραστηριότητες, ε, τις θαλάσσιες δραστηριότητες θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την προαγωγή και του ε, ρόλου αυτού όσον αφορά γεωργικές δραστηριότητες στις παράκτιες περιοχές. Πρόεδρος, με συγχωρείτε που σας διακόπτω Ας δώσουμε τον λόγο στη συνέχεια στον κύριο Μουρ για την παρουσίαση της τρίτης έκθεσης και στη συνέχεια θα ρυθμίσουμε τα θέματα που εκκρεμούν. Γιατί έχουμε και ένα σημείο στην ημερησία διάταξη του κυρίου Μιλάνα. Στις 12.30 πρέπει να ολοκληρώσουμε, θα αποχωρήσουν οι διερμηνείς. Έτσι λοιπόν, μια και ο επόμενο συζητητή έχει ένα θέμα το οποίο αναμειγνύεται με πολλέ ερωτήσει, ο κύριο Μουρ θα πάρει τον λόγο για 15 λεπτά το πολύ, παρακαλώ. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη τη Επιτροπής, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Θα έχω κατά νου, δεν έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας. Εξετάσαμε το θέμα της ανταγωνιστικότητας και των περιορισμών που υπάρχουν στην ευρωπαϊκή βιομηχανία και τις πιθανές στρατηγικές που μπορούμε να υιοθετήσουμε για να ρυθμίσουμε κάποια από τα προβλήματα που εντοπίσαμε. Ανάμεσα στόχους της μελέτης ήταν να εξετάσουμε αυτούς τους περιορισμούς του κλάδου και κυρίως το ότι αποτελεί φραγμό στην ανάπτυξη του δυναμικού του κλάδου. Εννιά τομείς εξετάσαμε συγκεκριμένα. Θα επανέλθω σε αυτό αμέσως. Είδαμε επίσης ε, τις ε, τελευταίες εξελίξεις στην έρευνα και στην τεχνολογία στην Ευρώπη και σε ποιο βαθμό είναι χρήσιμες αυτές οι εξελίξεις και αντισταθμίζουν κάπως τους περιορισμούς. Για να δούμε την αποτελεσματικότητα των ε, τεχνολογικών, της τεχνολογικής πλατφόρμας και τις επιπτώσεις και να κάνουμε την ανάλυση SWOT Κάποια πορίσματά μας ε, επιτρέπουν να διαμορφώσουμε την εικόνα του κλάδου. Κάποιες γενικότερες θεματικές ενότητες στον τομέα της ανταγωνιστικότητας είναι οι εξής. Έχουμε πολλά και διαφορετικά προϊόντα, πολλά και διαφορετικά παραγωγικά συστήματα και πολλούς και διαφορετικούς φορείς εμπορικούς φορείς. Υπάρχουν δυνατότητες οικονομίας κλίμακος σε κάποιες περιοχές ε, και ε, σε αυτούς τους τομείς έχουμε ε, ανταγωνιστικότητα υψηλής κλίμακος, αλλά συχνά υπάρχουν περιορισμοί λόγω των χώρων και των πόρων. Η ανταγωνιστικότητα έγκυται στις τιμές στον κλάδο αυτό και υπάρχουν κάποια προϊόντα με χαμηλότερες τιμές και φυσικά ε, ε, υπάρχει ανταγωνιστικότητα των φθηνών προϊόντων, των εισαγόμενων προϊόντων υδατοκαλλιέργειας. Ε, επίση η μεταποίηση και η διανομή είναι άλλη σημαντική τομή στην Ευρώπη παρότι η ανταγωνιστικότητα της παραγωγή είναι από μόνη της σημαντική. Πρέπει παρόλα αυτά να δούμε το γενικότερο πλαίσιο, δηλαδή ακριβώ που υπάρχει οικονομική προστιθέμενη αξία και ε, η μεγαλύτερη προσθέμενη αξία βρίσκεται στην μεταποίηση των ε, ευρωπαϊκών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και των προϊόντων από τις τρίτες χώρες. Τώρα για την έρευνα και την τεχνολογία ε, αυξάνεται ουσιαστικά η βάση των γνώσεων της βιομηχανίας, αλλά οι τελευταίες εξελίξεις ε, δεν αλλάζουν ούτε το εμπορικό περιβάλλον, ούτε την πολιτική που εφαρμόζεται. Είδαμε την ανάλυση SWOT ε, για διάφορα βασικά είδη και τη σχετική παραγωγή και μάλλον παρεμφερή αποτελέσματα καταλήξαμε. Η τεχνολογική πλατφόρμα, γιατί μία υπάρχει μόνο που έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την υδατοκαλλιέργεια, έχει τη δυνατότητα να αντισταθμίσει κάποιους από τους περιορισμούς. Έχουμε εννιά τομείς ανταγωνιστικότητας που μας απασχόλησαν στη μελέτη και είναι οι εξή, όπως βλέπετε και στη διαφάνεια. Ε, μάλλον ομαδοποιήσαμε τους τομείς σε θεματικές ενότητες γιατί υπάρχουν ε, είναι αλληλένδετοι οι τομείς ως προς επιπτώσεις που έχουν για την υδατοκαλλιέργεια. Τώρα, ε, ε, το πρώτο ζήτημα είναι οι ρυθμιστικές διατάξεις, αλλά θα το σχολιάσω τελευταίο, γιατί έχουμε ακούσει πολλά στοιχεία για αυτό το ζήτημα και θα προκύψει από την υπόλοιπη παρουσίασή μου. Το ζήτημα του περιβάλλοντος επίσης σχολιάστηκε σε προηγούμενες παρεμβάσεις. Υπάρχει το θέμα του ανταγωνισμού της αγοράς ε, και της ρύθμισης αγοράς ε, και το θέμα των τεχνολογικών ε, εξελίξεων και του κόστους παραγωγής. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι αλληλένδετα. Σε κάθε μία από αυτές τις θεματικές ενότητες κάναμε γενικές αναλύσεις SWOT και καταλήξαμε στα εξής συμπεράσματα. Ξέρετε, δεν έχω και πολύ χρόνο για να ε, μπω σε λεπτομέρειες, αλλά είναι μάλλον αυτονόητα τα συμπεράσματα. Το σημαντικότερο σε, αυτό το, σε αυτή τη θεματική ενότητα, όπως σας είπα, είναι ότι έχουμε περιορισμούς και οι υποχρεώσεις ε, με τις οποίες πρέπει να συμμορφωθούμε σε σχέση με άλλους χρήστες του περιβάλλοντος και η πρέπει να δούμε το ρόλο της υδατοκαλλιέργειας ε, στην ενδοχώρα και στις ε, παράκτιες ε, ζώνες και πόσο μπορούμε να εφαρμόσουμε τις μυστικές διατάξεις. Η σύσταση είναι να έχουμε έναν ευρύτερο ορισμό του οικοσυστήματος για να γίνεται καλύτερη περιβαλλοντική διαχείριση και να προάγουμε καλύτερες χωροταξικές πολιτικές και παρεμφερές κόστος για όλους τους παραγωγούς Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάμεσά τους και τους παραγωγούς Ένωσης σε σχέση με τους παραγωγούς των τρίτων χωρών για τον ανταγωνισμό και τη ρίχνη ρύθμιση της αγοράς, οι βασικοί είναι η εξής. Έχουμε μία ισχυρή αγορά στην Ευρώπη. Έχουμε καλές δυνατότητες για να προάγουμε, να προωθήσουμε τα προϊόντα της υδατοκαλλιέργειας ε, λόγω των, ε, του ωφέλους που έχουν. Έχουμε δυνατότητα να επιβάλλουμε ίσους όρους ανταγωνισμού για τους παραγωγούς Ένωσης και τους λοιπούς παραγωγούς. Προσπαθούμε να προάγουμε και συστήματα περιβαλλοντικής επιστοποίησης, eco-labeling κτλ. Αλλά δημιουργείται η σύγχυση λόγω της επληθώρας των σημάτων και των ε, συστημάτων ε, επιστοποίησεων. Ε, σύγχυση που δημιουργείται στο μυαλό των καταναλωτών πρέπει να ξέρουν τι αγοράζουν. Προκύπτει ε, εξ αυτού η εξή σύσταση. Θέλουμε η υδατοκαλλιέργεια να συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση του περιβαλλοντος. Αυτό φαίνεται στη, στα μέτρα και στην πολιτική που προτείνεται ε, πρέπει να έχουμε ένα, ε, ως Ευρώπη ηγετικό ρόλο για σαφή σαφή και καλά περιβαλλοντικά πρότυπα που θα ευθυγραμμίζονται με τα διεθνή πρότυπα στον τομέα αυτό. Τώρα για την τεχνολογία και το κόστος ε, ακούστηκαν διάφορα στοιχεία στις προηγούμενες παρεμβάσεις. Ε, μία από τις ε, βασικές ανησυχίε είναι φυσικά αυτό το θέμα των τροφών για τα ψάρια υδατοκαλλιέργειες έχει σημειωθεί σημαντική τεχνολογική πρόοδος τα τελευταία χρόνια. Ε, είδαμε τα στοιχεία για τη ζήτηση για τα ηχθιάλευρα και τα ηχθιέλεα, παραδείγματος χάρη. Ε, λοιπόν, βλέπουμε ότι ε, υπάρχει όλο ένα και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και καλύτερη απόδοση στον τομέα αυτό προσπαθούμε να εγκαταστήσουμε οικονομία κλίμακας χρησιμοποιώντας πιο προηγμένες τεχνολογίες στον τομέα αυτό. Υπάρχουν ε, περιορισμοί βέβαια ε, στις ανταλλαγές ε, τεχνογνωσίας στην Ευρώπη, αλλά υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Η σύσταση που θα έπρεπε να ακολουθήσουμε σε αυτό το τομέα είναι ότι χρειάζονται μεγαλύτερες επενδύσεις στη στοχευμένη έρευνα από πλευράς της βιομηχανίας για να αξιοποιήσουμε στο έπακρον τον ενιαίο ευρωπαϊκό ερευνητικό χώρο. Εξετάζοντας το θέμα της τεχνολογικής πλατφόρμας υπάρχουν και κάποια ειδικά ζητήματα και θα που πρέπει να μας απασχολήσουν. Ε, το νομικό και το διοικητικό πλαίσιο για τον ανταγωνισμό σχολιάστηκε από τους συναδέλφους μου. Ε, δεν έχω και πολλά να προσθέσω. Ε, απλά θα ήθελα να ενισχύσω το μήνυμα που πέρασαν και εκείνοι. Δηλαδή, ε, θα πρέπει να υπάρξει ένα mainstreaming της υδατοκαλλιέργειας σε ευρύτερε πολιτικές. Πρέπει να αφιερώσουμε ένα ειδικό χώρο στις πολιτικές που εκπονούμε στην ε, υδατοκαλλιέργεια. Κυρίως στην έμεση νομοθεσία για να μην υπάρξουν ε, επιζήμιες επιπτώσεις στην υδατοκαλλιέργεια, ε, όχι εκ προθέσεως, αλλά που θα προκύψουν από νομοθετήματα που έμεσα επηρεάζουν το δυναμικό του κλάδου. Και πάλι είναι σημαντικό να δούμε το θέμα των χώρων της περιβαλλοντικής ε, προστασίας ε, και του ε, διεθνούς ανταγωνισμού και την αντιπαραβολή ανάμεσα στις ευρωπαϊκές πολιτικές και σε πολιτικές που ακολουθούνται σε άλλα μέρη του κόσμου. Η τεχνολογική πλατφόρμα που για την υδατοκαλλιέργεια είναι η ETIP και πρόσφατα έγιναν προσπάθειες για να αναγνωριστεί ως τέτοια. Υπάρχουν 7 θεματικές ενότητες για να καλυφθούν οι ανάγκες της βιομηχανίας. Προς το παρόν υπάρχει ένα ε, αρκετά ευρύ φάσμα επιχειρήσεων που εμπλέκονται στην ετοχνολογική πλατφόρμα. Υπάρχει γραμματεία από την Ομοσπονδία των Ιδατοκαλλιεργητών ε, ε, στην Ευρώπη και εμπλέκεται σε ε, διάφορα ε, προγράμματα. Το στοιχείο κλειδί είναι να μεριμνήσουμε ώστε γέρος να αναγνωριστεί ε, ως τεχνολογική πλατφόρμα αυτό το δίκτυο να, για να έχουμε και μεγαλύτερη επιρροή ο κλάδος και ακόμη πιο σημαντικό είναι να ε, είναι σε άμεση επαφή με τις ανάγκες ε, της ε, βιομηχανίας. Δηλαδή, οι πρωτοβουλίες ως προς την έρευνα να αντιστοιχούν στις ανάγκες και στις επιθυμίες του κλάδου. Θα προτείναμε να υπάρχει ένας μηχανισμός παρακολούθησης των επιδόσεων της πλατφόρμας για να δούμε ποια είναι τα πρότυπα αποδόσεων ε, του κλάδου, να τα συγκρίνουμε με διεθνή πρότυπα και να δούμε ακριβώς ε, σε τι συνεισφέρει αυτή η τεχνολογική πλατφόρμα στο να αυξηθούν οι επιδόσεις. Έχουμε και τρεις εγκάρσεις ε, συστάσεις. Η πολιτική για την υδατοκαλλιέργεια πρέπει να προάγει τα διά, τις διάφορες διαθέσιμες υποδομές του κλάδου, δηλαδή είτε μιλάμε για μικρή είτε για μεγάλη κλίμακα, παραδείγματος χάρη, και αν θέλουμε ε, μεγάλη παραγωγή στον τομέα τη ιδιωτοκαλλιεργία, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε το ότι χρειαζόμαστε μονάδες ε, μεγάλη κλίμακα ε, που θα παράγουν με αποτελεσματικό τρόπο και με σωστά πρότυπα τα προϊόντα τους. Δεύτερον, θα πρέπει να ε, δούμε ολόκληρη την αξία της αγοράς ε, στην, ε, σε σχέση με την υπόλοιπη αλυσίδα, να αναγνωρίσουμε ότι η ευρωπαϊκή δατοκαλλιέργεια είναι σημαντική, αλλά δεν είναι και το μοναδικό στοιχείο για την, τα οικονομικά οικονομικά κέρδη αφενός και για να καλυφθούν οι ανάγκες ε, του καταναλωτή αφετέρου. Επίσης, ρυθμίσεις στον εμπορικό τομέα και οι ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τις επιδοτήσεις, για τον έλεγχο ε, της εφαρμογής των διατάξεων, ε, για την προστασία του περιβάλλοντος, για την ευημερία των ζώων κτλ. Ούτως ώστε ο κλάδος να έχει μια ισχυρή βάση για να επενδύσει και να έχουν και μεγαλύτερη επιλογή οι καταναλωτές με μεγαλύτερη διαφάνεια. Σας ευχαριστούμε πολύ και καθώς πιέζει πολύ ο χρόνος Τώρα αυτό το σημείο θα το συνδέσω με το επόμενο σημείο διάταξη που είναι η έκθεση του κυρίου Μιλάνα για την ανακοίνωση της Επιτροπής και σας υπόσχομαι κύριε Μιλάνα ότι στην επόμενη συνεδρίασή μας το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη θα είναι το δικό σας. Έτσι λοιπόν εδώ θα πρέπει να το λάβει υπόψη αυτό και θα υπάρξει χρόνος και από τη γραμματεία για σας. Τώρα έχετε την παρουσίαση και αν υπάρξει χρόνος για συζήτηση θα το συνδυάσουμε με τους εισηγητές μας που είναι εδώ και με όλα τα θέματα αυτά. Έχετε τον λόγο κύριε Μιλάνα, παρακαλώ. Σε σας ευχαριστώ πολύ. Και θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω λέγοντας ότι το βλέπω θετικά ότι τώρα αυτό από κοινού θα το συζητήσουμε και θα το εξετάσουμε και μπορώ το ένα ή άλλο θέμα να, συμπληρώσει, να συμπληρώσουμε σε σχέση με τις παρεμβάσεις που έγιναν πιο πριν συμπληρωματικά. Υπόσχομαι θα είμαι πολύ σύντομος. Λοιπόν, οι μελέτες ε, της ε, σημερινής πρωίας επιβεβαίωσαν αυτό που την τελευταία φορά είχα επισημάνει, είχα ε, σκιαγραφίσει. Έχουμε μια κατάσταση γενικότερη μπροστά μας, όπου όλα όσα η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε ως πρωτοβουλίες μέχρι σήμερα, ουσιαστικά συνδέονται με ένα, επιβαρύνονται με ένα πρόβλημα, πρόβλημα θεμελιώδες θα έλεγα, θέμα αρχής, θέματος αρχής. Καταδείχθηκε δηλαδή ότι εμείς δεν είμαστε υπαρκώς παραγωγικοί ότι σε σχέση με την εξέλιξη όσον αφορά την ενιαία εσωτερική αγορά δεν μπορέσαμε να ικανοποιήσουμε τη ζήτηση και ότι η δική μας η ε, παραγωγή δεν είναι επαρκώς ανταγωνιστική έναντι των εξωτερικών ανταγωνιστών τους. Δεύτερο πρόβλημα, οι μαζικές εισαγωγές. Ενώ μεταξύ αυτό έχει καταστεί ένα οικονομικό πρόβλημα πρώτου μεγέθους και αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας κίνδυνος σίγουρα για τους, και για τους καταναλωτές τους καταναλωτές μας όταν καταναλώνουν και αγοράζουν προϊόντα τα οποία προέρχονται από τρίτες χώρες. Πρόκειται εδώ λοιπόν ακριβώς για την ίδια την προστασία των καταναλωτών, την ίδια την υγεία και την ασφάλεια και διασφάλιση της υγείας τους. Πρέπει να προσπαθήσουμε λοιπόν να κάνουμε ένα ποιοτικό άλμα, ένα μεγάλο ποιοτικό άλμα προς τα εμπρός. Και θα πρέπει επιτέλους από την φάση των συστάσεων και όλων αυτών να ε, διαφύγουμε πλέον και να προχωρήσουμε προς τα εμπρός θα πρέπει να πάμε, ας το πω έτσι χειροπιαστά, να κάνουμε αυτό το ποιοτικό άλμα που θα πετύχουμε, πρέπει να το πετύχουμε από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιο ενισχυμένα πρέπει να δράσουμε προ αυτήν την κατεύθυνση. Πώ μπορεί να γίνει αυτό, Υπάρχει ένα κανονισμό, υπάρχει σίγουρα και εντωμεταξύ υπάρχουν σχέδια οι προτάσεις θα έλεγα σπέρματι για μια κοινή τέτοια πολιτική που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε. Πρέπει τώρα όμως να παρέμβουμε, να δράσουμε, να δραστηριοποιηθούμε. Τώρα πρέπει να κάνουμε κάτι χειροπιαστά. Η καιρή ουμενετή. Δηλαδή πρέπει με θετικό τρόπο να δράσουμε, να υιοθετήσουμε μια, ας το πω έτσι, θετική ε, αντιμετώπιση των πραγμάτων δραστηριοποιούμενοι. Και με τους κοιόδης συζητητές ε, ήδη μπόρεσα να συζητήσω αυτό το θέμα, να το εξετάσουμε. Πρέπει πιο ενισχυμένα να ενταχθούν και να εμπλακούν οι παραγωγοί, οι ενώσεις σύλλογοι παραγωγών και όλα αυτά να ενταχθούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Και εδώ δεν χρειάζεται ε, να αναλύσω κάποιες λεπτομέρειες και ούτε μπορώ να ξετυλίξω όλο το σκηνικό μπροστά σας. Δεν επαρκεί ο χρόνος. Όμως η κατάσταση είναι προβληματική και πιέζει ο τομέας νοσεί. Νοσεί από ένα πολύ χαμηλό ποσοστό ανάπτυξης, αν καν μπορούμε να κάνουμε λόγο για ποσοστό ανάπτυξης τα τελευταία αυτά χρόνια της αποτελμάτωσης που λιμνάζουν τα πράγματα στον τομέα της, των υδατοκαλλιεργειών υπάρχουν περιορισμοί, όροι προϋποθέσεις ε, όσο αφορά το περιβάλλον, την υγεία των, ε, ε, των έμβιων αυτών όντων. Είναι, χρειάζονται τεράστιες επενδύσεις που ουσιαστικά πρέπει να καλυφθούν για να ανταποκριθούμε στις ευθύνες και υποχρεώσεις μας. Πρέπει να καταφέρουμε να έχουμε μια καλύτερη βιομηχανική ανάπτυξη, να καταφέρουμε να λάβουμε τα αναγκαία εκείνα μέτρα που θα θέσουν τη νέα τροχιά, τη νέα πορεία προς το μέλλον. Και δεν είναι μόνο όλες οι υδατοκαλλιέργειες οι ίδιες η μία με την άλλη, όσον αφορά και την προστασία του περιβάλλοντος και των εμβιονόντων και την οικονομική του σημασία. Υπάρχουν διαφορές και πρέπει έχουμε τα ε, τους έχουμε ηχθειολογικά ε, γλυκού υδάτος, ε, εσωτερικών υδάτων, ψάρια, έχουμε ανοιχτή θάλασσα ψάρια. Υπάρχουν ιδιομορφίες και πρέπει να λάβουμε υπόψη τις διαφοροποιήσεις αυτές από υδατοκαλλιέργεια σε υδατοκαλλιέργεια. Πρέπει να λάβουμε υπόψη διαφοροποιημένα αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Οι Γάλλοι, οι Ιταλοί οι για παράδειγμα ίσως εσωτερικά μπορεί κανείς να πει σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανταγωνιστική, αλλά όχι διεθνώς. Δεν είναι διεθνώς ανταγωνιστική. Υπάρχουν προσκόμματα και εμπόδια για μια αηφορία και ε, θα έλεγα θετική ανάπτυξη. Και αυτές οι διαφορές που υπάρχουν όρων και προϋποθέσεων, ακόμα και σε διοικητικό επίπεδο, πολλά κράτη-μέλη ε, έχουν διαφορετικές διατάξεις. Εμείς οι ίδιοι επιβαρύνουμε τα πράγματα και δυσχεραίνουμε τα πράγματα για μας τους ίδιους με όλες αυτές τις ε, διατάξεις και επιπλέον δεν υπάρχει ενιαίος προγραμματισμός. Δεν υπάρχει προγραμματισμός θα έλεγα ή σχεδιασμός σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Υπάρχουν κάποιες προσεγγίσεις και προσπάθειες επιτόπου ένα εγχείρημα το ένα ή άλλο που ξεκινά ένα διάλογο με μια τοπική αρχή σε περιφερειακό επίπεδο. Όμως αλλού γίνεται ο σχεδιασμός όσον αφορά χωροταξικά θέματα και πολεοδομικά. Υπάρχει προγραμματισμός, αλλά εδώ σε αυτό τον τομέα λείπει αυτός ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός πανευρωπαϊκά και έτσι δεν έχουμε ένα ενιαίο πλαίσιο. Στο τέλος, τέλος τι απομένει. Απομένει το ζήτημα και τώρα πρέπει, ας το πω έτσι, να κάνω κάποια άλματα, να επιταχύνω. Χρειαζόμαστε αυτό το ποιοτικό άλμα που πρέπει να επιτευχθεί όπως προανέφερα και αυτό χωρίς νομοθεσία δεν γίνεται. Πρέπει να στραφούμε λοιπόν σε ένα μεγάλο βήμα που θα κάνουμε. Θα τολμήσουμε, θα αποτολμήσουμε να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα. Έχουμε προβλήματα και με την Τουρκία και με την Κίνα, με διάφορες χώρες. Εκεί τι βλέπουμε. Όλο το κόστος ε, εκμετάλλευσης από αυτές τις χώρες. Σε αυτές τις χώρες είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Το περιβάλλον δεν προστατεύεται. Οι, προ... οι διατάξεις για την προστασία της υγείας δεν είναι ίδιες όπως εμάς. Δεν υπάρχουν περιοριστικοί όροι και τέτοιες επιβαρύνσεις. Και υπάρχουν εδώ παράγοντες που μπορούν να είναι επικίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία και δεν, δεν αποκλείονται λόγω αυτής της ανεξέλεγκτης δραστηριότητας. Τώρα, ποιες δράσεις θα συμφωνηθούν από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει όποιες και να είναι αυτές οι δράσεις να λαμβάνουν πάντα υπόψη την αηφορία. Αυτή να είναι ο στόχος, η στοχοθέτηση, η αηφορία και στον τομέα του περιβάλλοντος και οικονομικά. Αηφορία λοιπόν διτή, δύο πράγματα που ιδιαίτερα όσον αφορά την αλία στο μέλλον πρέπει να λάβουμε ιδιαίτερα υπόψη. Και τούτων λεχθέντων με, πολλούς, με πολλές ενώσεις και συλλόγους ε, ε, που ασχολούνται με το περιβάλλον ήρθα σε επαφή. Όλοι λένε ότι είναι υγιές να καταναλώνουμε περισσότερα ψάρια. Αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το επίπεδο. Και σε μία από τις εκθέσεις καταδείχθηκε αυτό ανάγλυφα και αναφέρθηκε εξάλλου στην τοποθέτηση. Πρέπει να δημιουργηθούν οι εναλλακτικέ δυνατότητες επιλογής για τους καταναλωτές. Δυνατότητες να επιλέγουν. Χρειάζεται κανείς σε πρωτεΐνες μια πιο πλούσια διατροφή πλουσιότερα σε πρωτεΐνες τρόφιμα. Αυτές οι πηγές όμως πρωτεϊνών δεν μπορούν να αποκλείουν, για παράδειγμα, μια αυξημένη κατανάλωση ε, αλλιευμάτων που θα μπορούσε να επιλέγεται. Πρέπει να σκεφτούμε και να προβληματιστούμε. Οι δατοκαλλιέργειε είναι αυτό που θέλουμε να αναπτυχθούν. Ίσως όμως και άλλοι τομεί θα έπρεπε να προαχθούν. Χέρι με χέρι παράλληλα με τι δράσει μα για την υδατοκαλλιέργεια. Και όλα αυτά προ όφελο μια ευρύτερη παραγωγή, θα έλεγα θετική εξέλιξη ε, στην αύξηση των πρωτεϊνούχων ε, τροφίμων. Και αυτό θα μπορούσε να είναι κάτι θετικό και για την απασχόληση στη συνέχεια. Με άλλα λόγια, τα αναφέρω όλα αυτά ως παράδειγμα. Υπάρχουν επιχειρήσεις που ασχολούνται με τις υδατοκαλλιέργειες που οπωσδήποτε με φιλοπεριβαλλοντικές μεθόδους παράγουν σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν στο περιφερειακό, στο τοπικό επίπεδο. Φυσικά από την άλλη πλευρά οι πρωτεΐνες δεν πρέπει υποχρεωτικά να είναι ζωικής προέλευσης. Δεν είναι υποχρεωτικά τα πρωτεϊνούχα όλα τα τρόφιμα υποχρεωτικά ζωικής προέλευσης ή ιδιαίτερα και ε, όσον αφορά τα ψάρια. Υπάρχουν ε, και οι νέες τεχνολογίες κατά τα άλλα που είναι στη διάθεσή μας και που θα έπρεπε να εξεταστούν όσον αφορά τις ε, επιπτώσεις και τις ε, ε, τα αποτελέσματά τους. Πρέπει στα ερευνητικά προγράμματα και σχέδια να μεριμνούμε ώστε τα αποτελέσματα πραγματικά να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολυθούν περαιτέρω ποιοτικά άλματα τα οποία θα μπορέσουμε να κάνουμε. Ολοκληρώνω μέσω πρόεδρε, λέει ο μιλητής. Με άλλα λόγια, δεν πρέπει, δεν επιτρέπεται ακόμα περισσότερη ρήπανση να προκαλείται από αυτήν την αυξημένη ηχθειολογική ηχθειοπαραγωγή ή καλλιέργεια ηχθείων. Όπως είπα, σίγουρα υπάρχουν, όπως γνωρίζουμε, περιτώματα ή ε, απόβλητα τα οποία προκαλούν υδατοκαλλιέργειες, αλλά αυτές, αυτά δεν πρέπει να επιβαρύνουν υπερβολικά το περιβάλλον. Υπάρχουν κανόνες, πρέπει οι κανόνες να εφαρμόζονται με τη σωστή επιτήρηση και εποπτεία να ελέγχονται οι δραστηριότητες αυτές. Με άλλα λόγια πάλι, τι πρέπει να γίνει. Πρέπει μια σφαιρική προσέγγιση να αναπτυχθεί και να υιοθετηθεί, ώστε όλα αυτά να ταιριάζουν το ένα με το άλλο και να αλληλοσυνδέονται και να είναι αλληλοσυμβατά αμφίπλευρα. Δεν μπορεί κανείς να αυτό σχεδιάζει. Πρέπει σε βάθος να μελετηθούν και να εξεταστούν όλα αυτά και έτσι να μπορέσουμε να δράσουμε. Πρέπει να υπάρχει μια αξιόπιστη βιώσιμη βάση όλων αυτών ως δραστηριοτήτων και προς όφελος των πολιτών. Διότι είναι ένα επάγγελμα το επάγγελμα των αλλιέων και πρέπει να είναι ένα επάγγελμα με σίγουρο διασφαλισμένο μέλλον. Και όταν έχουμε και την επένδυση που επιτυγχάνεται σε έναν ε, επαγγελματικό τομέα και μια επαγγελματική δραστηριότητα, πρέπει να υπάρχει μελλοντική προοπτική για αυτό το επάγγελμα. Αυτές είναι οι προτάσει που σύντομα ήθελα να σα παρουσιάσω. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια εναρμονισμένη θα έλεγα δομή που μέσα σε ένα ενιαίο πλαίσιο θα διασφαλίσει την ταχύ ανάπτυξη του τομέα της υδατοκαλλιέργειας. Με τα αναγκαία φυσικά νομικά πλαίσια και νομοθετικές διατάξεις και ρυθμίσεις, ώστε αυτό το προϊόν το οποίο έχει μεγάλο δυναμικό να μπορέσει να ευδοκιμήσει και να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί, να εκμεταλλευτούμε αυτό το προϊόν θετικά όσο αφορά το δυναμικό του. Να δημιουργήσουμε τις συνθήκες πλαίσιο, με άλλα λόγια, ώστε αυτή η ανάπτυξη να μπορέσει να επιτευχθεί. Με άλλα λόγια, όλη η αλυσίδα των προϊόντων πρέπει να είναι με τέτοιο τρόπο διαφανής, ώστε τα αποτελέσματα να μπορούν να ειχνηλατηθούν από την αρχή της ε, ε, δημιουργίας του προϊόντος μέχρι το τέλος. Να ξέρουμε, να μπορούμε να ειχνηλατήσουμε, να ανοιχνεύσουμε από πού προέρχεται και πώς παράγεται ένα προϊόν. Όλα αυτά με αριθμητικά μεγέθη πρέπει να δομούνται. Παράδειγμα, βιομάζα καταλήγει ένα προϊόν στην αγορά και δεν γνωρίζουμε τι γίνεται με όλα αυτά τα στοιχεία, π.χ. την βιομάζα. Από πού προέρχεται αυτό το προϊόν, πού παρήχθη, η έδρα παραγωγή μα ενδιαφέρει επίση και οι τρόποι παραγωγή. Θέλουμε φυσικά επίση να γνωρίζουμε πόσα ψάρια ζουν, συμβιώνουν μέσα σε ένα κυβικό μέτρο νερού, για παράδειγμα, σε αυτές τις ηθιοκαλλιέργειες. Όταν γνωρίζει κάποιος όλα αυτά τα στοιχεία, τότε μπορεί να γνωρίζει και για την ποιότητα του προϊόντος το τι συμβαίνει. Χρειάζεται έλεγχος όλης συνολικά της αλυσίδας των προϊόντων και χρειαζόμαστε και ένα ταμείο όπου αυτά τα μέτρα της πολιτικής στους διάφορους τομείς και παιδεία θα μπορούν να στοχεύουν στην, σωστού ε, ε, στους στόχους ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί αμφίδρομα. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση όπου, πώς να το πω, έχουμε μια ε, μη επαρκή κάλυψη των αναγκών όσον αφορά τη ζήτηση με προϊόντα τα οποία θα μπορούσαν να είναι καλύτερα. Πρέπει τώρα να γίνει το βήμα εκείνο για την αυτάρκεια, την ε, κάλυψη των αναγκών και τη ζήτησή μας με τα δικά μας προϊόντα. Υπάρχει δυναμικό. Δεν έχουμε αρκετά ε, προϊόντα από πλευράς ε, των αλλιευμάτων. Υπάρχει τεράστιο κενό όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών μας. Έχουμε πολύ μικρή παραγωγικότητα όσον αφορά τις ε, συνολικές ανάγκες. Πρέπει να γίνουν επενδύσεις, πρέπει να μπορέσουμε αυτό το κενό να το καλύψουμε. Ένα τεράστιο βήμα πρέπει να γίνει. Έκανα λόγο για αυτό το ταμείο προηγούμενα. Πρέπει η προσπελασιμότητα να ρυθμιστεί, η προσβασιμότητα σε αυτό το ταμείο, να διευκολυνθούν τα πράγματα. Πρέπει να γίνουν περισσότερες έρευνες όσον αφορά την θάλασσα, το υδάτινο περιβάλλον, την πολιτική για τους ωκεανούς και τις θάλασσες, το υδάτινο περιβάλλον. Στόχος αυτής της έρευνας πρέπει να είναι να καταλήξουμε σε αξιόπιστους συγκεκριμένους δείκτες για την πολιτική μας, μελλοντική αλληλευτική πολιτική. Ίσως τα ρίξα όλα ισοπεδωτικά σε ένα ε, και ίδιο πλαίσιο, αλλά και τα κάλυψα όλα αυτά βιαστικά. Ε, και ίσως λείπει ο μύτος της Αριάννης, αλλά είχα πολλές ιδέες και μια και πίεζε ο χρόνος προσπάθησα να τα παρουσιάσω όλα αυτά φίρδιν μίγδιν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, είσαστε σαφεί, θα έλεγα. Στι 12.30 ακριβώ πρέπει να ολοκληρώσουμε. Θα δώσω τον λόγο στον κύριο Τσουκαλά που τον ζήτησε να παρέμβει και στη συνέχεια σε κάποιους άλλου, η Επιτροπή και μετά ο κύριο Μιλάνα. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο για Τσουκαλά. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, εγώ από την παρουσίαση των τριών μελετών θα φύγω σήμερα σοφότερος. Νομίζω ότι θα συμφωνήσω με τον κύριο Μιλάνα ότι οι μελέτες δεν μπορούν να αποτελέσουν πολιτική, όμως μας δίνουν ε, και τουλάχιστον με την εμβρήθεια που ασχολήθηκαν με το περίπου συνολικό πλέγμα των προβλημάτων της υδατοκαλλιέργειας, μου φάνηκαν ε, πάρα πολύ χρήσιμες. Δεν θα επεκταθώ πολύ, θα ήθελα να εστιαστώ σε δύο σημεία. Το πρώτο σημείο είναι οι επενδύσεις σε έρευνα και τεχνολογία. Ίσως μάλιστα αυτό θα έπρεπε η τρίτη μελέτη μας το τόνισαν με μεγάλη εμφαντικότητα. Θα έπρεπε ίσως οι καινοτόμες λύσεις που μπορεί η τεχνολογία να βρει να δίνουν ε, ε, καλύτερα αποτελέσματα από τις κλασικές που σήμερα ξέρουμε. Για παράδειγμα, ε, γνωρίζω ένα πρόσφατο πρόγραμμα που έγινε στο MIT όπου αναπτύχθηκαν κινητές ρομποτικές μονάδες ηχθειοκαλλιέργειας, δηλαδή μεγάλα κλουβιά αυτοκινούμενα με προπέλες και με αυτή τη μέθοδο ισχυρίζονται ότι επιτεύχθηκε μεγάλη παραγωγικότητα σε συνδυασμό με ελάχιστη επίπτωση στο περιβάλλον. Επομένως, ε, ένα στο οποίο εστιάζομαι είναι οι επενδύσεις με όλα τα εργαλεία που μας είπε η τρίτη μελέτη σχετικά με την τεχνολογική ανάπτυξη στον τομέα. Τώρα, για να δώσουμε μια απαραίτητη όθηση σε μια βιώσιμη τατοκαλλιέργεια, η οποία είναι προφανές ότι είναι σημαντική και κοινωνικά και οικονομικά και περιφαντολογικά και για να αντιμετωπίσουμε τη ραγδαία ανάπτυξη της παραγωγής που ακούσαμε στις ε, τρίτες χώρες. Αν θυμάμαι καλά τους αριθμούς, μισό της εκατό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 7,2% σε τρίτες χώρες, για να αντιμετωπίσουμε την, το ποιοτικό ζήτημα που ο κύριος Μιλάνα μας είπε προη, ε, ε, προηγουμένως, καλό θα ήταν πράγματι να υπάρξει μια ενιαία νομική βάση και να ληφθούν μέτρα δεσμευτικά για όλους. Δεν γνωρίζω ακριβώς πώς θα γίνει αυτό, με οδηγία, με κανονισμό. Νομίζω όμως ότι πρέπει να γίνει. Τέλος, ε, έτσι απλώς για να το αναφέρω, μου έκανε εντύπωση η προαγωγή των κορμοράνων σε τρομοκράτες, ενώ στη βάση δεν έχουμε παρά μια διένεξη μεταξύ δύο ειδών περί της τροφής. Είναι human animals και non-human animals και έχει μεγάλο ενδιαφέρον πόσο τα χρειάζεται η ανθρωπότητα στην ηθική της όταν πρέπει να εφαρμόσει τις μεγαλόστομες ε, αρχές της ε, διατήρησης της βιοποικιλότητας ή της προστασίας του περιβάλλοντος. Απλώς λίγο να τονίσω όταν το κάνουμε αυτό ότι και ο κινέζικος πληθυσμός αυξάνεται πολύ. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε κύριε Τσουκαλά έχουν εγγραφεί η κυρία Λεβίν και η κυρία Πατρόνες. καθώ καθώς ε, έχουν παρέμβει, παρακαλώ, για να καταφέρουμε να απαντήσουν, να έχουμε απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μόνο ερώτηση να διατυπώσουν, όχι σχόλια. Κυρία Λεβίν, παρακαλώ. Ε, ε ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μίλαν ε, για τη δουλειά που κάνετε. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής ε, για τη σχέση με τις ε, ε, τροφές για τα ψάρια, τα ηχθιάλευρα και τις σχέσεις ανάμεσα στα εκτρεφόμενα και τα άγρια ψάρια. Ε, για, ε, θα ήθελα να αναφέρω στο, το ότι στη Νορβηγία έχουν γίνει ε, σοβαρές προσπάθειες για να καταναλώνται λιγότερα άγρια ψάρια για να εκτραφούν ε, τα ψάρια των υδατοκαλλιεργειών. Ε, και είναι πάρα πολύ δύσκολο να χρησιμοποιήσουμε φυτικά λίπη και όχι θαλάσσια λίπη, λίπη από τα ψάρια για να φρέψουμε ε, τα ε, ψάρια της υδατοκαλλιέργειας. έχετε περισσότερα στοιχεία για αυτό το θέμα, κυρία Παντρονέβε. Μία ερώτηση, λοιπόν, και πολύ σύντομα. Ποιος είναι ο χώρος, ο ίδιος ο χώρος για την υδατοκαλλιέργεια που θέλουμε να δούμε να αναπτύσσεται. Είναι ένας χώρος ξεχωριστός, ιδιαίτερος λόγω της ανάπτυξης της επιστημονικής και τεχνολογικής που υπάρχει. Είναι ένας ενσωματωμένος, ολοκληρωμένος χώρος μέσα στον ευρύτερο τομέα των, της αλίας και έχοντας δράση και ρόλο συμπληρωματικό όσον αφορά την, το εισόδημα των αλιαίων και την αξιολόγηση και αναβάθμιση και επαγγελματική από πλευρά τους. Κατά τα άλλα, δεν θα ήταν δυνατόν να έχουμε υδατοκαλλιέργεια αν δεν είχαν και δεν ανέπτυσαν δραστηριότητε όσοι δραστηριοποιούνται στο τομέα τη αλίας. Θα ήθελα απλώ να μου αποσαφηνίσετε αυτό το ερώτημα. Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Ολοκληρώνουμε με μια ερώτηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα δώσουμε τον λόγο στην Επιτροπή και μετά τον κύριο... Ε, θα απευθύνω μια ερώτηση προ την Επιτροπή και μετά θα δώσει τον λόγο και ο, ο κύριος Μιλάνα. Είχαμε και τους ε, εκπροσώπου του τομέα που μα είπαν ότι υπάρχει ε, dumping όσον αφορά τα εισαγόμενα την Τουρκία προϊόντα συγκεκριμένα συγκεκριμένα ηθιοπροϊόντα και όσον αφορά την παραγωγή και την ε, εξαγωγή. Θα ήθελα να ξέρω για αυτό το θέμα τι γίνεται. Τώρα λοιπόν θα λάβετε τον λόγο εσείς για πέντε λεπτά, μετά ο κύριος Μιλάνα και θα ολοκληρώσουμε τη συνεδρίαση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι στο επίκεντρο του προβληματισμού ε, τίθεται η ιδέα ε, της συγκέντρωσης των διαφόρων μέτρων ε, της ε, υδατοκαλλιέργειας υπό ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο. Όπως γνωρίζετε η κατάσταση αυτή τη στιγμή δεν έχει καθόλου έτσι. Η κοινοτική ε, αρμοδιότητα, κάτι το οποίο έχει τονιστεί πολλές φορές, ε, στον τομέα αυτό είναι περιορισμένη η κοινοτική αρμοδιότητα στο πλαίσιο της κοινή αλλιευτικής πολιτικής, παρά το γεγονός ότι η υδατοκαλλιέργεια αναφέρεται στον ε, βασικό κανονισμό της κοινή αλλιευτικής πολιτικής, περιορίζεται επίσης η κοινοτική αρμοδιότητα και σε ένα πλαίσιο που θα επέτρεπε να ε, συγκεντρωθούν όλα αυτά τα ζητήματα που δημιουργούν πρόβλημα στο τομέα τη υδατοκαλλιέργεια. αλλά η υδατοκαλλιέργεια είναι αντικείμενο πολλών ε, νομοθετικών ε, διατάξεων όσον αφορά την ευημερία των ζώων, όσον αφορά το περιβάλλον, όσον αφορά τη θαλάσσια πολιτική, στο πλαίσιο τη θαλάσσιας χωροταξίας που επίση είναι αντικείμενο τη γενική μα διεύθυνση. Η υδατοκαλλιέργεια λοιπόν είναι αντικείμενο πολλών πολιτικών ε, κοινοτικών, αλλά δεν είναι αντικείμενο κοινή πολιτική. Και το ζήτημα που έθεσε ο εισηγητή σα είναι ακριβώ αυτό. Αν είναι σημαντικό, αν έχει νόημα να υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο να συγκεντρώνει όλα αυτά τα ε, νομοθετήματα. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε όμω σήμερα, γιατί είδα το καλλιέργεια είναι αντικείμενο αξιολόγησης και διαβούλευσης στο πλαίσιο τη κοινή αλληλευτική πολιτική. Είδα το καλλιέργεια λοιπόν είναι τμήμα όλου αυτού του προβληματισμού και ε, οι απαντήσεις ε, θα δοθούν ενδεχομένως ε, εν μέρη κατά το τέλος της διαβούλευσης και εν μέρη όταν θα μπορέσει η Κομισιό να τοποθετηθεί ποιόσον, θα έχει ακούσει σε σχέση με το θέμα αυτό. Αυτά ήθελα να σας πω και αυτά είναι τα σχόλιά μου σε σχέση με όσα κατάλαβα και από την παρέμβαση του κυρίου Μιλάνα. Υπήρξαν και κάποιες ερωτήσεις ε, που απευθύνθηκαν συγκεκριμένα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα προσπαθήσω με τον συνάδελφο ε, να, με τη βοήθεια και του συναδέλφου να απαντήσω. Το ζήτημα που τίθεται συνεχώς είναι η σχέση μεταξύ της ε, ε, διατροφής και το, της υδατοκαλλιέγριας. Δηλαδή πρέπει ένα άγριο ψάρι να χρησιμοποιείται ως τροφή σε ένα εκτρεφόμενο ψάρι. Ε, ποια είναι η απόδοση πρωτεϊνική όλης αυτής της προσπάθειας και όλης αυτής της μεταποίησης που πρέπει να γίνει. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι ε, κατ' ουσίαν να ξέρουμε μήπως είναι προτιμητέο ε, να έχουμε κάποια συγκεκριμένα ψάρια τα οποία δεν καταναλώνουν ιδιαίτερα οι άνθρωποι ε, ή για παράδειγμα μερλούκιο ή βακαλάο ε, και να χρησιμοποιούμε τα πλεονάσματα αυτά ε, για να τρέφουμε τα εκτρεφόμενα ψάρια. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα Υπάρχει ένα πρόβλημα διάρθρωσης όμως ε, σε σχέση με, τη με την διατροφική αλυσίδα. Δεν είναι πολύ εύκολο δηλαδή να απαντηθεί αυτό το ερώτημα. Αν οι μελέτες είναι σωστές, η απόδοση της υδατοκαλλιεργίας δεν είναι καθόλου αμεληταία. Ε, είναι τόσο καλή μάλιστα που να μπορούμε να ε, συμπεριλάβουμε και φυτικής προέλευσης πρωτεΐνες στο, στις ηχθειοτροφές. Επίσης, όσον αφορά το Ταμείο που θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε για την υδατοκαλλιέργεια. Έχουμε ήδη ένα ταμείο αλίας σήμερα, το οποίο δίνει τη δυνατότητα προ... πρόσβασης ε, στο πλαίσιο του άξονα 2. Ε, υπάρχει ένας προγραμματισμός ε, πλήρως διαφοροποιημένος, ε, ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί από την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργεια ε, σε κράτη-μέλη τα οποία έχουν ε, ζητήσει να υποφεληθούν από τα διαρθρωτικά ταμεία. Ε, κάτι το οποίο δίνει τη δυνατότητα βέβαια να υπάρξει μια επιπλέον και σημαντική χρηματοδότηση για τις δραστηριότητες αυτές. Τώρα, το γεγονός ότι Υπάρχει ενίσχυση και των εξαγωγέων μας ε, σε αγορές ε, εκτός ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένωσης τι, θέτει ένα ζήτημα του ποιος είναι, πώς διέπονται όλες αυτές οι εξαγωγές αλλά ο συνάδελφος νομίζω ότι είναι πιο αρμόδιος να μας απαντήσει για το θέμα του dumping ε, της ε, Τουρκίας που έθεσε η κυρία Φράγκα. Ναι κυρία Πρόεδρε, απλώς ήθελα να απαντήσω στο ερώτημά σας για την Τουρκία μετά από την ακρόαση που, έγινε ε, σήμερα στην Επιτροπή, ε, στην Επιτροπή σας, ε, υπήρξαν συγκεκριμένες αγωγές, τις οποίες αυτή τη στιγμή εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμως είναι μια μακρόχρονη διαδικασία αυτή και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού ζήτησε περισσότερες πληροφορίες από τον κλάδο, γιατί κάποια στοιχεία έπρεπε να αποσαφινιστούν. Αν θέλετε όμως μπορώ να ενημερωθώ, να μάθω περισσότερες λεπτομέρειες και να σας πω. Κύριε Μιλάνα, τώρα έχετε δύο λεπτά στη διάθεσή σα για να ολοκληρώσετε. Λοιπόν, φτάνει και λιγότερο για να ολοκληρώσω. Ευχαριστώ. Ξεκινώ. Βλέπετε, είμαστε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εντάξει, δεν είμαστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και, πώς να το πω, Πρέπει να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε επί μια ανακοίνωση και γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ. Αυτό είναι το νόημα του εγχειρήματο. Θέλουμε να επιτύχουμε μια αηφόρο πολιτική όσον αφορά την υδατοκαλλιέργεια για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι και ο τίτλο του πονήματο που μα απέστειλε και κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με άλλα λόγια, αν επιθυμείτε μια γνωμοδότηση από εμά, θα πρέπει να λάβετε υπόψη και τι επιθυμίε μα και όσα διατυπώνουμε, γιατί διαφορετικά περιτεύει να συζητούμε για οποιαδήποτε τέτοια θέματα όσον αφορά πολιτική. Και να προσθέσω και τούτο. Πιστεύω, θεωρώ προσωπικά ότι αυτά που πιέζουν ούτως ή άλλως και χρονικά είναι και ότι δεν είχαμε μια τέτοια πολιτική μέχρι σήμερα. Ομολογουμένω η αλλω και χρονικα ειναι και οτι δεν ειχαμε μια τετοια πολιτικη μεχρι σημερα ομολογουμενως η υπάρχουν πτυχές όσον αφορά το περιβάλλον, την υγεία, όσον αφορά ε, τις, ε, τα θέματα επιπτώσεων στην υγεία. Όλα αυτά τα γνωρίζουμε. Πρέπει όμως να αποφασίσουμε κάτι. Θα συνεχίσουμε τώρα να εξαρτώμεθα από εισαγόμενα ψάρια από τον υπόλοιπο κόσμο, από το Φαντάζιους για παράδειγμα, από το Βιετνάμ, αν είναι κιόλα και υγιέ αυτό για την κατανάλωση. Είναι καλό αυτό μακροπρόθεσμα για την Ευρώπη. Μήπως θα έπρεπε να σκεφτούμε και να προβληματιστούμε αν θα ήταν καλύτερο εμείς ως Ευρωπαίοι ίδιοι να προαγάγουμε μια νέα στρατηγική, να αποφασίσουμε να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί, να είμαστε στο τέλο τέλο ανταγωνιστικότεροι έναντι των χωρών που μα ανταγωνίζονται για παράδειγμα όσον αφορά και θέματα χειροτροφίας ε, και εκμεταλλεύσεις ε, χειροτροφικές και αυτές δημιουργούν επιβάρυνση και επιβαρύνουν το περιβάλλον. Και υπάρχει εδώ μια κοινή αγροτική πολιτική και για τα τα ζώα στην Ευρώπη υπάρχει και μια κοινή προσέγγιση πάλι και για αυτά ευρωπαϊκά, πανευρωπαϊκά. Να κάνουμε κάτι για τα ψάρια, το ίδιο λοιπόν. Γιατί να μην υπάρχει κάτι παρόμοιο όσον αφορά τις υδατοκαλλιέργειες ε, και ε, σε σχέση με την ε, προλαλή σας, εκείνο που θα ήθελα να πω είναι το εξής. Προσέξτε, χρειαζόμαστε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, μονάδες υπό την κλασική έννοια. Χρειαζόμαστε όμως και βιολογικές ε, προσπάθειες ε, και εξοπλισμό και μονάδες. Πρέπει η ποιότητα να έχει πρωτεύοντα ρόλο και να, να είμαστε πρωτοπόροι και να υπάρχουν οι μονάδες οι παραγωγικές ε, για να τα καταφέρουμε. Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις στην κλασική προσέγγιση, έναντι των κλασικών προσεγγίσεων της αλληλείας για παράδειγμα όπως αυτήν ε, ακολουθούσαμε και να υπάρξει μια μετάθεση όσον αφορά ε, τις, ε, τους απασχολούμενους. Να διασφαλιστούν οι θέσεις τους αλλά να δούμε σε ποιο τομέα δραστηριοτήτων θα διασφαλιστούν οι θέσεις αυτές και με ποιον τρόπο. Και στην Πράσινη Βίβλο για το μέλλον της ε, πολιτικής της αλίας, για την αλία, πρέπει να πούμε κάτι συγκεκριμένο σχετικά για τις υδατοκαλλιέργειες. Δεν μπορούν να αποσυνδεθούν οι υδατοκαλλιέργειες από την αλλιευτική πολιτική, μια και αποτελούν μέρος της αλλιευτικής δραστηριότητας. Ευχαριστώ, ολοκληρώνουμε τη συνεδρίασή μας, ευχαριστώ τους διερμηνείς. Αυτή η έκθεση θα συνεχίσει να συζητείτε τους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ όλους σας. Λίγη συνεδρίασή μας μέχρι το απόγευμα. Γεια σας.